Συνεχίζουμε λοιπόν ε, τη συνεδρίασή μας. Καλησπέρα. Χαίρομαι που παρευρίσκεστε σήμερα όλοι εδώ. Θα συζητήσουμε για τις επόμενες δύο ώρες ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον ε, θέμα. Το Σεπτέμβριο είχαμε προβεί σε μια fact-finding mission στην Ελλάδα και επισκεφθήκαμε εκεί 7 έργα και συζητήσαμε βέβαια με τις αρμόδιες αρχές από την πλευρά της Ελλάδας. Δεν είχαμε ακόμα επαφές με την ελληνική κυβέρνηση γιατί τότε βέβαια προκυρήσονταν ε, και πάλι εκλογέ στην Ελλάδα οπότε δεν θέλαμε να θέσουμε ενδεχομένω κάποιου σε δύσκολη θέση. Όμω ε, είχαμε τότε δεσμευτεί ότι θα υπάρξει ένα follow-up θα δώσουμε δηλαδή μια συνέχεια στη διαδικασία με βάση τις εμπειρίες που αποκομίσαμε εκεί από την Ελλάδα και ακριβώς σε σχέση με τα προβλήματα που είδαμε εκεί σε σχέση με την υλοποίηση των απαλωτριώσεων. Ακριβώς και γι' αυτό αποφασίσαμε να θέσουμε στο σήμα της ημερήσιας διάταξή μας το ζήτημα των απαλωτριώσεων. Υπάρχει ένας αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα, το οποίο έχουν κατασκευαστεί ήδη 25 ε, χιλιόμετρα, αλλά δεν μπορεί κανείς να εισέλθει σε αυτό το αυτοκινητόδρομο, ούτε να εξέλθει ακριβώ γιατί τα σχετικά κομμάτια ε, ε, δηλαδή τη εισόδου και εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο, δεν είχαν απολωτριωθεί ακόμα. Και προφανώ αυτό θα πρέπει να συζητηθεί αφού κάθε επιτυχία την οποία καταφέρνουμε με κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική επιτυχία. Και ένα αυτοκινητόδρομο ο οποίο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ακριβώ επειδή υπάρχουν τέτοιου είδου πρακτικά προβλήματα χρήζει συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν ε, χαιρόμαστε που μπορούμε να, το, να έχουμε αυτή τη συζήτηση εδώ και με εκπροσώπου και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κύριο Ρενό, ο οποίος ε, ε, συμμετείχε και στην Task Force ε, για την Ελλάδα. Χαιρόμαστε που βρίσκεται εδώ η κυρία Πούσιο, η οποία έχει συμμετάσχει και σε μια συγκριτική μελέτη, η οποία είχε γίνει σε ό,τι αφορά τις απαλωτριώσεις και σε άλλα κράτη-μέλη και η οποία μελέτη βέβαια είχε ασχοληθεί και με τα ζητήματα ε, και της Ελλάδας. Ε, χαιρόμαστε που βρίσκεται ο κύριος ε, Δελής εδώ από το Υπουργείο Μεταφορών της Ελλάδας και ο κύριος Ψαθάς που είναι σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών για τα ζητήματα των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Προφανώς θέλουμε να υπάρξει επιτυχία στην Ελλάδα και να υπάρχει και επιτυχής διαχείριση και αξιοποίηση των κορδιλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καθώς υπάρχουν και ε, έργα που τρέχουν στην Ελλάδα με συγχρηματοδότηση του ύψους 100% και αυτά τα έργα θα πρέπει να είναι ορατά. Όμως ε, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται, είναι παρούσα επιτόπου στην Ελλάδα και δαπανά περισσότερα χρήματα για τις απαλωτριώσεις από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και βλέπουμε πως υπάρχουν ακόμη απαιτήσει οι τρέχουν στο πλαίσιο απαλωτριώσεων και βλέπουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση όταν έχει να κάνει με αξιώσει που προέρχονται από ολοκληρώσει που ξεπερνάνε το 10% να είναι υποχρεωμένη να συγχρηματοδοτεί και αυτέ τι ε, περιπτώσει. Ε, να καλωσορίσω τον ε, κύριο Σλότερος, ο οποίο είναι γενικό διευθυντή από την ομάδα τη DG Regio για την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχετε τον λόγο για τη δική σα παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν που οργανώσατε τη σημερινή εκδήλωση και αυτό αποτελεί και μια συνέχεια των όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια τη δική σας αποστολή. Στη δική μου παρέμβαση θα τα πω γρήγορα. Χαίρομαι που έχουμε εδώ μια πολύ εντυπωσιακή παρουσία εμπειρογνωμόνων για θέματα πολιτριώσεων στην Ελλάδα, κάθονται δίπλα μου και θα ήθελα να κάνω μια αναδρομή στην όλη ιστορία αυτής της υπόθεσης, να σας εξηγήσω από πού ξεκινάμε και γιατί θεωρήσαμε πως είναι τόσο σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στο μεγάλο βαθμό στον οποίο σήμερα μας απασχολεί. Λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα στην DG Regio που χρησιμοποίησε και το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ για να χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο αριθμό υποδομών στην Ελλάδα ε, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε το θέμα των απαλωτριώσεων και σε όλη αυτή την περίοδο που ασχοληθήκαμε με το θέμα καταλάβαμε πως οι διαδικασίες απαλωτριώσεων στην Ελλάδα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρες πολύ συχνά ε, κατέληγαν στα δικαστήρια και ξέρετε πως οι δικαστικές αυτές ε, διαδικασίες στην Ελλάδα έτσι και αλλιώς χρειάζονται πολύ χρόνο. Εάν σε αυτό προσθέσουμε και τη δυνατότητα να ακολουθηθεί ε, κάποιου είδους ε, πρωτοβάθμιας προσφυγής από ένσταση, προσφυγή εκ νέου κτλ. Καταλαβαίνετε πως η διαδικασία αυτή χρειάζεται ακόμα περισσότερο χρόνο. Και όπως είπατε κι εσείς, οι τιμές της γης που έχει απαλωτριωθεί ε, ήταν αρκετά υψηλές και βέβαια με μεγάλες διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή και από εποχή σε εποχή. Εμείς μέσω των διαρθωτικών ταμείων ε, πρέπει να σας πω ότι προστατευόμαστε γιατί στον κανονισμό μας έχουμε το όριο του 10% αλλά καταλαβαίνετε πως μπορεί εμείς με τον τρόπο αυτό να προστατευτούμε από τις ψηλές τιμές της γης στην Ελλάδα το δημόσιο χρειάζεται να καταβάλει το υπόλοιπο ε, της αποζημίωσης για την απαλωτρίωση και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. τι κάναμε τα τελευταία χρόνια και να παρουσιάσω τι κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια πιο συγκεκριμένα. Ή μάλλον να το πω καλύτερα τι έκανε η Ελλάδα για το θέμα αυτό τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό το οποίο έχει συμβεί σε μία σειρά υποθέσεων είναι ότι εμείς δώσαμε τη δυνατότητα της προσωρινής κατάληψης γης. Αυτό είναι ένα είδος ε, προσωρινού μέτρου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση όπου μία απαλωτρίωση πραγματικά χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να έρθει σε πέρας. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα ε, μια εταιρεία και για παράδειγμα μια κατασκευαστική η οποία έχει αναλάβει κάποια από τα έργα οδοποιίας στα οποία αναφερθήκατε μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γη στην οποία θα κατασκευάσει τον αυτοκινητόδρομο παρόλο που δεν έχει περατωθεί ακόμα η διαδικασία παλωτρίωσης. Αυτή είναι η μία ε, δράση που αναλάβαμε. Δεύτερον, καταφέραμε να μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό τις προθεσμίες που έχουμε ε, στην δικαστική διαδικασία. Αυτό έγινε μέσω τροποποίησης νομοθεσίας και σίγουρα οι εμπειρογνώμονες που κάθονται δίπλα μου θα σας κάνουν μια πιο λεπτομερή περιγραφή του τι συνέβη, αλλά αυτή η μείωση η σύντμηση των προθεσμιών ε, στην περίπτωση των απολωτριάσεων για συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι πλέον υποχρεωτική και όσο το κατανοώ εγώ τουλάχιστον, δεν είναι όμως τόσο δεσμευτική όταν πρόκειται για έργα τα οποία δεν είναι αντικείμενο συγχρηματοδότησης. Επίσης καταφέραμε να έχουμε αυτή την ανεξάρτητη αξιολόγηση, εκτίμηση, αποτίμηση της γης που πρόκειται να απαλωτριωθεί. Θα θυμόσαστε πως ε, στην Ελλάδα παραδοσιακά μια ε, διαδικασία παλωτρίασης ξεκινούσε από μια τιμή που υπολογίζεται πάνω στην αντικειμενική αξία. Είναι δηλαδή μια αξία την οποία έχει ουσιαστικά ορίσει η εφορία. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτές οι αξίες πολύ συχνά είχαν πολύ μικρή σχέση με την τιμή αγοράς. Άρα λοιπόν οδηγούσαν πολύ συχνά σε προσφυγές από τους ιδιοκτήτες της γης γιατί θέλανε να λάβουν μια υψηλότερη αποζημίωση. Με αυτή τη δυνατότητα ανεξάρτητης αποτίμησης ουσιαστικά έχουμε μια τιμή που ορίζεται ε, βασιζόμενη στον υπολογισμό διεθνώς αναγνωρισμένων παραμέτρων. Και η αποτίμηση αυτή, ακριβώς της αξίας για να είναι ανεξάρτητη, γίνεται από εκτιμητές που προέρχονται από ένα αναγνωρισμένο σώμα εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για να το κάνουν και οι οποίοι έχουν επιστοποιηθεί για να κάνουν τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Τέλος υπάρχει υποχρέωση ο δικαστής ή εν του το δικαστήριο σε περίπτωση που όντως προσφύγει κάποιος κατά της ε, τιμής που ορίζεται από τον ανεξάρτητο εκτιμητή. Έχει λοιπόν την υποχρέωση το δικαστήριο να δικαιολογήσει μια οποιαδήποτε απόκληση από την τιμή που έχει ορίσει ο ανεξάρτητος εκτιμητής. Εάν λοιπόν ο δικαστής θέλει να ορίσει μια υψηλότερη αποζημίωση από αυτή που έχει εκτιμηθεί, θα πρέπει να τεκμηριώσει συγκεκριμένα τους λόγους για τους οποίους οδηγείται σε αυτή την απόφαση. Ενώ στο παρελθόν το δικαστήριο είχε ένα μεγάλο βαθμό ελευθερίας απόκλησης από τις αντικειμενικές αξίες. και οι οποίες θεωρούνται τότε και η βάση για τους υπολογισμού αυτούς. Έτσι λοιπόν αυτά τα μέτρα έχουν ε, ε, επηρεάσει και την όλη διαδικασία, δηλαδή ε, τη διάρκεια της όλης διαδικασίας. Έχουν περιορίσει και το πεδίο για προσφυγές και έχουν δώσει και τη δυνατότητα μιας ανεξάρτητης τεκμηριωμένης αποτίμησης της γης που πρόκειται να παλουτριωθεί. θεωρώ πως αυτό ήδη είναι μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση όπως ήταν πριν από 5-6 χρόνια. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό πως ε, δεν χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις. Θα έλεγα πως κομμάτι αυτών που περιγράφω είναι κάποιες μη δομικές λύσεις. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή η προσωρινή κατάληψη γης. Αυτό γίνεται ε, στα πλαίσια μιας ρήτρα εξαίρεσης και αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί εγκάρσια, γιατί βέβαια τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαίρεση. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος για το μηχανισμό αυτό, εάν ε, συνεχίζουμε να τον χρησιμοποιούμε γιατί είναι χρήσιμος, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ενταχθεί στην συνήθη ε, νομοθεσία που εφαρμόζεται έτσι ώστε να μην εφαρμόζεται ε, στα πλαίσια αυτής της ρήτρα ως εξαίρεση. Κάτι το οποίο επίσης χρειαζόμαστε επιγόντως είναι μια κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα με την νομοθεσία στην Ελλάδα, η οποία είναι εξαιρετικά περίπλοκη και όπου υπάρχουν νομοθετήματα τα οποία πρέπει να κωδικοποιηθούν από τους εμπειρογνώμονες από διάφορους κώδικες έτσι ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ορίζει η νομοθεσία και αυτό ισχύει βέβαια και για την νομοθεσία που διέπει τις απαλωτριώσεις. Και αυτό λοιπόν είναι για μας απαραίτητο έτσι ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωρίζουν σε περίπτωση απαλωτρίωσης τι ακριβώς ισχύει. Η ανεξάρτητη εκτίμηση της τιμής είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ε, και μια κίνηση που μας οδηγεί στο μέλλον. Όμως, ο ανεξάρτητος εκτιμητής θα δώσει μια τιμή η οποία συνήθως απέχει από την αντικειμενική αξία, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία δυνατότητα συζήτησης. Συγκρίνοντας διαφορετικές τιμές για τα ίδια χωράφια, γιατί για τέτοιο πράγμα μιλάμε, θα χρειάζεται και μια πιο ε, δομημένη λύση σε αυτές τις διαφορετικές κατηγορίες τιμών έτσι ώστε οι αντικειμενικές αξίες να προσεγγίσουν τις εμπορικές αξίες ή τις αξίες που θα έδινε ένας ε, ανεξάρτητος εκτιμητής σε ένα κομμάτι γης. Και τέλος, κάτι το οποίο δεν συζητάμε σήμερα αλλά δεν είναι μικρή σημασία, είναι το ότι για να καταλάβουμε τι απαλωτριώνεται θα πρέπει να έχει κανείς ένα πολύ σαφή ορισμό και ε, μητρό που να περιγράφεται κάθε κομμάτι γης. Και βέβαια, για να γίνει αυτό, χρειάζεται ένα κτηματολόγιο λειτουργικό σωστό. Είναι ένα έργο για το οποίο κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες μαζί με την ελληνική κυβέρνηση. πριν να πω ότι είναι άριστη συνεργασία μας, αλλά είναι ένα έργο το οποίο θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί και πάλι είναι ένα κομμάτι αναφέρεται από το σύστημα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι όπως έχει κατάσταση με ό,τι ήδη έχουμε στα χέρια μας, αλλά υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που δεν θα κλείσουν εάν δεν έχουμε ακριβώς αυτό το κτηματολόγιο στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Διαπιστώσαμε λοιπόν όλα όσα δεν λειτουργούν ακόμα σωστά και βέβαια θα πρέπει κάποια στιγμή να αναφερθούμε στα όσα θα πρέπει τελικά να λειτουργούν ε, σωστά. Ε, και βέβαια δεν ακούσαμε κάτι σχετικό. Μήπως λοιπόν θα μπορούσατε να μας ε, πείτε τι κάνει η Επιτροπή από την πλευρά της ούτως ώστε να επιτύχει το να λειτουργήσουν αυτά τα κόμματα λίγο καλύτερα. Μπορείτε να προσθέσετε κάτι ακόμα. Maybe not been uh, enough, Chairman, but Δεχομένως να μην ήμουν απόλυτα σαφή, κυρία Πρόεδρε. Πολλά πράγματα έχουμε κάνει προκειμένου να προωθήσουμε μία σειρά από λύσεις. Λύσεις οι οποίες ήδη έχουν εντοπιστεί, όπως για παράδειγμα το να δίνεται η δυνατότητα προσωρινής κατάληψης γης, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή πιο ευραία. Έχουμε συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να δημιουργηθεί μια διπουργική επιτροπή η οποία επιβλέπει μια σειρά από σημαντικά έργα και η οποία διπουργική επιτροπή πρόσφατα σε πολλές περιπτώσεις αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό αυτό της προσωρινής κατάληψης γης προκειμένου να προχωρήσουν διάφορα έργα. Έχουν γίνει επίσης και νομοθετικές και νομικές αλλαγές, στις οποίες αναφέρθηκα, όπως για παράδειγμα όσον αφορά τις προθεσμίες για τη δικαστική διαδικασία ή όσον αφορά την δημιουργία του σώματος πιστοποιημένων εκτιμητών, ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται αυτοί οι εκτιμητές. Όλες αυτές οι νομοθετικές τροποποίησεις γίνανε με την βοήθεια, με την πίεση που άσκησαν οι υπηρεσίες μας. Θα συνεχίσουμε προφανώς τη συνεργασία αυτή, θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση, ιδίως όσον αφορά την ε, ευθυγράμμιση και τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας και προσπαθώντας να βρούμε πιο διαρθρωτικές ε, λύσεις, ιδίως μέσω της κωδικοποίησης της ελληνικής νομοθεσίας. Και προσπαθώντας παράλληλα να έχουμε μια πιο διαρθρωμένη πλέον εφαρμογή μιας διαδικασίας που αυτή τη στιγμή θεωρείται εξαιρετική διαδικασία, διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατ' εξαίρεση. Αναφέρουμε για παράδειγμα στην προσωρινή κατάληψη γης. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μόνο κατ' εξαίρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικώ και ευρέω αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια γιατί ενδεχομένως να μην θεωρείται ακόμα συνταγματική, ενδεχομένως επειδή μια τέτοια μέθοδος βάλει κατά συγκεκριμένων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε αυτή τη στιγμή να βρούμε μια πιο οριστική λύση. Δεν είναι εύκολο βέβαια το χείρημα αυτό, αλλά θα συνεχίσουμε εμείς να ασκούμε πίεση προκειμένου να επέλθουν περαιτέρω τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία, προκειμένου να καταλήξουμε τελικά σε έναν μόνιμο μηχανισμό όπως αυτός της προσωρινής ε, κατάληψης γης, ο οποίος όμως δεν θα έχει προβλήματα έκτακτης ε, εφαρμογής ή κατεξαίρεση μόνο εφαρμογής. Και για να γίνω ακόμα πιο σαφής ε, σε σχέση με αυτά που είπα για το κτηματολόγιο, το κτηματολόγιο αποτελεί για μας ένα πολύ σημαντικό έργο για την Ελλάδα, αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα η οποία χρηματοδοτείται από τα κοινοτικά κονδύλια. Προβεβλημένη λοιπόν προτεραιότητα η οποία θεωρούμε ότι μπορεί κατά τρόπο πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να βοηθήσει την κατάσταση και να καταστήσει τελικά τη διαδικασία παλωτριώσεων στην Ελλάδα πολύ πιο ομαλή και πολύ πιο σύντομη. Ακριβώς επειδή θα παράσχει μια καλύτερη περιγραφή των φυσικών πτυχών των ε, κτημάτων της ακίνητης περιουσίας και επίσης θα είναι πολύ δύσκολο να τεθούν να αμφιβόλου οι προτινόμενες εκτιμόμενες τιμές για τις συγκεκριμένε εκτάσεις, εφόσον δηλαδή υπάρξει ένα πλήρες κτηματολόγιο, αλλά το σχέδιο είναι ακόμα μακρόπνο, θα απαιτηθεί χρόνος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Ρενό, ο οποίος είναι αρμόδιος ε, για ζητήματα πολιτικής ε, από τη Μονάδα για την Καταπολέμηση της Απάτης και ο οποίος συμμετείχε επίσης στην Task για την Ελλάδα. Παρακαλώ. Thank you. Um, uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή σας που με προσκάλεσε σήμερα για να μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό των απαλωτριώσεων. Όντω εργάζομαι για την ε, υπηρεσία υποστήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υπηρεσία αυτή αποτελεί συνέχεια τη Task Force που είχε συσταθεί για την Ελλάδα και η οποία είχε ασχοληθεί με ζητήματα τεχνική υποστήριξη προκειμένου να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση αλλά και άλλοι τομεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί σήμερα και το οποίο έχει να κάνει πιο συγκεκριμένα με τις απαλωτριώσεις, θα ήθελα προφανώς να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα. Όντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέβαλε με την συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης στην προώθηση διαφόρων δράσεων κατά της διαφθοράς, οι οποίες με την σειρά του συνέβαλαν στη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά τις απαλωτριώσεις η Task Force για την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άσκησαν πίεση προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια συγκεκριμένη στρατηγική για την Ελλάδα, η οποία εγκρίθηκε και από την Όλαφ και που πήρε τη μορφή συγκεκριμένων συστάσεων όσον αφορά την κατάσταση των απαλωτριώσεων στην Ελλάδα και που οι συστάσεις αυτές οδήγησαν στις τροποποίησεις νομοθεσίες, οποίες αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κύριος Λόιτερς. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, θα ήθελα και εγώ να περάσω τώρα στη δική μου την παρουσίαση, πώς έχει κατάσταση στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε και το είδατε κι εσείς οι ίδιοι όταν πήγατε στην Ελλάδα, όταν πήγατε στην Αθήνα, ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες οι οποίες συνδέονται με τις απαλωτριώσεις, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία έργων υποδομών στην Ελλάδα. Έτσι έχει κατάσταση αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις αλλά και σε περαιτέρω δαπάνες για τα έργα αυτά. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και νομίζω ότι και ο Βιλ Μπροτ το είπε πριν από λίγο, είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί στην κατάσταση αυτή για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Βραχυπρόθεσμα μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι έχουν λυθεί τα περισσότερα προβλήματα όσον αφορά τις απαλωτριώσεις στην Ελλάδα. Θα επανέλθω στο σημείο αυτό. Οφείλω πάντως να πω ότι όντως η ελληνική κυβέρνηση άρχισε να χρησιμοποιεί πιστοποιημένους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες προβλέπονται νέες διατάξεις όσον αφορά τη λειτουργία των δικαστών, πώς μπορούν αυτοί να πάρουν ανεξάρτητες αποφάσεις για την τιμή των ακτιμάτων και ξέρετε ότι υπάρχει και μια επιταχυμένη διαδικασία μέσω της λεγόμενης Ολυμπιακής νομοθεσίας που έχει ως στόχο να επισπεύσει την όλη διαδικασία απόκτησης γης. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σας προτείνω και να σας παρουσιάσω τα εξή σημεία. Πρώτον, κάποιες γενικές παρατηρήσεις που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, για ποιο λόγο οι απαλωτριώσεις αποτελούν πολλές φορές πηγή καθυστερήσεων και δαπανών στα πλαίσια των έργων υποδομών και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και φαινόμενα διαφθοράς και αυτό έχει να κάνει πολλές φορές με τα υποκείμενα κίνητρα που υπάρχουν στα έργα αυτά. Όπως είπε και ο Βιλ Μπρόντους πριν από λίγο, θα αναφερθώ και στην αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης και πώς προσπάθησε να θεραπεύσει την κατάσταση και θα ήθελα στη συνέχεια να δούμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση των απαλωτριώσεων. Όσον αφορά τις απαλωτριώσεις ε, ως πηγή καθυστερήσεων και δαπανών, στον τομέα στον κλάδο των πολιτικών μηχανικών. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό βέβαια, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει και προκύπτει συνεχώς και στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου. Η Task Force δεν έκανε μια συγκεκριμένη έρευνα όσον αφορά την Ελλάδα, επομένως οι συστάσεις που βλέπετε στη στρατηγική κατά της διαφθοράς των κοινοτικών κονδυλίων έχουν να κάνουν μια γενικότερη ανάλυση που κάναμε, η οποία συνδέθηκε με μελέτες που είχαν γίνει από τις ελληνικές αρχές όσον αφορά τη συγκεκριμένη ελληνική κατάσταση. Προκειμένου όμως να καταλάβουμε ακριβώς πώς έχει κατάσταση με την απαλωτρία, θα ήθελα να αφαιρθώ στην περίπτωση της Γαλλίας. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας πω πώς, ε, πώς δημιουργήθηκαν τα πράγματα, πώς είχαν παλαιοτριώσεις όταν δημιουργήθηκε το σύγχρονο Παρίσι. Θα ήθελα να αφαιρθώ λοιπόν σε ένα βιβλίο του Εμίλ Ζολά που ονομάζεται «The Kill, La Cure» στα γαλλικά και που αναφέρεται στην εποχή εκείνη που ο Βαρόνος Οσμάν δημιουργούσε το σύγχρονο Παρίσι, τη σύγχρονη ρημοτομία του Παρισιού όπως τη γνωρίζουμε σήμερα και αναφέρεται αν θέλετε στους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της εποχής εκείνης. Πώς έχουν λοιπόν τα πράγματα, θα αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα σημεία. Η απαλωτρίωση έχει αποτελέσει αντικείμενο, ή τουλάχιστον την εποχή εκείνη αποτελούσε αντικείμενο απάτη. Καταρχά είχαμε πολλά φαινόμενα χρησιμοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών. Ορισμένοι γνωρίζαν ακριβώ, για παράδειγμα πού θα δημιουργείται μια συγκεκριμένη λεωφόρο στο Παρίσι και θα φρόντισαν εκ των προτέρων να πουλήσουν εκτήματα στην περιοχή αυτή προκειμένου να κερδίσουν από την προστιθέμενη αξία της πώληση αυτής και από την αύξηση της τιμής που θα είχαν οι περιοχές αυτές. Η δεύτερη μορφή απάτης έχει να πουλησουν εκτηματα στην περιοχη αυτη προκειμενου να κερδισουν απο την προστιθεμενη αξια τη πωληση αυτή και απο την αυξηση τη τιμή που θα ειχαν οι περιοχέ αυτέ. η δευτερη μορφη απατης εχει να κανει με την ίδια την τιμή της ακίνητης περιουσίας. Την εποχή εκείνη δεν είχαμε ένα συγκεκριμένο σαφές μητρό κτημάτων στην Γαλλία. Επομένως, μπορούσε πάρα πολύ εύκολα κανείς να πει ότι σε μια συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε απλώς ένα σπίτι, μια κατοικία, αλλά μια επαγγελματική κατοικία. Δημιουργούσε δηλαδή ένα ψευδές μητρό τελικά, προκειμένου να αποδείξει ότι υπήρχαν διάφορες ε, βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες σε μια συγκεκριμένη περιοχή και ότι η τιμή της συγκεκριμένη περιοχής είχε πολύ ψηλότερη αξία από ότι η αντικειμενική αξία την εποχή εκείνη. Επομένω, είχαμε τέτοια φαινόμενα πάθη όσον αφορά την αξία τη ακίνητη περιουσία. Επίση, είχαμε και πάρα πολλέ καθυστερήσει και ξέρετε στον κλάδο των πολιτικών μηχανικών αυτό μα απασχολεί όλο ιδιαίτερο. Στην εποχή λοιπόν εκείνη υπήρχαν ορισμένε εταιρείε ή νομικά γραφεία τα οποία Συναντούσαν κατόχους ιδιώτες διαφόρων τέτοιων περιοχών που επρόκειτο να απαλωτριωθούν και τους έλεγαν δεν θα πρέπει να συμφωνήσουν με αυτή την απαλωτρίωση. Στη συνέχεια πήγαν και έβλεπαν και έναν δικαστή και πολλές φορές χρηματοδοτούσαν τον δικαστή αυτό προκειμένου να καθυστερήσει τη δικαστική διαδικασία. Και Μέσω δωροδοκίας επίσης μπορούν να επηρεάσουν τόσο την αποτίμηση της αξίας εκείνης της περιουσίας ή να επηρεάσουν ακόμα και την ίδια την απόφαση του δικαστή. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι υπήρχαν πολλά διαφορετικά κίνητρα. Κάθε φορά που υπάρχει ένα συγκεκριμένο έργο πολιτικών μηχανικών, η καθυστέρηση μπορεί πραγματικά να αποτιμηθεί σε ένα πολύ σημαντικό ποσό. Η καθυστέρηση αυτή μπορεί να αποτιμηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εξαρτάται από το πόσες μέρες καθυστερεί τελικά ένα έργο. Κάθε φορά λοιπόν που έχουμε μια σύμβαση παραχώρησης ή ένα κατασκευαστικό έργο το οποίο έχει αναλάβει ο ιδιωτικό φορέα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα προκειμένου η διαδικασία να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα. Επομένω, οι καθυστερήσει λειτουργούν σε συγκεκριμένη περίπτωση ιδιαίτερα αρνητικά. Να λοιπόν πώ είχαν τα πράγματα την εποχή εκείνη, στο Παρίσι του 19ου αιώνα. Κάθε φορά που εξετάζουμε λοιπόν την περίπτωση των απαλωτριώσεων, βλέπαμε ότι προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στην Ελλάδα, αναφέρομαι σε προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει ή εξακολουθούν και προκύπτουν σε πάρα πολλέ χώρε τη Ευρώπη και εκτό. Σαφώ η διαδικασία τη απαλωτρίωση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη από νομοθετική ε, πλευρά και πολλέ φορέ όταν προσπαθούμε να αποτιμήσουμε την αξία τη γη, Υπάρχουν ε, πάρα πολλέ εκπλήξει που μπορούν να προκύψουν και πάρα πολλέ καθυστερήσει, οι οποίε μπορεί πολλέ φορέ να είναι και συναισθηματικά φορτισμένε. Ιδιώτε δηλαδή οι οποίοι δεν θέλουν να πουλήσουν τη γη του. Από προσωπική πλευράς πιστεύω ότι ε, η ελληνική ανταπόκριση στην κατάσταση αυτή έδωσε μια αξιόλογη λύση τουλάχιστον ε, βραχυπρόθεσμα. Θα ήθελα καταρχάς λοιπόν να αναφερθώ στην χρήση υπάρξει να γίνεται από πιστοποιημένους εκτιμητές. Μια διαδικασία που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2013 τροποποιήθηκε η νομοθεσία προκειμένου να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένοι εκτιμητές. Είναι περίπου 300 αυτοί οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, άνθρωποι, εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα και την επίσημη πιστημο... Ε, πιστοποίηση να κάνουν αποτίμηση, εκτίμηση αξίας ακινήτων. Ακολουθούν ένα συγκεκριμένο δοντολογικό κώδικα, και για τα μεγάλα έργα υποδομή μπορούν να εμπλέκονται ακόμα και τρει τέτοιοι εμπειρογνώμονε, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτίμηση τη αξία τη ακίνητη περιουσία. Έχουμε ένα υψηλό επίπεδο λοιπόν επαγγελματισμού αλλά και ανεξαρτησία όσον αφορά την αποτίμηση τη τελική τιμή. Η δεύτερη πολύ σημαντική απόφαση που ελήφθηκε από την ελληνική πλευρά ήταν το ότι θα έπρεπε οι αποφάσει των δικαστών είναι πλέον πλήρω αιτιολογημένε. Ο δικαστή στο τέλο τη δικαστική διαδικασία πρέπει να πάρει μια τελική απόφαση και να αποκλίνει από την τιμή που έχουν προτείνει οι εμπειρογνώμονε, το είπε και ο προλαλή σα, πρέπει να παράσχει μια πλήρη αιτιολόγηση. Καταλαβαίνετε ότι το περιθώριο μου περιορίζεται σε σχέση με το παρελθόν. Κάτι το οποίο δεν έχω καταγράψει στην παρουσίασή μου και θα έπρεπε να το είχα συμπεριλάβει είναι ότι το 2014, αν δεν κάνω λάθος, λίγο πριν τη δική σας την επίσκεψη, αποφασίστηκε από τις ελληνικές αρχές να μην ζητούν πλέον από τον δικαστή να λάβει μια απόφαση για την τιμή, αλλά να βασίζονται μόνο στην τελική απόφαση του εφετείου. Κατά αυτόν τον τρόπο εμπλέκονται λιγότεροι δικαστές στην όλη διαδικασία καθορισμού της τιμής και κατά αυτόν τον τρόπο έχει μειωθεί και η διακύμαση των προτινόμενων τιμών. Και έχουμε τέλος και την Ολυμπιακή νομοθεσία, συγκεκριμένη η οποία εγκρίθηκε για τα Ολυμπιακά έργα και η οποία είχε ως στόχο να επισπευθεί η ε, κατοχή της ε, ακίνητης περιουσίας και χρησιμοποιήθηκε η νέα αυτή νομοθεσία κυρίως για τα μεγάλα έργα υποδομής. Οι Έλληνες ε, συνάδελφοι θα μας δώσουν για αυτά περισσότερες πληροφορίες. Καλύπτονται πολλά έργα από τη νέα αυτή νομοθεσία και από πρακτικής πλευράς Αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι μια έκταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για λόγους δημόσιοφελίας και αυτή τη στιγμή γίνει μια αποτίμηση της τιμής και υπάρχει και ένα ποσό το οποίο μπορεί να δοθεί ως αποζημίωση πλέον στον ιδιοκτήτη, μπορεί να κατασχεθεί η έκταση αυτή και μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να ξεκινήσει το κατασκευαστικό έργο. Κατά αυτόν τον τρόπο μειώνονται πάρα πολύ οι απαιτούμενε ε, χρονικές περίοδοι προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο, Συντομεύεται λοιπόν η όλη διαδικασία πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Οι Έλληνε πάντω θα μα δώσουν για αυτά περισσότερε πληροφορίε. Ολοκληρώνοντα, πρέπει να σα πω ότι μολονότι μέσω των λύσεων αυτών η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να επιλύσει γρήγορα μια πολύ δύσκολη κατάσταση που είχε προκύψει, παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα κάποια όρια στι προτινόμενε αυτέ λύσει. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι η νομοθεσία για τα Ολυμπιακά έργα έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογή. Δηλαδή όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα και όσον αφορά τα έργα τα οποία καλύπτει. Υπάρχουν ε, ακόμα πολλά έργα τα οποία καλύπτονται από νομοθεσία αυτή, αλλά και πολλά άλλα τα οποία δεν μπορούν να αποφεληθούν από την νέα αυτή νομοθεσία. Και επίσης ε, το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται αυτή τη στιγμή είναι αρκετά περιορισμένο και πρέπει να γίνουν ε, και κάποιες τροποποιήσεις στην όλη αυτή νομοθεσία προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και στο μέλλον. Και παρόλα αυτά Μολονότι έχουμε νομοθεσία αυτή, υπάρχουν ακόμα μεγάλε διακοιμάνσει όσον αφορά την εκτιμόμενη τιμή, οπότε και αυτό πρέπει να μα απασχολήσει περισσότερο. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιε πιο μόνιμε λύσει. Θα ήταν καλό να υπήρχε μια τυποποιημένη διαδικασία όσον αφορά την εκτίμηση του κόστου. Μια τυποποιημένη διαδικασία που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πιστοποιημένοι εκτιμητέ και από την άλλη θα ήταν καλό να υπήρχε και μια κοινή βάση δεδομένων όσον αφορά τι εκτιμόμενε αυτέ τιμέ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να καταγράψουμε όλες αυτές τις τιμές πώληση και απαλωτρίωσης, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από τους εμπειρογνώμονες και στο μέλλον. Επίσης, η ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Πρέπει προφανώς να ακολουθούν κάποιους δεοντολογικούς κανόνες, τους οποίους ασπάζονται τη στιγμή που εντάσσονται στο επάγγελμα αυτό, αλλά κάθε φορά που έχουμε προσφυγές θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ολοκληρωθούν οι σχετικέ δικαστικέ διαδικασίε αν κάθε εμπειρογνώμονα είχε υπογράψει μια δήλωση απουσία σύγκρουση συμφερόντων για κάθε έργο. Και νομίζω επίση ότι θα μπορούσαν να είχαν υποβάλει και μια δήλωση περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου σε κάθε περίπτωση να μπορεί να αποδεικνύει το ελληνικό κράτο ότι δεν υπήρχε περίπτωση κερδοσκοπία εκ μέρου ενό εμπειρογνώμονα. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προσαρμόσουμε την νομοθεσία των Ολυμπιακών έργων ώστε να αποτελεί πλέον μια τυποποιημένη διαδικασία που θα επιτρέψει την κατοχή της ακίνητης περιουσίας κατά τρόπο πολύ πιο διαφανή και πολύ πιο αποτελεσματικό. Θεωρώ λοιπόν ότι η προβλεπόμενη από τη νέα αυτή νομοθεσία διαδικασία θα πρέπει να παγιοποιηθεί και να αποτελέσει πλέον μόνιμη πλατφόρμα όσον αφορά τη διαδικασία των απαλωτριώσεων. Τέλος, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά στο κλιματολόγιο και όσον αφορά στα χωροταξικά σχέδια, προκειμένου να έχουμε μία καλύτερη εκτίμηση της αξίας των διαφόρων κτημάτων στην ελληνική επικράτεια. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν θα επαφιόμαστε κάθε φορά στην χρήση που έχει κάνει ο εν λόγω ιδιοκτήτης, αν για παράδειγμα έχει φυτέψει συγκεκριμένη περιοχή με δέντρα ή οποροφόρα ή αν έχει κτίσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πιο αντικειμενικό τρόπο περιγραφής της χρήσης της γης μέσω του κτηματολογίου και μέσω των χωροταξικών σχεδίων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάντως τις ελληνικές αρχές για την οικοδομητική του στάση, έχουν ήδη κάνει πολύ σημαντικά βήματα και απλώς πρέπει να βελτιωθεί τώρα η κατάσταση με περαιτέρω αποφάσεις. Φάτος βρίσκονται στο σωστό δρόμο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία που μας ε, κοινοποιήσατε. Διαπιστώνουμε ότι ε, όταν επιβάλλεται μια ε, νομοθεσία χωρίς να υπάρχει κάτι ε, προηγουμένως ε, είναι πάντα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χαίρομαι που είναι σήμερα μαζί μας εδώ η κυρία Πότση, η οποία ήταν μία από τους συντάκτες της εκδικής έκθεσης ό,τι αφορά την νομοθεσία για τις απαλωτριώσεις της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δίνουμε κατευθείαν το λόγο. Καλησπέρα. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ σήμερα εδώ και θα προσπαθήσω μέσα σε λίγα λεπτά να σας κάνω την παρουσίασή μου. Καταρχήν να σας συστηθώ, λέγομαι Χρυσή Πότσιου, είμαι επίκουρη καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ε, ε, όπου διδάσκω μεταξύ άλλων και ε, χωροταξικό συνδυασμό και εκτίμηση ακινήτων και είμαι πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Τοπογράφων, οπότε ως πρόεδρος αυτής της Ένωσης ε, γνωρίζω πολλές από τις έρευνες οι οποίες έχουν ε, διεξάχνει ε, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων στην οποία συμμετέχουν βέβαια τοπογράφοι από όλο τον κόσμο και να σας πω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή, πολύ χρήσιμη δημοσίευση την οποία μπορείτε να αναζητήσετε μέσω Google και να την κατεβάσετε η οποία περιγράφει τις ευέλτιστες πρακτικές των καλύτερων εμπειρογνωμών μας από αυτό το τομέα. Καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά λοιπόν σε αυτό το έγγραφο. Θα ήθελα να σας αναφέρω περιληπτικά, με βάση και την εμπειρία που έχω, ε, το τι συμβαίνει διεθνώς και τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Με βάση λοιπόν τις έρευνες που έχουμε κάνει στην ε, Διεθνή Συνομοσπονδία των ε, τοπογράφων, οι βέλτιστες πρακτικές είναι εκείνες που εφαρμόζονται στις χώρες που προτιμούν την άμεση αγορά. Υπάρχει εκτεταμένη εμπειρία δηλαδή σε αυτό το τομέα, ειδικότερα με φιλικούς διακανονισμούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται χρήματα, εξοικονομείται χρόνος και το κυριότερο ε, διασφαλίζεται έτσι η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κρατικό μηχανισμό. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η καταναγκαστική απαλωτρίωση είναι μια, ένα πολύ ευαίσθητο, λεπτό ζήτημα, γιατί στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς βασιζόμαστε ε, πάρα πολύ και στην εύρυθμη λειτουργία της ε, αγοράς ακινήτων και κατά συνέπεια βασιζόμαστε και πολύ στις επενδύσεις ε, σε ακινητά. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια στο πλαίσιο νομική δηλαδή ασφάλεια, στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι συχνά υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Για παράδειγμα, υπάρχει δηλαδή ένα επενδυτή ο οποίο έχει επενδύσει σε ένα ακίνητο και ε, θέλει να είναι σίγουρος ο λόγο επενδυτής ότι μπορεί να εμπιστευτεί την κυβέρνηση. Ότι δηλαδή έκανε μια σωστή επένδυση και ότι το κράτος θα ε, προστατεύσει αυτή την επένδυση και την ιδιοκτησία. Από την άλλη πλευρά, προφανώ ε, ε, υπάρχει και το κράτο το οποίο θέλει να προβλήσει σε κάποια δημόσια έργα, υπάρχουν κάποια, κάποια συγκεκριμένα κονδύλια που πρέπει να απορροφηθούν και κάποιε συγκεκριμένε προθεσμίε που θα πρέπει να τηρηθούν. Και ακριβώ γι' αυτό είναι τόσο λεπτό το ζήτημα. Στι περισσότερε λοιπόν χώρε όπου υπάρχουν καλέ εμπειρίε με τι απολωτριώσει, ε, βασίζονται συχνά σε φιλικού διαγωνισμού. Και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρχει καλό μηχανισμό εκτίμηση, ούτω ώστε να συμφωνούν και τα δύο μέρη σε αυτήν την τιμή, την εκτιμόμενη τιμή και επίση, στο πλαίσιο αυτή τη συσβέντη πρακτική ανήκει και το να καταβάλλεται και η αποζημίωση πριν από οποιοδήποτε κατάληψη ε, τη γη. Γιατί ε, θα πρέπει να έχουμε κατά ότι προφανώ κάποιο προβαίνει σε μια επένδυση σε ένα οικόπεδο, σε ένα κινητό και πρόκειται για μια περιουσία με την οποία μπορούν να λάβουν ένα δάνειο, με την οποία μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους, των οικογενειών τους, την εκπαίδευση των παιδιών τους και ούτω καθεξής. Άρα, όταν υπάρχει καταναγκαστική ε, τέτοια απαλωτρίωση, τότε θα πρέπει να ε, καταβάλλεται και άμεσα η αποζημίωση. Προτού δηλαδή γίνει αυτή η κατάληψη, Ακριβώ προκειμένου ο ιδιοκτήτη μπορεί να, ξεκινήσει μια άλλη επιχειρησιακή δραστηριότητα ή, για παράδειγμα, να βρει μια άλλη ε, κατοικία. Άρα λοιπόν αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία στο πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν ε, οι άλλες χώρες έχουν ε, δημιουργήσει και άλλα πρόσθετα εργαλεία σε ό,τι αφορά την κατάληψη. Ε, για παράδειγμα υπάρχει ανταλλαγή των Αγιών και επίσης και υπάρχει και ο αναδασμός ο οποίος προωθείται πάρα πολύ και από τη Γερμανία. Και η, η δηλαδή ο ανακαθορισμός των δικαιωμάτων χρήσης των, της υγείας αυτής και έχω ακούσει επανειλημμένο ότι υπάρχουν πολύ καλές εμπειρίες με αυτούς τους μηχανισμούς. Και η τελευταία επιλογή είναι η καταναγκαστική απαλωτρίωση. Τώρα, περνώντα στην Ελλάδα, ποια είναι η πρακτική που εφαρμόζεται εδώ. Ε, έχουμε πολύ εκτεταμένους ε, περιορισμούς σε ό,τι αφορά την χρήση των διών, οι οποίες όμως δεν μας απασχολούν πότε σε ό,τι αφορά και τον αντίκτυπο, σε ό,τι αφορά την αξία ε, τη γη και δεν προβλέπονται οι σχετικέ αποζημιώσει εκτό κι αν οι άνθρωποι προσφύγουν στα εθνικά και στα δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε, όταν έχουμε μια καταναγκαστική απαλωτρίωση ε, ή αποζημίωση, ε, καταβάλλεται πάρα πολύ αργά. Υπάρχει και αυτή η αποζημιωση καταβαλλεται παρα πολυ αργα υπαρχει και αυτη τη αρχη της αυτό. Αποζημίωσης δηλαδή, ε, όταν ένα κομμάτι απαλωτριώνεται, τότε το υπολοιπόμενο, το υπολοιπόμενο ακίνητο ε, θεωρείται πως έχει κερδίσει περισσότερη αξία και γι' αυτό ε, καταβάλλεται χαμηλότερη αποζημίωση. Ε, πράγμα όμως που δεν ισχύει πάντοτε. Και επίσης υπάρχει και το ζήτημα του χωροταξικού σχεδιασμού που επηρεάζει τις απαλωτριώσεις, για παράδειγμα όταν μια περιοχή εντάσσεται στο σχέδιο πόλης. Μετά, σε ό,τι αφορά την άμεση αγορά ε, εδώ ουσιαστικά αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Και αυτό γιατί, γιατί η πλειοψηφία των πολιτών δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση, ακριβώ γιατί υπάρχει και αυτή η μεταχείριση ό,τι αφορά του τύπου ιδιοκτησία. Και από εκεί και μετά ε, οι εκπρόσωποι ε, του κράτου είναι φοβισμένοι. Δεν έχουν δηλαδή ε, τι αρμοδιότητε για να προβαίνουν στι σχετικέ αποφάσει, να λένε ότι αυτή είναι η πραγματική αξία του ακινήτου. Φοβούνται δηλαδή ότι θα οδηγηθούν στο δικαστήριο, θα του κατηγορήσει κάποιο ότι έχουν δωροδοκηθεί και ούτω Χωρίς αυτό να ισχύει φυσικά. Προφανώς μπορεί να ε, συμβαίνει ενίοτε να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, αλλά δεν αποτελούν αυτά τον κανόνα. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την ανταλλαγή γεών, εμεί έχουμε ξεκινήσει στην Ελλάδα ε, την ανάπτυξη του σχετικού εργαλείου στο κτηματολόγιο για να είναι δυνατό κάτι τέτοιο, αλλά ακόμα δεν έχουμε επιτυχία. Πολύ μεγάλη πρόβλημα. Άρα λοιπόν τα προβλήματα και αδυναμίες του συστήματος στην Ελλάδα που αναγνωρίστηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης είναι ότι για όλα στην Ελλάδα θα πρέπει να υπάρξει μια δικαστική διαδικασία. Λέμε ότι δεν υπάρχει κλιματολόγιο, ναι, ακόμα. Αλλά ε, προκειμένου να γίνει αυτή η επιδίκαση σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να, ε, υπάρξει και συνεδρίαση δικαστηρίου και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή όπως είπαμε στην αρχή, ε, κάποιες χώρες όπου μόνο το 1 με 2% των περιπτώσεων καταλήγουν στα δικαστήρια. Ενώ στην Ελλάδα το 100% των περιπτώσεων πρέπει ακριβώς να περάσει δια ε, ε, να διέρχεται διά της δικαστικής οδού και γι' αυτό βέβαια είναι πολύ φορτωμένα τα δικαστήρια και δεν υπάρχει και κάποιο εξειδικευμένο δικαστήριο για τις απαλωτριώσεις θα πρέπει λοιπόν να απευθύνονται κανονικά στα δικαστικά δικαστήρια ε, Επίση, σε ό,τι αφορά την εκτίμηση τη αποζημίωση, και άλλοι ε, πρέπει να απευθυνθούν στα δικαστήρια. Ακριβώς γιατί η εκτίμηση της ε, αποζημίωσης ε, γινόταν με βάση τις προηγούμενες αξίες χωρίς δηλαδή να σχετίζονται αυτές οι τιμές με την τρέχουσα αξία του ακινήτου. Και βέβαια θα πρέπει ταυτόχρονα σε μια παλωτρίωση να λαμβάνονται υπόψη και συμπληρωματικέ δαπάνε, πέραν δηλαδή από την αξία του ακινήτου, την τρέχουσα αξία. Άρα λοιπόν γι' αυτό αυτέ είναι οι αδυναμίε και προφανώ υπάρχουν και αδυναμίε στον νόμο του 2000, στον κώδικα του 2001 σε ό,τι αφορά τι ε, διαδικασίε ε, και οι οποίε εν μέρει διορθώθηκαν με τον νέο νόμο του, του 4070. Υπήρχαν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την διαφάνεια τη διαδικασία των απαλωτριώσεων, όπου έχουν επιτευχθεί κάποιε βελτιώσει ακόμα συνεχίζονται και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις διοικητικέ δυνατότητες τι δυνατότητε δηλαδή του κρατικού μηχανισμού. Επίση, ε, δεν υπάρχει επαρκή κρατική χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται ανέκαθεν στην Ελλάδα και ακριβώ και γι' αυτό δεν, δεν έχει δοθεί και κατάλληλη έμφαση σε ό,τι αφορά τι ε, αποζημιώσει, την κατάλληλη του γεών και Και αναφερθήκαμε ήδη στο φαινόμενο ε, του υπερβολικού φόρτου εργασία των ε, δικαστηρίων. Και βέβαια υπάρχει ε, και αστάθεια, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο κοινωνική, γιατί υπάρχουν όλε αυτέ οι απεργίε που επηρεάζουν και την εκδίκαση των υποθέσεων και ούτω καθεξή. Είχαμε τώρα ε, και τι ειδικέ τροποποιήσει των νόμων ε, ακριβώ για να ε, λάβουν χώρα τα τα έργα για τις Ολυμπιακές υποδομές. Βέβαια αυτό αποτελούσε μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση, αλλά είχαμε, καταφέραμε έτσι να κλείσουμε την κατάλληλη εμπειρία και έτσι φτάσαμε στον νόμο 4070 του 2012 και ο οποίος βελτίωσε τον εφιστάμενο νόμο του 2001. Οι ε, βελτιώσεις οι οποίες ε, έγιναν ε, πρόβλημα μεταξύ άλλων τον αριθμό των εμπλεκόμενων αρχών, την τροποποίηση της τη διαδικασία χαρτογράφηση για το κτηματολόγιο, το να μπορούν να τρέχουν παράλληλα οι διαδικασίε παροτρύνση και αποζημίωση, έγιναν βελτιώσει ό,τι αφορά του ελέγχου που θα πρέπει να γίνονται από τη διδασκομική υπηρεσία ε, βελτιώσει σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εκτίμησης, ε, γιατί ε, επιτρέπεται πλέον η εκτίμηση να γίνεται και από ανεξάρτητους ελεύθερους επαγγελματίες εκτιμητές και επίσης προβλέπει ο νέος νόμος τη δυνατότητα κατάληψης αυτής της γης προτού ακόμα αποφασιστεί και καθοριστεί η τελική, το τελικό ύψος της ε, αποζημίωσης. Όπως βέβαια ήδη ανέφερα, αυτό δεν μπορεί να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά εδώ προβλέφθηκε αυτή η δυνατότητα ε, γιατί ακριβώ βρισκόμαστε υπό πολύ ειδικέ ε, συνθήκε στην Ελλάδα. Δηλαδή μια τέτοια δικασία επί τη αρχή αντιβαίνει στι βέλτιστε πρακτικέ. Και επίση υπήρξαν και βελτιώσει ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα και ό,τι καθεξή. Υπήρξε λοιπόν κάποια πρόοδο. Από εκεί και μετά ε, ε, ε, έκανα μία ακόμα έρευνα σε ό,τι αφορά απαλωτριώσεις κανονικές, αν θέλετε, όχι δηλαδή για στατικές επενδύσεις και διαπιστώσαμε εκεί, διαπίστωσα σε αυτή την ενημερίδα ότι χρειάζεται, χρειάζεται τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί κανονική μια κανονική διαδικασία απαλωτρίωσης. Άρα προφανώς υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Όμως τονίζω ότι εάν δεν προωθήσουμε το μηχανισμό του φοινικού οικονομισμού, δεν θα μπορέσουμε εδώ να επιτύχουμε μεγάλη πρόοδο, δηλαδή πολύ συντομότερη διαδικασία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η δικαστική διαδικασία είναι πάντοτε ακριβή και είναι πάντοτε χρονοβόρα. Τώρα, η, τα, τι μας πρότειναν οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτήν την, ε, στην ε, μελέτη. Καταρχήν, ε, μας πρότειναν να αυξήσουμε το ρόλο της δημόσιας διαβούλευσης ε, και ενημέρωσης ε, του κενού. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες ξεκινάει αυτή η διαδικασία διαβούλευσης και ενημέρωσης πριν από την διαδικασία της απαλωτρίωσης. Πρέπει δηλαδή να συμμετέχει το ευρύ κοινό σε ό,τι αφορά το πώ ακριβώ θα υλοποιηθεί το έργο, να ενημερώνονται και οι πολίτε σε ό,τι αφορά το ρόλο που μπορούν να παίξουν και τα δικαιώματα που έχουν. Ε, μία ακόμα σύσταση των εμπειρογνωμόνων ήταν να υπάρξει ε, συντονισμός των τεχνικών προδιαγραφών, δηλαδή τεχνικής φύσης αυτή η σύσταση, δηλαδή να τηρούνται για παράδειγμα αρχεία απαλωτριώσεων και εκτιμήσεων του ώστε να μην ε, μπορούν να λαμβάνουν χώρα απάτες και ούτω καθεξής. Να υπάρχουν μητρώα, λοιπόν για όλα αυτά. Να υπάρχει ε, για παράδειγμα ε, ε, τοπογράφηση όλων των ε, συνόρων των εν λόγω ακινήτων, οικοπαίδων και των υπολείπων τμήματων από, άλλες, από άλλα ακινήτα για να μην υπάρχουν προβλήματα και αργότερα με τις αποζημιώσεις. Και από εκεί και μετά, πολύ σημαντική σύσταση ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική φύση λύση σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δασικών περιοχών και των σχετικών χαρτών, γιατί αυτό αυτό το ζήτημα δημιουργεί καθυστερήσεις σε, όλες τις, σε όλο τον τύπο της επενδύσεις, της απαλωτριώσης, το κτηματολόγιο και ούτω καθεξής. Άλλη πρόταση ήταν να διοργανωθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, ώστε να ε, υπάρξει καλύτερη ενημέρωση και ε, βελτίωση της ειδικής κουλτούρας στην ίδια την, ε, στον κρατικό, στην κρατική διοίκηση. Επίσης προτάθηκε να υπάρχει καλύτερη εξέταση των δαπανών απαλωτρίωσης με πιο κριτικά κατά την ε, προπαρασκευή των σχετικών έργων. Είπατε δηλαδή ότι ε, συχνά ε, το κόστος της απαλωτρίωσης σε σύγκριση με το συνολικό κόστος του έργου ήταν πολύ συχνά υπερβολικά υψηλό. Ναι, αυτό μπορεί να ίσχυσε σε περιπτώσεις όπου ε, το έργο βρισκόταν σε ιδιαίτερα ανεπτυγμένες και ακριβές περιοχές. Όταν δηλαδή ε, κανείς ε, υλοποιεί ένα έργο σε μια τέτοια περιοχή, προφανώς είναι αναγκασμένος να καταβάλει τις σχετικές αξίες. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Αλλά υπάρχουν κάποια έργα τα οποία μπορούν να μετεγκατασταθούν, να λάβουν χώρα αλλού και να μην δηλαδή υλοποιηθούν στις πλέον ακριβές περιοχές. Αυτό είναι λοιπόν άλλη μια σημαντική πτυχή. Μια ακόμα σύσταση θα πρέπει επιτέλους να υιοθετήσουμε τις ε, διεθνείς ε, πρακτικές σε ό,τι αφορά τις ε, εκτιμήσεις, τις μεθόδους εκτιμήσεις και την, να βελτιώσουμε και την διαθεσιμότητα των δεδομένων σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή μια δίκαιη εκτίμηση αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα δεδομένα για την αγορά κινητών. και παρόλο θα υπάρξει μια διάσεψη το ε, Σεπτέμβριο από την πλευρά της Νομοσπονθίας ε, των ε, τοπογράφων ακριβώς για την ε, παρακολούθηση των ε, τιμών της αγοράς ακινήτων, πώς γίνεται δηλαδή η εκτίμηση και αφορά βέβαια ε, ε, όλες τις περιοχές του κόσμου και όχι μόνο την Ελλάδα και θα σας καλούσα να συμμετάσχετε εκεί. Ε, ε μία ακόμα σύσταση της διεθνούς κοινοτητα ήταν να δημιουργηθεί μία ανεξάρτητη και διεπαγγελματική επιτροπή εκτίμησης που θα, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και των δύο πλευρών, ώστε ακριβώς να διευκολυνθεί και η εφαρμογή φιλικών διακανονισμών. Ε, και ε, τα δικαστήρια σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει απλώς να εκκοινώνουν τις αποφάσεις που θα λαμβάνουν η σχετική επιτροπή. Δεν θα πρέπει δηλαδή να επισέρχεται το δικαστήριο στις λεπτομέρειες της εκτίμησης. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Μία ακόμα σύσταση είναι να ε, υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες, περισσότερος αριθμός δικαστών για τις απαλωτριώσεις και να εξεταστεί και η δημιουργία ενός ειδικού δικαστηρίου απαλωτριώσεων με εξειδικευμένο δικαστή. επίσης αναφέρθηκε και το ζήτημα βέβαια της προώθησης της ε, αρχής της, ε, του μηχανισμού της ανταλλαγής ε, μετά λοιπόν από την ολοκλήρωση τη μελέτη υπήρξαν μία σειρά από τροποποιήσει στον νόμο και αναφέρονται εδώ όλε οι επιμέρου τροποποιήσει και τα επιμέρου άρθρα του νόμου και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η εφαρμογή των τίτλων ε, ε, των, της μεταβίβασης των τίτλων ε, ιδιοκτησίων και όλα αυτά περνούν στο αρχικό τμήμα της διαδικασίας και ότι χρειάζεται και μια γνωμοδότηση από την πλευρά της υπηρεσίας, πράγμα το οποίο είναι εξίσου επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης σημειώνω ότι η δυνατότητα κατάληψης της της ε, γης ενδεχομένως να είναι ε, κάτι το θετικό γιατί με αυτόν τον τρόπο επιταχύνει τη διαδικασία από το δικαστήριο και ε, προβλέπεται και εδώ μία άμεση ε, ένας άμεσος καθορισμός ε, ε, της ημερομηνία της συνεδρίασης του δικαστηρίου και το γεγονός ότι δεν θα είναι δυνατόν να τροποποιηθούν, να τροποποιηθεί η σχετική προθεσμία και όλα αυτά είναι πολύ θετικά εφόσον όμως έχει καταβληθεί αποζημίωση των ιδιοκτητών πριν από οποιαδήποτε έξωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν αναφέρομαστε μόνο σε τοπικού ε, επενδυτέ ε, και πολιτέ. γιατί προφανώς ελπίζουμε να προσελκύσουμε και διεθνεί επενδύσεις. Κάτι ακόμα ε, που είναι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική τροποποίηση είναι ότι για τις περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο 7α, δηλαδή δεν είναι στρατηγικές επενδύσεις, προβλέπεται κάτι το θετικό, ότι δηλαδή υπάρχει μόνιμη έξωση η οποία ξεκινάει από, τον, ε, από την μερμένα του καθορισμού της ε, προσωρινής αποζημίωσης. Ε, και επίσης σημαντική αλλαγή είναι η υποχρεωτική εφαρμογή των προθεσμιών σε ό,τι αφορά την έκδοση απόφαση του δικαστηρίου για την αποζημίωση. Σημαντικές είναι και οι τροποποίησεις σε ό,τι αφορά την διαδικασία και, τη βελτίωση της διαδικασίας εκτίμησης της αξίας και η πρόβλεψη να, είναι υποχρεωτική μια έκθεση από την Επιτροπή Εκτίμησης και από ανεξάρτητο εκτιμητή για σχηματοδοτούμενα έργα. Και εδώ θα ήθελα να πω δεν αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικές είναι οι τροποποιήσεις που έγιναν σε ό,τι αφορά την ε, ευθύνη. Ε, εκείνο Πάντως το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι το άρθρο το οποίο αυξάνει το μέγιστο όριο σε ό,τι αφορά την ε, διοικητική επιδίκαση ε, σε ό,τι αφορά τον ε, διοκτήτη της περιουσίας η αύξηση από δηλαδή σε 10.000 ευρώ ήταν ένα θετικό βήμα αλλά πραγματικά θα πρέπει να είναι πιο μεγάλη αυτή η αύξηση. Ε, επίσης κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι είναι ότι στον προηγούμενο νόμο, το 4070, προβλεπόταν υποχρεωτικά να υπάρξει μία δημόσια ε, πρόσκληση ε, πριν από ε, την επίσημη κήρυξη ε, της ε, διαδικασίας της ε, απαλωτρίωσης για να είναι δυνατή η εφαρμογή στο μέλλον ενός μιας διαδικασίας φιλικού διακονισμού. Αυτό τώρα δεν προβλέπεται πλέον με τη βάση τη νέα τροποποίηση, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά ένα βήμα προς τα πίσω και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί έγινε τελικά αυτή η τροποποίηση. Ε, εντάξει. Δεν θέλω να σα ε, κουράσω εδώ. Ήταν κάποιε συστάσει εδώ σημαντικέ ε, σε συνέχεια τη μελέτη. Αυτά από την πλευρά μου σα ευχαριστώ που με ακούσατε και τι σκέψει μου για αυτό το ζήτημα. Πρόεδρο, ε, σα ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την πολύ κατανοητή και περιεκτική παρουσίαση σε ό,τι αφορά τα προβλήματα και της κατάληψης αλλά και της αγοράς γενικά ακινήτων στην Ελλάδα. πραγματικά θα πρέπει να μαθαίνουμε λίγο περισσότερο σε αυτή τη συζήτηση και θα ήταν ενδιαφέρον κάποια στιγμή να ακούσουμε και από εσά ε, ε, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον ε, στην Ελλάδα. Κυρία Απότσιου, προηγουμένω είπα κύριο Πότσιου, έκανα λάθο, λέω λίτρα, Σα ζητώ συγγνώμη για αυτό το λάθο. Να δώσω όμω τώρα τον λόγο στον κύριο Δελέο, ο οποίο εκπροσωπεί το Υπουργείο Ταφρών και Υποδομών της Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, για την πρόσκληση που απευθύνατε στο Υπουργείο μου και εύχομαι να βοηθήσουμε ως προς την, το, το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας με, τον, με τη διαδικασία της απαλωτρίωσης. Πράγματι όσα υπόθηκαν ε, είναι είναι ορθά, ε, έχουν καθυστερήσει έργα, τα, οι καθυστερήσεις έχουν οδηγήσει σε απώλεια πόρων ή τέλος πάντων στην καλύτερη περίπτωση μη αξιοποίησή τους. Ε, όπως θα έπρεπε και θα έπρεπε να συμβαίνει στη χώρα μας η οποία έχει ανάγκη, αυτή, είναι πολύτιμη αυτή όλη η πόρη από τα συγχρηματοδοτούμενα από τα προγράμματα της ΕΕ. Ε, ε, να σας το περισσότερο, ε, εργάζομαι στην Διεύθυνση Απολωτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, όπου διαχειρίζεται ένα πλήθος απαλωτριώσεων που ίσως αντιστοιχεί ίσως το 50% όλων των απολωτριώσεων που αφορούν στη δεδομένη χρονική περίοδο για έργα, για έργα υποδομής. Ε, ε, ετοίμασα μια, ύστερα από την προσκλησία σας, μια ε, παρουσίαση, η οποία απαριθμώ τη διαδικασία που, που της απαλωτρίωσης στα κέρια μια συνοπτική παρουσίαση. Ε, αντιλήφθηκα <laughs> πολύ έγκαιρα ότι ήδη η Επιτροπή σας και οι συνομιγυρίες έχουν μπει σε πολύ πιο ουσιαστικά θέματα και με με κορύφωση την μελέτη, τη συγκριτική μελέτη η οποία ε, έτυχε, ε, μου γνωστοποιήθηκε και είδα πράγματι ότι προσέγγισε το θέμα των απολωτριώσεων στην Ελλάδα με πάρα πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Λοιπόν, ε, ήθελα ωστόσο να τρέξουμε λίγο αυτή την παρουσίασή μου ε, ως προς τα βασικά της κεφάλαια. Πράγματι, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα προστατεύεται και όπως σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, λοιπόν, με έναν τρόπο επαρκή. Ε, έχει ένα σύνταγμα το οποίο ε, είναι, μάλιστα θα το έκρινα προσωπικά, ε, υπερπροστατεύει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, γιατί θέτει και προϋποθέσεις στην αφαίρεση της ιδιοκτησίας ε, ενώ αντίθετα όλα τα ευρωπαϊκά συντάγματα του, ε, της Ευρώπης δεν εξειδικεύουν και δεν, δεν περιορίζουν τον νομοθέτη σε, μια τέτοια, ε, σε τέτοια είδου ζητήματα. Δηλαδή, οι προϋποθέσεις που θέτει το Σύνταγμα το, ελληνικό είναι ότι θα πρέπει η αποζημίωση να καθορίζεται από τα δικαστήρια, λοιπόν, να καταβάλλεται η αποζημίωση πριν την, ε, ε, πριν κατάληψη της διοκτησίας και σε κάθε περίπτωση ε, η δημόσια ωφέλεια να, έχει να είναι νομοθετημένη. Λοιπόν, η, ένα ζήτημα που δημιουργείται σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά συντάγματα είναι η δικαστική απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό της αποζημίωσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση Ε, θα μπορούσε στην Ελλάδα, αν το επιτρέπουν οι, κοινωνικο, οι κοινωνικες συνθήκες και εν ώψη της ε, αναθεώρησης του συντάγματος να επαναξεταστεί το άρθρο για την προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας αν θα μπορούσε να, ε, να απαλληφθεί δηλαδή η υποχρεωτική δικαστική ε, δικαστικός καθορισμός της αποζημίωσης. φυσικά αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο για να, για να ξεφύγουμε και να, και να προχωρήσουμε σε διαδικασίες ε, φιλικού διακανονισμού για την απόκτηση των ακινήτων, όπως πολύ εύστοχα η κυρία Πότσιου ε, έχει παρατηρήσει και μελετήσει, ε, στις χώρες της, της Ευρώπης ε, ο φιλικός διακανονισμός υπερβαίνει το 80% των περιπτώσεων. Έτσι. Λοιπόν, ενώ στην Ελλάδα είναι κάτω από τη μιας ε, ποσοστιαίας μονάδας. Στην... Η ελληνική πολιτεία χρησιμοποιεί τακτικά μέσα για την αφαίρεση της ιδιοκτησίας για δημόσιους σκοπούς η οποία είναι η ελεύθερη εξαγορά, αυτή που λέμε ο φιλικός διακανονισμός, δηλαδή και που να συμπίπτει η βούληση και των δύο πλευρών, και δεύτερον η αναγκαστική απαλωτρίωση. Για όλες τις περιπτώσεις απόκτηση των αναγκαίων ακινήτων για δημοσίους σκοπούς είναι το μέσο που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά όπως είπαμε είναι η αναγκαστική απαλωτρίωση. Υπάρχουν, ε, διαθέτει και κάποια εργαλεία έκτακτης ανάγκης όπως είναι η επίταξη, η οποία χρησιμοποιείται κατά, σε περιόδους ε, ε, άμεσης δημόσιας ανάγκης, όπως είναι οι στρατιωτικές ανάγκες η, και η προστασία, και ο, η προστασία από κινδύνους της δημόσιας τάξης και δημόσιας υγείας. Το 1992 και πάλι με το ίδιο, ε, το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Ελλάδα και μάλιστα οξύτερο, ε, θεσμοθετήθηκε για τα δημόσια έργα η επίταξη να επεκταθεί και στις περιπτώσεις της, ε, ε των συγχρηματοδοτημένων έργων ό, για να μην απολεστούν ανθρωπ, ε, συγχρηματοδοτημένοι πόροι. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή πολλά έργα στην Ελλάδα και στο δεύτερο και του τρίτου και με λιγότερα φυσικά στο τέταρτο ε, πλαίσιο στήριξης τα έργα προχώρησαν με τη διαδικασία της επίταξης, η οποία είναι διαφορετική από το 7α. Λοιπόν, η επίταξη φυσικά ε, κατηγορείται στη χώρα μας, κυρίως από τη νομική επιστήμη, από τη νομική θεωρία, ότι είναι ένα μέτρο ε, που κινείται στα όρια της συνταγματικής ανοχής. Ωστόσο όμως ένα μεγάλο μέρος των έργων ε, προχώρησαν με αυτή τη διαδικασία και ιδίως και αυτά τα Ολυμπιακά έργα που την ε, περίοδο προετοιμασίας της χώρας ε, έγιναν με επιτάξεις. Ε, πράγματι, σήμερα η ελληνική η πολιτεία βγάζει από την ατζέτα της την επίταξη και πολύ σωστά κάνει γιατί πλέον δεν, δεν έχει ερίσματα να κάνει να χρησιμοποιεί ένα έκτακτο μέτρο για τόσο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αντικατέστησε αυτό το μέτρο με, την, με τη διαδικασία την αποκαλούμενη του 7α, δηλαδή μια προσωρινή κατάληψη, παρέχοντας ένα τμήμα της εύλογης αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη. Εδώ πράγματι παρατηρούμε ότι κερδίζουμε σε χρόνο και μειώνει τη διαδικασία από 22 μήνες που ένας καλός διαχειριστής της απαλωτρίωσης μπορεί να την προσδιορίσει, δηλαδή να συντελέσει, να συντελέσει απολωτρίωση σε 22 μήνες από τη σύνταξη των κτηματογραφήσεων και μπορεί να περιορίσει αυτή την περίοδο των 22 μηνών που είναι ο κανονικός χρόνος ε, σε 15. Επομένως έχουμε μια, το 7α επιφέρει σε ό,τι αφορά την χρονική, το χρονικό κέρδος κατά 7 μήνες. Ήδη αυτό το πείραμα έγινε, επιτεύχθηκε με, με την προώθηση απολωτριώσεων ειδικά των έργων παραχώρησης ε, στο τρέχον εξάμεινο του έτους 2016 με αποτελέσματα δηλαδή να μπορέσουμε να περιορίσουμε την κατάληψη, την προσωρινή κατάληψη, να επιτύχουμε προσωρινή κατάληψη στους 15 μήνες. Λοιπόν, φυσικά ε, όλα αυτά τα έκτακτα μέτρα έχουν και κάποιες δυσάρεστες ε, επιπτώσεις σε, στην άλλη πλευρά στους πολίτες, στους στιγόμενους ιδιοκτήτες. Όπως πολύ καλά εντόπισε η κυρία Μπότσιου, ε, καταθέτει το δημόσιο το εύλογο τμήμα της αποζημίωσης, προκειμένου να, κάνει, να προβεί στην προσωρινή κατάληψη. Ωστόσο όμως δεν μπορούν οι δικαιούχοι να τα πάρουν στο συγκεκριμένο χρόνο σε πραγματικό χρόνο της κατάληψης. Γιατί θα πρέπει να υποχρεωθούν σε μια διαδικασία αναγνωρισή τους ως δικαιούχων μέσα από πάλι από δικαστήριο και ύστερα από αίτησή τους. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία τους παίρνει 6 ως 8 και πολλές φορές και ένα χρόνο ενώ τα λεφτά από τον φορέα, από τον υπόχρεο της αποζημίωσης έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων Ωστόσο όμως οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα ε, εισπράξουν αν δεν αναγνωριστούν δικαστικά. Λοιπόν, ε, στην... Τα μεγάλα προβλήματα που, που εγώ πιστεύω μάλλον ποιοι τρόποι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε δηλαδή τα προβλήματα της, ε, της απαλωτρίωσης ε, τα οποία κινούνται σε δύο άξονες. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το χρόνο και δεύτερον, σε ό,τι αφορά το κόστος. Ο χρόνος, αν πιστεύω ότι αν με, τα, με τις ειδικέ εξαιρετικές διαδικασίες ε, ε, υπάρξει και σταθεροποιηθεί στους 15 μήνες, ε, νομίζω ότι είναι, μια, ένα, είναι ένα καλό ε, ένα, ένας καλός χρόνος για την, και μπορεί να τύχει προγραμματισμού δηλαδή και να μην δυσχεράνει την εξέλιξη του έργου. Το κόστος ε, είναι μια παράμετρος η οποία ε, με μεγαλύτερη δυσκολία μπορεί να, να ελεγχθεί. Πρώτον, γιατί όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, έχουμε ε, έλλειψη ενός χωροταξιακού, χωροταξικού σχεδιασμού για να μπορούμε να προσεγγίσουμε τις αξίες των ακινήτων εκτός αστικού χώρου για να μπορέσουμε δηλαδή να, προσδιορίσουμε την, αξία της, της γης. Ε, φυσικά η έλλειψη του, εθνικού κτηματολογίου επηρεάζει και προς αυτή την κατεύθυνση και το σπουδαιότερο είναι ότι ε, δεν υπάρχει, λειτουργεί το, η φορολογική διοίκηση με το περίφημο σύστημα αντικειμενικών, προ, ε, αξιών, ε, οι οποίες είναι φορολογικές διοικητικές τιμές, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί μια γενικότερη σύγχυση και στα δικαστήρια και στους θυγόμενους πολίτες και σε κάθε περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν δεν αντιπροσωπεύουν τις αξίες γης. Ε, ε, μετά την ε, εισαγωγή του, του, μετά την θεσμοθέτηση δηλαδή των, της, έχω ξεφύγει στην εντάξει. <laughs> Συγγνώμη. Ε, η, μια προς τη σωστή κατεύθυνση κινήθηκε η διαδικασία να οι, οι εκτιμήσεις των απολυτρωμένων ακινήτων να διενεργούνται από πιστοποιημένους εκτιμητές ε, ενώ μέχρι, μέχρι πρότινος ήταν να γίνονται από κρατικούς υπαλλήλους με τη συμμετοχή φυσικά και κάποιου εμπειρογνώμονα ιδιώτη αλλά με, χωρίς ε, επιστημονικά και πρότυπα αποτίμησης ε, των αξιών. Ε, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο δικαστής, ο οποίος λάμβανε σαν πρόταση από το δημόσιο να καθοριστεί τιμή σε αντικειμενικές τιμές ή σε μη αιτιολογημένες εκτιμήσεις των κρατικών επιτροπών ε, ε, απλά απαξίωνε αυτές, δεν τις αξιολογούσε καν και προχωρούσε ε, με δικά του κριτήρια να μπορέσει να προσδιορίσει την αξία, την αξία των ακινήτων και πολλές φορές το δημόσιο συμφέρον ζημιωνόταν γιατί δεχόταν τα πιο τεκμηριωμένα ή κατ' επίφαση, επίφαση τεκμηριωμένα στοιχεία της άλλης πλευράς των ιδιοκτών. Λοιπόν, σήμερα ε, υπάρχει ένα, πιστεύω, ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να, να απασχολήσει την, ε, την ελληνική διοίκηση. Ε, είναι ότι ε, η βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των υπηρεσιών που, που ασχολούνται με τις απαλωτριώσεις. Σημειωτέων δεν είναι ότι με τις απολωτριώσεις ο κάθε φορέας γίνεται, που υλοποιεί έργα γίνεται διαχειριστής και αν υποθέσουμε ότι είναι πάνω από 500 φορείς στην Ελλάδα οι οποίοι διενεργούν, διαχειρίζονται απολωτριώσεις. Ε, είναι εύκολο να, κάνουμε σε κάποια, να γίνει σε κάποια υπουργεία, να γίνουν οργανωμένες δομές με, με μια βελτιωμένη διαχειριστική ικανότητα των υπηρεσιών, κυρίως στα Υπουργεία, αλλά είναι πολύ δυσκολότερο αυτό να επιτευχθεί σε επίπεδο περιφερειακό και ιδίως στους Δήμους και κοινότητες που έχουν μια ποιοτική, ε, μια ποσοτική και ποιοτική υποστελέχωση. Ε, ε, εγώ δίνω μεγάλη σημασία από την εμπειρία μου στην διαχειριστική ικανότητα για να μπορέσει να ελέγξει και το χρόνο και το κόστος ε, γιατί από ό,τι γίνεται εύκολα αντιληπτό η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Δηλαδή έχουν εξαντληθεί όλα τα, μέσα, έχουν σμικρινθεί όλες οι δικονομικές προθεσμίες με, σε σημείο που να έχουμε φτάσει να μην παρέχεται μια δίκαιη δίκη στους ε, θυγόμενους ιδιοκτήτες. Δηλαδή αρχίζουμε να προσκρούμε πλέον και να προσβάλλουμε ως ένα σημείο το πυρήνα του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Γι' αυτό κατά την άποψή μου θα ήταν ενδιαφέρον να βελτιωθεί και υπάρχουν πολλά περιθώρια προς αυτήν την κατεύθυνση η διαχειριστική ικανότητα των υπηρεσιών και των φορέων που διαχειρίζονται τις απολωτριώσει, ούτως ώστε ε, να υπάρξει και χρονική βελτίωση και φυσικά ε, ε, βελτίωση ο εξορθολογισμός του κόστους. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε, ε, σε μια διαρκή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, οι, οποία, ε, οι οποίες έχουν την ευθύνη ε, ελέγχου και αρμοδιότητα για το θεσμικό πλαίσιο των απολωτριώσεων να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ούτως ώστε να, να, πάμε να επεξεργαστούμε μια εκ νέου και εκ βάθρων ανα, αναδιάρθρωση, δηλαδή ανασχηματισμό του δικαίου της απαλωτρίωσης. Ούτως ώστε να, να μέσα από αυτό να, να υπάρξει και μια διαχειριστική παρέμβαση, μια κανονιστική παρέμβαση και να υποχρεωθούν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες οι οποίες ε, ε, μπαίνουν στη διαχείριση, συμμετέχουν στη διαχείριση της απολυτρίωσης, ούτως ώστε να υπάρχει ένας διοργανικός προγραμματισμός πλέον, ε, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθείται σε κάθε περίπτωση και να επιβάλλεται μέσω του, του νόμου με, με υποχρεωτικά πεδία. Αυτές είναι σε γενικέ γραμμές ε, ε, οι απόψεις μας και καταβάλουμε καθημερινά σε επίπεδο πραγματικό ε, να βελτιώσουμε και να μπορέσουμε να, να βοηθήσουμε δηλαδή τα έργα να σταματήσουν τουλάχιστον από την αιτία αυτή των απολυτριώσεων να επιφέρουν πρόσθετες καθυστερήσεις με συνεχή προβλήματα στη διαχείριση των, των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης. Ε, σας ευχαριστώ για την σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία. Γνωρίζετε ε, πόσα έργα συγχρηματοδοτούμενα ιδιαίτερη ε, σημασία ε, βρίσκονται ακριβώ σε καθυστέρηση λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν, λόγω των απαλωτριώσεων. Έχετε κάποιον αριθμό κατά νου, γνωρίζετε κάτι. αριθμός έργων ε, το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων διαχειρίζεται ένα, ένα, μέρος των, ε, των προγραμμάτων ε, και μάλιστα στις μεταφορές. Λοιπόν, θεωρώ όμως ότι υπάρχει μια καθυστέρηση σε 50% τα έργα που έχουν καθυστερήσει, δηλαδή άλλοτε μικρότερη καθυστέρηση, άλλοτε μεγαλύτερη, άλλοτε επικίνδυνη, άλλοτε που να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Είναι διαφόρων ειδών οι καθυστερήσεις που έχουν επισυμβεί στο πρόγραμμα λόγω των απολωτριώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη διευκρίνηση. Έχουμε ένα ακόμα ομιλητή, τον κύριο Ψαθά, ε, ο οποίο ε, βλαμβάνει των διαρθρωτικών ε, δομίων από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομίας και ανάπτυξη τη. Λέω Να πούμε ότι έχουμε, είχαμε προσκαλέσει και το Υπουργείο Οικονομικών. Στην αρχή μα είπαμε ότι θα υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο, τελικά δεν υπήρξε εκπρόσωπο, αλλά έχουμε λάβει ένα έγγραφο. Ο λόγο όμω στον κύριο Ψαθά, παρακαλώ. Ε, Καλησπέρα σε όλους, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση του σεμιναρίου αυτού και για την πρόσκλησή σας που μου δίνει τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω το θεσμικό πλαίσιο των παλωτριώσεων στην Ελλάδα, ιδίως όσον αφορά τις αποζημιώσεις για τους θυγόμενους ιδιοκτήτες και θα ήθελα να παρουσιάσω και ιδιαίτερα την περίπτωση που έχει να κάνει με την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα. Καταρχάς όμως, θα ήθελα να σας πω ότι εργάζομαι ως σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα για τα Διαρθρωτικά Ταμεία στα πλαίσια του Υπουργείου Οικονομικών στην Ελλάδα. Ασχολούμαι με την τοπογραφία, με μηχανικός και ανήκω στο σώμα πιστοποιημένων εκτιμητών και είμαι ειδικευμένο ε, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αποτίμηση της ε, αξίας ε, κτημάτων υγιής και ως το 2013 εργαζόμουν ως εμπειρογνώμων σε ζητήματα απολωτριώσεων, ιδίω όσον αφορά την κατασκευή των νέων αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα και το 2014 και το 2015 εργαζόμουν στα πλαίσια του Αγωγούα ΤΑΠΑ που ανήκει στον λεγόμενο νότιο διάδρομο μεταφοράς ε, φυσικού αερίου και που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα, τα οποία βέβαια οδηγούν και σε περιπτώσεις απαλωτριώσεων. Ας δώσουμε κάποιους ορισμούς. Η αναγκαστική απαλωτρίωση οδηγεί σε υποχρεωτική στέρηση της διοκτησίας για λόγους δημόσιας ωφελίας. Οδηγεί λοιπόν στη στέρηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί παρά μόνο αν συντρέχουν λόγοι δημόσια ωφελία. Λέγεται στο ελληνικό σύνταγμα ότι κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο όταν και όπως ο νόμος ορίζει και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση. Κατά τον ίδιο τρόπο, το πρώτο πρωτόκολλο της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών λέει τα ακόλουθα. Ουδή στερείται τα υπάρχοντά του παρά μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με τις προποθέσεις προβλέπονται από την αρμόδια νομοθεσία και από τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αυτές συμβάσεις όσον αφορά την αποζημίωση, πλήρης αποζημίωση πρέπει να υποβάλλεται και αυτή συνιστά αποκατάσταση της ζημίας και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι πλήρης. Η πλήρης αποζημίωση αντιστοιχεί στην πραγματική αξία του παλαιτρωταίου ακινήτου και όχι τόσο στην υποκειμενική αξία. Πραγματική αξία αντιστοιχεί τελικά στην αξία αντικατάστασης ή άλλο στην αγοραία αξία. Η πλήρης αποζημίωση δεν περιορίζεται μόνο στην εκτιμόμενη και προσδιοριθήσα αξία του απολυτριωτέου ακινήτου, αλλά περιλαμβάνει και οποιαδήποτε άλλη αποκατάσταση ζημίας που έχει προκύψει από την απαλωτρίωση. Έχουμε εδώ πέρα, στα πλαίσια της αποζημίωσης, την αξία του ακινήτου και αποζημίωση οποιοδήποτε κτισμάτων, απόσβεση των απομείναντος τμήματος ιδιοκτησίας, δαπάνες μετεγκατάστασης και δικαστικά έξοδα. Όλα αυτά πρέπει να καλύπτονται από την αποζημίωση. Στο σημείο αυτό πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποια επιμέρους ε, σημεία αυτού του οποίου ονομάζομαι πλήρης αποζημίωση. που πολλές φορές επηρεάζει ακόμα και το ποσό εκείνο το οποίο επιστρέφεται στον ε, δικαιούχο μέσω της φορολογικής του δήλωσης ή πολλές φορές έχει να κάνει με άλλες μορφές πλήρους αποζημίωσης. Όπως σας είπα, ακολουθούμε την αγοραία αξία ...και την οποία προβλέπεται συγκεκριμένος ορισμός όσον αφορά την συμφωνία της Βασιλείας. Αγορέ αξία το εκτιμόμενο ποσό, έναν του οποίου θα ανταλλασσόταν το ακίνητο κατά την ημέρα της αποτίμησης, μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πολιτή που εκφράζουν ελεύθερα τη δικαιοπρακτική τους βούληση, συναλλάσσονται από υποκανονικές συνθήκες συνταγωνισμού μετά από κατάλληλη εμπορική διαπραγμάτευση και ενεργούν καθένας εν πλήρη γνώση, με σύνεση και χωρίς καταναγκασμό. Βασιζόμαστε λοιπόν στην καλύτερη δυνατή χρήση του ακινήτου, κατά αυτόν τον τρόπο αποτιμάται η αξία, και πρέπει να καταλήγουμε στην υψηλότερη δυνατή αξία. Η διαδικασία αποτίμησης τώρα της αξίας στα πλαίσια της απαλωτρίωσης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία εφαρμόζεται από δύο φορεί. Από την Επιτροπή προβλέπεται στη νομοθεσία 2882 του 2001, όπου έχουμε δύο αξιωματούχου του Υπουργείου Οικονομικών και ένα εξωτερικό εμπειρογνώμονα. Και δεύτερον, έχουμε μέλη από το Μητρό Πιστοποιημένων Εκτιμητών που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Το επάγγελμα του οπισθοποιημένου εκτιμητή, του ορκωτού μάλλον εκτιμητή, απελευθερώθηκε το 2013. Μέχρι το 2013 μόνο το σώμα ορκωτών εκτιμητών μπορούσε να αποφανθεί για την αποτίμηση της αξίας ακινήτου, ήταν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Πρόκειται για ένα σώμα αρκωτών λοιπόν εκτιμητών που συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Ενώσεων Εκτιμητών και ακολουθούσαν συγκεκριμένα πρότυπα αποτίμησης ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με την νομοθεσία λοιπόν αυτή, τόσο η κυβέρνηση όσο και άλλοι δημόσιοι φορείς έπρεπε να ακολουθούν τη συμβουλή του σώματος ορκωτών εκτιμητών και προβλέπουν για αυτού συγκεκριμένες αμοιβέ από το Υπουργείο Οικονομικών. Το σώμα αυτό λοιπόν ορκωτών εκτιμητών διέκοψε την παροχή υπηρεσιών του το 2013. Με την κατάργηση λοιπόν του σώματος ορκωτών εκτιμητών, δημιουργήθηκε ένα μητρό πιστοποιημένων εκτιμητών με νομοθεσία 4152 του 2013. Εδώ πέρα τα μέλη πιστοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς που ακολουθούν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αποτίμησης. Οι φορείς αυτοί είναι η Τεγκόβα, το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Εκτιμητών, καθώς επίσης και το Star Register. Επίσης προβλέφθηκαν κατάργηση των καθορισμένων αμοιβών των εκτιμητικών υπηρεσιών, δημιουργήθηκε ένα πειθαρχικό συμβούλιο και αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών, λίγο πιο αργά αν μπορείτε, στα πλαίσια λοιπόν του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών, επί του παρόντος έχουμε 412 φυσικά πρόσωπα και 41 νομικά πρόσωπα. Με μια σειρά τώρα νομοθετικών μέτρων, η χρήση αυτού του Μητρώου Πιστοποιητικών Εκτιμητών γίνεται πλέον και σε άλλες περιπτώσεις, σε περιπτώσεις παραχωρήσεων νέων αυτοκινητοδρόμων, σε έργα μεγάλου οικονομικού συμφέροντος, αλλά και σε έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα δερθωτικά ταμεία και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο Φιλέτης, ο επιβαρημένος λοιπόν με την καταβολή της, πλήρης και της πλήρους θα πρέπει να ακολουθεί την έκθεση που υποβάλλεται από τον ανεξάρτητο αυτό φορέα εκτίμησης. Πέρα λοιπόν από τον ορισμό αυτό για τις απαλωτριώσεις και για την αποζημίωση, θα ήθελα να αφαιρθώ τώρα πιο συγκεκριμένα στα έργα νέων αυτοκινητόδρομων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, γιατί εδώ μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν από τη μία προβλήματα και καθυστερήσεις, από την άλλη όμως έχουμε και την έγκριση κάποιων νέων θετικών διαδικασιών για τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Όπως βλέπετε στον πίνακα αυτό, από το 2007 και μετά προβλέπονται και έχουν υπογραφεί πέντε νέα έργα αυτοκινητοδρόμων, περίπου 1.300 ε, χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων πρόκειται να κατασκευαστούν και έχουμε περίπου 80.000 στιγόμενους ιδιοκτήτες εξαιτία των έργων αυτών. Με τους νέους λοιπόν αυτούς αυτοκινητοδρόμους πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε σε κάποια νέα σημεία που έχουν να κάνουν με την αγορά γης, την απόκτηση γης και την παράδοση της γης. Ο σχεδιασμό των απολυτριώσεων πολλέ φορέ οδήγησε σε καθυστερήσει και 9 χρόνια μετά την υπογραφή τη σύμβαση παραχώρηση, οι περισσότεροι αυτοκινητόδρομοι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Όσον αφορά τι συμβάσει παραχώρηση, η αρχική πρόβληψη για την παράδοση της γη προς τον ανάδοχο ήταν 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης παραχώρησης. Η απόκτηση και η παράδοση της γης όμως είναι 22 μήνες όταν ακολουθεί τη συνήθις διαδικασία. Συνεπώς, είναι προφανές ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος της πιο σύντομης διαδικασίας που οδήγησε βέβαια σε πάρα πολλές καθυστερήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε αδυναμία απορρόφησης πιστώσεων, στο ότι δεν δημιουργήθηκαν θέσεις απασχόλησης, το ότι περιπλάκησαν πάρα πολλέ φορέ τα έργα και πολλέ φορέ δεν συνέβαλαν στην αύξηση οδική ασφάλεια, αλλά περισσότερο στην αύξηση των ατυχημάτων. Επίση, υπήρξε μια καθυστέρηση όσον αφορά την καταβολή τη αποζημίωση στου δικαιούχου και πολλέ φορέ ακόμα και οι ίδιοι οι ανάδοχοι ζητούσαν υψηλέ αποζημιώσει εξαιτία των καθυστερήσεων στην εκτέλεση του έργου από το ελληνικό κράτος. Από την άλλη τώρα, και στον αντίποδα της ανεπαρκούς αυτής σχεδίασης των απαλωτριώσεων, όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τη δικασία της αποζημίωσης, Είχαμε θετικές τροποποιήσεις που οδήγησαν στην εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με την κοινοτική και παγκόσμια νομοθεσία. Σύμφωνα με την νομοθεσία 3555 του 2007, το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ήταν πλέον υπεύθυνο για την εκτίμηση της αποζημίωσης που έπρεπε να δοθεί σε σχέση με τι απαλωτριώσει που προέκυψαν εξαιτία των έργων αυτών αυτοκινητοδρόμων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι εκτιμήσει για τι αποζημιώσει για πρώτη φορά βασίζονταν σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αποτίμηση, τα οποία ακολουθεί ο φορέα Τεγκόβα. Για πρώτη φορά επίσης είχαμε κεντρικό σχεδιασμό για τα περισσότερα αυτά έργα. Επίσης είχαμε τη δημιουργία μιας ενοποιημένης βάσης δεδομένων όσον αφορά την γη που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, τα υπόλοιπα κτίσματα που βρισκόταν στη γη αυτή και επίση είχαμε πολύ σημαντική μείωση του ποσοστού υψηλή αποζημίωση που συνήθω ζητούν τα δικαστήρια. Ένα 70% των δικαστικών αποφάσεων τελικά συμμορφωνόταν με την αρχική εκτίμηση που είχαν κάνει εκτιμητέ. Από το 2013 και μετά και με την κατάργηση του σώματος ορκωτών εκτιμητών, το μητρό πιστοποιημένων εκτιμητών ήταν υπεύθυνο για την εκτίμηση της αποζημίωσης που έπρεπε να κατατεθεί, να υποβληθεί. Όσον αφορά τους νέους αυτούς αυτοκινητοδρόμους, μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο είχαν προκύψει κάποιες καθυστερήσεις. Είχαμε ανεπαρκή σχεδιασμό της διαδικασία Πολλές φορές ε, η προβλεπόμενη περίοδος των 12 μηνών που δεν μπορούσε να τηρηθεί αποτελούσε πρόβλημα του αρχικού σχεδιασμού. Επίσης γινόντουσαν πάρα πολλές τροποποιήσεις στα αρχικά σχέδια γιατί δεν είχαν σχεδιαστεί εξ αρχής πολύ καλά τα σχέδια αυτά κατασκευής αυτοκινητοδρομών και επίσης είχαμε καθυστερήσεις διότι δεν υπήρξε ενεργοποίηση τελικά του άρθρου 7α που προβλέπεται στην νομοθεσία για τα Ολυμπιακά έργα και προβλέπει επιταχυμένη διαδικασία. Πέρα από τι καθυστερήσει όμω, είχαμε και βελτιώσει του νομικού πλαισίου όσον αφορά την καταβολή τη αποζημίωση. Πιο συγκεκριμένα, άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτερα το σύστημα διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων όσον αφορά την αποτίμηση της αποζημίωσης για όλα αυτά τα νέα έργα αυτοκινητοδρόμων, αλλά και για τις χρηματοδοτούμενα έργα. Επίσης είχαμε και μια νέα νομοθεσία που προβλέπει ειδική δικαιολόγηση από τον δικαστή σε περίπτωση μεγάλης απόκλησης της απόφασής του από την εκτίμηση την αρχική που έχουν κάνει οι εκτιμητές όσον αφορά την αξία του ακινήτου. Τέλος, ότι οι αρχές αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στη δικασία της απαλωτρίωσης, θα μπορούσαν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις. Για παράδειγμα, καλύτερο σχεδιασμός των απολωτριώσεων. Θα πρέπει να ληφθεί νομοθετική δράση προκειμένου να δημιουργηθούν μη δικαστικέ, εθελούσιε δηλαδή διαδικασίε για την απόκτηση γη, θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερο συντονισμό όλων των μπλεκόμενων υπηρεσιών και θα μπορούσαν να, δημιουργηθούν, να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, γεωχωρικών δεδομένων συγκεκριμένα, προκειμένου να υπάρχει καλύτερος υπολογισμός και της αξίας της γης αλλά και της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί. Θα ήθελα επίσης να πω ότι πριν από δύο μήνες η ελληνική κυβέρνηση θεώρησε ότι ένας μεγάλος αριθμός έργων θα πρέπει να αποτελέσουν έργα ιδιαίτερη προτεραιότητα, μεγάλου οικονομικού εθνικού συμφέροντο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλο και περισσότερα έργα τελικά υπάγονται στην νέα νομοθεσία η οποία είχε προβλεφθεί για τα Ολυμπιακά έργα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τουλάχιστον για ένα μεγάλο αριθμό έργων θα αποφευχτούν οι καθυστερήσει του παρελθόντο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα έργα για τα οποία εσεί είστε αρμόδιος στο δικό τομέα, τα οποία πλήττονται από αυτήν την ε, κατάσταση. Γνωρίζετε. the that uh, still have some problems, but we Τα έργα τα οποία θεωρούμε ότι παρουσιάζουν κάποια προβλήματα, αλλά τα οποία θα επιληθούν με την νομοθεσία αυτή για τα Ολυμπιακά έργα, είναι τα πέντε αυτά έργα για τους αυτοκινητοδρόμους που έχουν τεράστιο προπολογισμό, 4 δισεκατομμύρια περίπου, Ενεργοποιήθηκε λοιπόν αυτή η επιταχυμένη διαδικασία προβλέπεται στην νομοθεσία για τα Ολυμπιακά έργα και περιμένουμε ότι τους επόμενους μήνες όλα αυτά τα προβλήματα θα έχουν επιληθεί. Δεν ξέρω ποιος αν το γνωρίζετε, αλλά προβλέπεται μία υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων να ολοκληρωθούν τα πέντε αυτά έργα μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2017. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε 10 μήνε μόνο μπροστά μα. Διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα χρειαστεί να επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία έχει λάβει για την κατασκευή αυτών των έργων. Ναι, ναι, νομίζω πως ε, έως την 1η Μαρτίου του 2017 θα τα θα προλάβετε, νομίζετε, θα, θα τα καταφέρετε. Will you, will you manage to, will you manage to do it? Yeah, we are sure about that. Ναι, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Πρόεδρο, χαίρομαι που τα ακούω. Σας ευχαριστώ ε, όλους αυτές τις πολύ εντυπωσιακέ ε, παρουσιάσεις. Εγώ, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, έμαθα πολλά σήμερα. Αλλά βέβαια το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε από εδώ ε, και μετά. Έχουμε του ε, τρει εμπειρογνώμονε εδώ από την Ελλάδα και του ρωτάω τι μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε την κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί θέλουμε προφανώ να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα. Ε, και με τα έργα τα οποία είδαμε κι εμείς, ε, ε, διαπιστώσαμε ότι πραγματικά κατά κάποιο τρόπο είναι αξιοζήλευτη η Ελλάδα γιατί λαμβάνουν χώρα τόσα πολλά έργα υποδομής αυτή την περίοδο και είναι πλημμυρά τα όσα ακούσαμε σήμερα εδώ οπότε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις καθυστερήσεις οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω εδώ από τα αριστερά τους προηγούμενους αυτή δηλαδή η απαραίτητη τροπή του συντάγματος η οποία έχει αναφερθεί επανειλημμένα. γνωρίζω ότι πάντοτε υπάρχουν κάποια συμφέροντα εκεί ε, τα οποία εμπλέκονται σε τέτοιε διαδικασίε. Άκουσα και την άποψη από την πλευρά κάποιων δικηγόρων. Οπότε σα ρωτάω, είναι πραγματικά απαραίτητη μια τέτοια. Αλλά γιατί ο, ο ένα μόνο από του τρει εμπειρογνώμου αναφέρθηκε σε αυτό. Οπότε ρωτάω πόσο απαραίτητη είναι μια τέτοια αλλαγή. Και μπορούμε να αναμένουμε ρεαλιστικά ότι θα λάβει χώρα, δηλαδή θα υπάρξει μια τροποποίηση τέτοια συνταγματική. Και από εκεί και μετά, δεύτερο ερώτημα, πώς μπορούμε εμείς από την πλευρά να σας βοηθήσουμε. Ε, αυτό λοιπόν να, να, να ξεκινήσω να, να απαντήσουμε τη σειρά τη συμπληρωμόνων και ενδεχομένω ε, ε, θα θέσω και κάποια ερωτήματα στην Επιτροπή και βέβαια και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ, τα μέλη του Κοινοβουλίου τη Επιτροπή, αν θέλουν να θέσουν ερωτήματα, θα έχουν και αυτή τη δυνατότητα. Ε, καταρχάς, νομίζω ότι δεν υπήρχε κάποια συνταγματική αλλαγή που να επηρεάζει το καθεστώς της προστασίας ε, των περιουσιακών ε, δικαιωμάτων. Δεν ξέρω αν εννοείται για το Ολυμπιακό άρθρο το οποίο ε, μιλήσαμε εκτενώς ότι έχει ενεργοποιηθεί. Ε, σας ρωτώ για να είναι ξεκάθαρη και η, απαντήσή μου, επειδή ε, συνταγματική αλλαγή που να έχει να κάνει με, ε, με την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων στη χώρα ε, δεν, δεν προβλέπεται. Ε, έκανα πράγματι μια αναφορά σε ό,τι αφορά το ελληνικό σύνταγμα το οποίο έχει μια δέσμευση ότι απαραίτητα θα πρέπει να η αποζημίωση να καθορίζεται από τα δικαστήρια. Ε, και αυτό αφορά φυσικά μια προσωπική μου άποψη κατά πόσο θα μπορούσε και φυσικά είναι μια, αυτό είναι σοβαρή πολιτική απόφαση δηλαδή του, πολιτικού συστήματος για να δει αν πράγματι ε, θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτή η διάταξη του συντάγματος ούτως ώστε να εξαιρέσει την δικαστική συμμετοχή στον καθορισμό της αποζημίωσης. Είναι ευνόητο ότι εφόσον δεν συμφωνήσουν τα μέρη, τα δικαστήρια πάλι θα αποφασίζουν την αποζημίωση, αλλά να μην θεωρείται σαν προαπαιτούμενο για την συντέλεση της απαλουτρίωσης, για την κατάληψη της ιδιοκτησίας. Αυτό έχει το νόημα, δεν έχει ανοίξει στην, ε, στην χώρα μας τέτοιο ζήτημα, αλλά ε, ήταν καθαρά προσωπική μου άποψη κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Λοιπόν, ε, γιατί μην ε, θέλω να σημειώσω ότι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, επομένως είναι θέμα ε, πολιτικών συνθήκων και κοινωνικών. Αυτό ως προς το ζήτημα. Το κύριο, κύριο θέμα που πολύ σωστά κυρία Πρόεδρε θέσατε, τι μπορούμε να κάνουμε πλέον από εδώ και πέρα ούτω ώστε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες. Ε, ε εμείς, ε, ε, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την, τα διαχειριστικές μας αριθμίες όπου υπάρχουν και σε ένα συνολικό επίπεδο. Δηλαδή θα πρέπει τα προγράμματα, τα φορείς υλοποίησης είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο κάποια υπουργεία ή κάποιες υπηρεσίες, κάποιοι φορείς νομικά πρόσωπα τα οποία διαχειρίζονται ε, μεγάλα έργα. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια ολιστική ε, βελτίωση της διαχείρισης όλων των φορέων που υλοποιούν έργα συγχρηματοδοτούμενα. Τότε θα φανεί μια σοβαρή ε, βελτίωση της, της κατάστασης. Επομένως, εκείνο που εντοπίζω εγώ στο διαχειριστικό μέρος, που υπάρχουν πολλοί τεχνικοί τρόποι να βοηθήσει και η η Επιτροπή σας προς αυτή την κατεύθυνση και μπορεί να μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε στο μέλλον πιο ε, τεχνικά θέματα, πώς μπορεί αυτή η βελτίωση να επέλθει. σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, αναφέρθηκα εκεί στον κατάλογο των συστάσεων που προέκυψαν από τη μελέτη και ε, δεν μπορώ να θέσω αυτέ τι συστάσει σε προτεραιότητα, γιατί όλε του είναι σημαντικέ. Δηλαδή και η ευαισθητοποίηση του ευρωστηνού είναι ε, σημαντική και η αύξηση τη εμπιστοσύνη των πολιτών στο ε, κράτο. Και νομίζω πω ακριβώ με την ασφάλεια του δικαιώματο ιδιοκτησία μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό. Και αυτό βέβαια αφορά μόνο, όχι μόνο επενδύσεις για παράδειγμα σε ακίνητα, αλλά και για παράδειγμα στον τραπεζικό τομέα επενδύσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή εδώ να παίζουμε με αυτό το ζήτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα. Ε, σε ό,τι αφορά ε, την δικαστική διαδικασία που προβλέπει το ελληνικό σύστημα, ναι, ε, θα πρέπει να ε, κυρώσει το δικαστήριο μια εκτίμηση. Αλλά αν αυτή η εκτίμηση έχει γίνει ε, μια επιτροπή ανεξαρτήτων εκτιμητών, προφανώ μιλάμε για μια πολύ πιο απλουστευμένη διαδικασία σε σύγκριση με αυτή που έχουμε, δηλαδή το, να είναι το δικαστήριο το αρμόδιο για την, για την εκτίμηση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ακριβώ ένα βιώσιμο μηχανισμό αγορά, να αυξήσουμε τη διαφάνεια και να βελτιώσουμε και τη διαθεσιμότητα δεδομένων. Και ε, πραγματικά βρίσκεται πολύ πίσω η χώρα μα σε σχέση με αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Είναι προφανώς ότι υπήρχαν ε, δεκάδες προβλήματα τα οποία σιγά σιγά έχουν μπει σε μια γραμμική νομοθεσία, έχει βελτιωθεί και ιδίω η διαδικασία υπολογισμού των αποζημιώσεων. Από τη στιγμή όμως αυτό που έχει γίνει και νομίζω ότι το κράτος πρέπει να σταθεί γενναία είναι να σταματήσει να συμπεριφέρεται λιγάκι πονηρά απέναντι στους ιδιοκτήτες ταλαιπωρώντας τους και να βάλει μπροστά την απευθείας εξαγορά, τον φιλικό διακανονισμό, ούτως ώστε όταν το κράτος θέλει να σχεδιάσει και να κάνει ένα ε, σημαντικό project ε, να, στο μεγαλύτερο ποσοστό των ε, ιδιοκτητών να συμφωνεί μαζί του σε μια φιλική διαφανή διαδικασία εκ των προτέρων και με αυτόν τον τρόπο και τα έργα θα γίνονται στην ώρα τους και τα ε, περιουσιακά δικαιώματα δεν θα θίγονται και ταυτόχρονα για όποιον δεν συμφωνεί θα υπάρχει δικαστική οδός να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει ε, το πλέον σημαντικό που επειδή ασχολούμαι και αρκετά χρόνια είναι αυτό το πράγμα, να φύγει όλη αυτή η ιστορία από την εμπλοκή με τα δικαστήρια, τους δικηγόρους. Πρέπει να εδρωθεί μια εμπιστοσύνη, όπως είπε και η κυρία Πότσου πριν, ότι οι προτινόμενες αξίες είναι οι πραγματικές, είναι οι market values, ότι το κράτος δεν πρόκειται να σε κοροϊδέψει, να αποζημιώνει το περιουσιακό δικαίωμα εξ ολοκλήρου και από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο οποίος έχουν απέναντί τους ε, στέκεται απέναντι με έναν δίκαιο τρόπο, οπότε δεν έχουν κανένα συμφέρον να εμπλακούν σε δικαστικές διαμάχες και να πάρουν τα χρήματά τους σε δύο, τρία, τέσσερα χρόνια και να δημιουργούν προβλήματα στο project και όλη αυτή τη σειρά γεγονόταν. Άρα νομίζω ότι ε, θα επαναλάβω ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει είναι η θέσπιση εθελοντικών διαδικασιών όπως ισχύουν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Äh, Ευχαριστώ προφανώ ε, οποιοδήποτε δηλαδή δικαστικό σύστημα σε οποιοδήποτε κράτο μέλο, αν βρισκόταν μέτωπο με τόσε υποθέσει, θα, θα, ήταν υπερφορτωμένο. Δηλαδή αυτό είναι αδιαφεσβήτητο όταν προβλέπεται μια τέτοια διαδικασία. Όμω, αν κατάλαβα σωστά, ε, ουσιαστικά αυτό τελικά αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει η ίδια η Ελλάδα. Δηλαδή, οι ελληνικέ αρχέ θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση ή όχι. Προφανώ υπάρχει εδώ ανάγκη να γίνει κάτι και θα ήταν ε, πολύ θετικό. Αλλά εσείς ε, ποιες θεωρείτε είναι οι πιθανότητες αν θέλετε να γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρξει δηλαδή μια επιτυχημένη αλλαγή και να ε, εφαρμόσετε τελικά ένα σύστημα το οποίο είναι αντίστοιχο με άλλα κράτη. για παράδειγμα, στη Γερμανία τέτοια εργαλεία όπως έχουμε αυτό του αναδασμού είναι, έχουν αποδείξει την αξία τους εδώ και πολύ καιρό και υπάρχουν όμως μηχανισμοί επίλυσης διαφορών οι οποίοι παρακάμπτουν τα δικαστήρια δεν αντιλαμβάνομαι τελικά γιατί δεν αλλάζει κάτι στην Ελλάδα. Γιατί δηλαδή δεν λαμβάνεται μια αποφάση να αλλάξει κάτι. Η ασφάλεια δικαίου δηλαδή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες διαδικασίες μπορεί να εξασφαλιστεί και εδώ. Οπότε αναρωτιέμαι γιατί δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αφού αποτελεί τόσο μεγάλο εμπόδιο για όλα αυτά τα ε, έργα. Και ακριβώ επειδή και αυτό το ε, ζήτημα δεν εξασφαλίζει ασφάλεια δικαίου. Ακριβώ γιατί η ασφάλεια δικαίου έχει να κάνει ακριβώ και με τι σχετικέ προθεσμίε, τη διάρκεια των υποθέσεων κ.ο.κ. Οπότε εσεί να σα ρωτήσω για μία ακόμα φορά ποιε θεωρείτε ότι είναι πιθανότητε επιτυχία, αν θέλετε, πιθανότητε να αλλάξει κάτι. Γιατί δεν θέλουμε σε δύο-τρία χρόνια να επισκεφθούμε και πάλι την Ελλάδα, να δούμε και πάλι τα έργα, τα συγχρηματοδοτούμενα και να διαπιστώσουμε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αν μπορούμε εμεί να κάνουμε κάτι από την πλευρά μα για να πιέσουμε τα πράγματα, να μα το πείτε. Θέλει να πάρετε πάλι το λόγο, παρακαλώ. Είναι εντάξει φιλοσοφικό το ερώτημα, μου το ξέρω, αλλά το θέτω παρόλα αυτά. Όχι, καταρχά νομίζω ότι είναι πολύ πρακτικό. Ο λόγο καταρχά που θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, που είχαμε τι πολύ πολύ μεγάλε καθυστερήσει αυτά τα χρόνια, ιδίω στα πέντε μεγάλα project τα οποία τον αυτοκινητοδρόμο πήραν και τη μερίδα του λέοντα από τον κρατικό προπολογισμό, δεν ήταν το γεγονό ότι δεν υπήρχαν νομικά εργαλεία. Υπήρχαν, αλλά δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ. Τα εργαλεία αυτά φτιαχτήκαν μια τριετία πριν γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ακριβώς για να πετύχουμε πολύ σφιχτέ πολύ χρονοδιογράμματα ε, και τότε. Και το ε, πολύ άσχημο κατά την άποψή μου είναι ότι αυτά δεν υπήρχαν. Άρα λοιπόν νομικά εργαλεία προκειμένου να μην έρθουμε αντιμέτωποι με αυτές τις καθυστερήσεις είχαμε αλλά δεν ενεργοποιήθηκαν. Τώρα, αν αυτά τα νομικά εργαλεία πραγματικά βρίσκονται λίγο στα όρια του, της προστασίας των περιουσιακών ε, δικαιωμάτων, ας πούμε, δηλαδή συζητώντας με κάποιους φίλους δικαστές μου λέγανε ότι έχουμε κάνει τόσο σφιχτές τις, ε, τις ε, προθεσμίες που έτσι εν είδη χιούμορ μου έλεγε ότι οδεύουμε προς το Σοβιετικό Σύνταγμα πλέον. Έτσι. Ε, ε, Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε εκεί. Είναι θέμα βούληση. Ότι όταν ξεκινά να κάνει ένα project και πει ότι ε, εγώ σε ένα χρόνο θέλω να ξεκινήσω να κάνω ένα project, είναι προφανέ από τη στιγμή που εσύ έχει πει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για την οικονομία τη χώρα, ότι θα βρω τον τρόπο και θα εφαρμόσω ό,τι ακριβώ χρειαστεί για να πάρω τη γη και να τη δώσω στον κατασκευαστή. Τώρα, το αν το νομικό αυτό εργαλείο χρήζει βελτίωση, ε, ε, είναι, επιτρέψτε μου την άποψη, είναι κάτι που είναι μια άλλη συζήτηση μεταξύ νομικών. Ε, μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να γίνει το project. Το θέμα είναι ότι θέλω τη γη και πρέπει να την αποκτήσω. Αυτά τα εργαλεία υπήρχαν, αλλά δεν χρησιμοποιηθήκαν ποτέ. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ε, προφανώ και υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσει και όπω σα είπα και πριν, ε, δεν ξέρω αν το ελληνικό κράτο μπορεί να γίνει τόσο γενναιόδωρο και να ξεκινήσει μια προσπάθεια ε, δημιουργίας μηχανισμών εξοδικαστικών ε, επίλυση των διαφορών. Νομίζω ότι ε, εσείς θα μπορούσατε ενδεχομένως να πιέσετε σε μια τέτοια κατεύθυνση, η οποία θα οδηγούσε και στην κατεύθυνση που περιγράψα, αυτή της ασφάλειας, της δημιουργίας ασφάλειας δικαίου πλέον. Αν συγκρίνω ε, την κατάσταση μεταξύ του γερμανικού και του ελληνικού συστήματος, να πω ότι στη Γερμανία υπάρχει καταρχήν εμπιστοσύνη ακριβώς των πολιτών ε, στο κράτος και αυτό Υποδεικνύεται και από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το κράτος. Δηλαδή ε, λέει το κράτος ότι θα υπάρξει μια ε, δίκαιη εκτίμηση και είμαστε διατεθειμένοι από την πλευρά μας να υπάρξει μια ένα φιλικό διακανονισμός. Δεν θέλουμε δηλαδή να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου τελικά θα μένουν κάποιοι χώρε ε, τη γη τους. Οπότε και ακριβώς ε, ε, χρησιμοποιείται και το ζήτημα της αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων χρήση. Γίνονται όλε σχετικέ διαδικασίε διαούλευση και ούτω καθεξή ακριβώ για να μην οδηγηθούμε στην κατάσταση ότι κάποιοι πολίτε δηλαδή να μην έχουν τελικά αυτέ τι γη του. Και ακριβώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια τέτοια προσέγγιση. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, όταν ε, υπάρχει ένας νόμος ε, και προβλέπει ε, συγκεκριμένη προθεσμία και ακολουθεί ένας ακόμα νόμος ο οποίος αναφέρει ότι αυτές είναι οι προθεσμίες και δεν είναι δυνατόν να αναβάλλονται είναι, είναι λίγο παράλογο. Δηλαδή να λέμε στον δεύτερο νόμο ότι δεν είναι δυνατόν να παραβιάζονται οι προθεσμίες του πρώτου νόμου ε, είναι κάτι το παράλογο. Χρειαζόμαστε λοιπόν αποφασιστικότητα, χρειαζόμαστε συνεργασία και θα πρέπει να κερδίσουμε και πάλι την πολιτών στο κρατικό μηχανισμό και νομίζω πως δεν ακολουθούμε την ε, σωστή κατεύθυνση αυτή τη στιγμή δυστυχώ ε, και πραγματικά με φοβίζει αυτό λίγο. Τι θέλεις; Ε, πιστεύω ότι όλα αυτά για να μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερή ανάπτυξη της ε, συνεργασίας με τον, τον θυγόμενο ιδιοκτήτη, ούτως ώστε να έχουμε σαφή και συγκεκριμένα αποτελέσματα στην, ε, ε, στην, στο φιλικό διακανονισμό. Ε, θέλει πρώτον να, να οι εμπορικές αξίες να αντικατασταθούν οι αντικειμενικές αξίες από τις εμπορικές αξίες. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών ε, εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και έχει υποσχεθεί στο, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να, να, να στήσει ένα αξιόπιστο σύστημα εμπορικών αξιών, δηλαδή να αντικαταστήσει τις αντικειμενικές αξίες. Αντιλαμβάνεστε ότι ε, επειδή το εγχείρημα είναι νέο, ε, θα χρειαστεί κατά την άποψή μου χρόνος για να αποκτήσει μια αξιοπιστία το νέο σύστημα των εμπορικών αξιών. Ε, και μην ξεχνάμε ότι λόγω της μεγάλης πτώσης αξιών της, ε, των ακινήτων στην Ελλάδα λόγω της ε, οικονομικής κρίσης έχει δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόσκομα στο να μπορέσουμε να βρούμε πάλι τις εμπορικές αξίες ε, των ακινήτων στη χώρα μας. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι για τους φιλικούς διακανονισμούς προϋποθέτει και ένα σώμα εμπειρογνωμόνων πιστοποιημένων εκτιμητών όπου πράγματι θα έχουν κερδίσει την αξιοπιστία τους μέσα από την πραγματική αγορά. Ε, όπως ξέρετε υπήρχε ε, ένα σώμα ορκωτών εκτιμητών από το 1978 το οποίο λειτουργούσε μέχρι το 2012 λειτουργούσε σε ένα περιορισμένο ε, καθαρά περιβάλλον Επομένως δεν καν, ο κόσμος καν δεν το γνώριζε ότι υπήρχε αυτό το σώμα αρκωτών εκτιμητών εκτός από τους εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας. Ε, από το 2013 που θεσμοθετήθηκε πλέον και άνοιξε το επάγγελμα των πιστοποιημένων εκτιμητών. Πράγματι τώρα υπάρχουν από ό,τι ξέρω στο Μητρό εγγεγραμμένοι 400 φυσικά πρόσωπα και 50 εταιρείε ε, εκτιμητών, ε, οι οποίοι θα πρέπει ε, να αποκτήσουν και να διασώσουν δηλαδή την αξιοπιστία, να, ενδυναμώσουν την αξιοπιστία του θεσμού στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική αγορά, ούτω ώστε μετά να καρποθούμε και εμείς σαν διαχειριστές της απολυτρίωσης την αξιοπιστία των εκτιμήσεων ε, που θα μπορέσουν να επιτρέψουν να συνεργαστούμε με τους ιδιοκτήτες της γης. Πλέον των άλλων, δηλαδή που θα πρέπει να συμπληρωθεί και από το, έναν ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί είμαστε πάλι πίσω εκεί. Γίνεται μια προσπάθεια από τις περιφέρειες σήμερα που ξεκίνησε από το 2011 και συντάσσονται γενικά πολυδομικά σχέδια, ειδικά στους μεγάλους δήμους της, της ελληνικής περιφέρειας και ας ελπίσουμε ότι αυτά στην επόμενη πενταετία ε, θα μπορέσουμε να έχουμε ασφαλέστερα εργαλεία για να μπορούμε να ελευθερωθούμε σαν διαχειριστές της απολυτρίωσης και να πάμε σε μια ε, καλύτερη συνεργασία με τους ε, θυγόμενους ιδιοκτήτες και να μην αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε εξαιρετικά μέτρα τα οποία πολλές φορές αδικούμε και δημιουργούμε κοινωνικά ακόμα και κοινωνικά προβλήματα. Ε, ήταν και μια άλλη ιδέα που θα μπορούσε το... και έχει γίνει μια σχετική συζήτηση είναι να οι, οι και η απαλωτρίωση να αυτονομηθούν από την ανάθεση του έργου. Δηλαδή να προηγούνται ε, οι απαλωτριώσεις και η, και η διαχείριση όλων των αδειοδοτήσεων, δηλαδή ε, ο έλεγχος των αρχαιολογικών ανασκαφών, οι μετατοπίσεις των δικτύων κοινής ωφέλειας, ε, να προηγούνται σε μια, σε μια διαδικασία χρονική πολύ πριν ανατεθεί και τότε μόνο να ανατίθεται το έργο ε, για να μπορεί να μην επηρεάζεται από αδειοδοτήσεις, από απαλωτριώσεις ε, και να υπάρξει ένα ε, τουλάχιστον μία μη διατάραξη της, του χρονοδιαγράμματος του, του, του έργου. Αυτά ευχαριστώ. Ja, vielen Dank, Renault. Κύριε Σλάουτερς, ε, κύριε Ρενό, τι θα κάνουμε από εδώ και μετά. Και εσείς προφανώς ε, ελπίζετε τα πράγματα να βελτιωθούν, αλλά δεν φτάνει αυτό. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας συγκεκριμένα. I think that Professor Potsu has... Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυρία Πότσιου έθιξε τα πράγματα επακριβώς. Είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν οδηγήσει σε προβληματικές καταστάσεις, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το ζήτημα της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης. Αν ο πολίτης δεν εμπιστεύεται τη διαδικασία παλωτρίωσης που ακολουθεί το κράτος και αν ο πολίτης δεν πιστεύει τελικά ότι όλη η διαδικασία είναι διαφανής Ιδίω η διαδικασία εκτίμησης της αξίας του ακινήτου του, τότε προφανώς ο πολίτης αυτός θα συνεχίσει να προσφεύγει συνεχώς στα δικαστήρια. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Αν λοιπόν πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα εν προκειμένου, πρέπει αφενός να δώσουμε στην Ελλάδα όλη την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη, όλα τεχνικά μέσα, δηλαδή κλιμα, ε, κτηματολόγιο το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά και άλλα τεχνικά μέσα, προκειμένου όλη η διαδικασία απαλωτρίωσης να γίνει διαφανής. Και διαφάνεια χρειαζόμαστε βέβαια σε όλη τη διαδικασία, αλλά ιδίω στο ζήτημα της απαλωτρίωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο πολίτης να πιστεύει ότι πραγματικά αποζημιώνεται δικαίω για την ιδιοκτησία την οποία παραχωρεί στο κράτος. Αυτό είναι ουσιώδου σημασίας. Από την άλλη, και στο ίδιο πνεύμα χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιεί αυτόν τον υφιστάμενο μηχανισμό των εξάρτητων εκτιμητών. Οι ανεξάρτητοι αυτοί εκτιμητές αποτελούν τεράστιο βήμα πρόοδου σε σχέση με το καθεστώς το οποίο προϋπήρχε στην Ελλάδα. Νομίζω όμως ότι μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες αυτούς τους ανεξάρτητους εκτιμητές αν μείνουμε λίγο περισσότερο στον τρόπο πιστοποίησή του, αν διασφαλίσουμε ότι όντω δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίω σε σχέση με τη γη εκείνη την οποία καλούνται να αποτιμήσουν και το καθεξής. Πρέπει να επιμείνουμε πιστεύω στα σημεία αυτά. Κάθε φορά που ερχόμαστε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές. Νομίζω ότι σε αυτά τα σημεία θα πρέπει να επιμείνουμε και επ' αυτών των σημείων θα συνεχίσουμε την εργασία μας με την ελληνική πλευρά, ο Σεβαστιάν. Να προσθέσω απλώς ότι συμφωνώ προφανώς απόλυτα με τα όσα είπε ο Βίλι Ο διοκτήτης, ακίνητης περιουσίας επίσης θα πρέπει να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει ότι το κράτος θα προχωρήσει σε απαλωτρίωση με τρόπο γρήγορο και ότι δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από την αποτίμηση μιας δίκαιης τιμής. Αυτή τη στιγμή καθοριστεί μια δίκαιη λοιπόν τιμή και αυτή τη στιγμή ο πολίτης θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένα παραθυράκι στο όλο σύστημα, τότε δεν θα χρειάζεται να προσφεύγει και στη δικαιοσύνη τόσο συστηματικά. Θα καθορίζεται λοιπόν εκ των προτέρων η τιμή αυτή, πράγμα το οποίο γίνεται και στη δική μου χώρα και στη δική σας τη χώρα και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία της απαλωτρίωσης. Ως προς αυτό λοιπόν, και αν με ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι όλη η συλλογική εργασία που έχει γίνει από τους Έλληνες και τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδήγησε σε μια διαδικασία που είναι βελτιωμένη τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο σε σχέση με αυτό που είχαμε στο παρελθόν και έχουμε και στα πλαίσια του μνημονίου κατανόησης του μνημονίου αυτού για το πρόγραμμα προσαρμογής συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένες προθεσμίες. Αυτό σε συνδυασμό με την στρατηγική που ακολουθείται για την καταπολέμηση των φαινόμενων απάτης όσον αφορά τα κοινοτικά κονδύλια έχει οδηγήσει σε νέα συστήματα ελέγχου, σύμφωνα με τα οποία καλούνται να λάβουν δράση οι ελληνικές αρχές στα πλαίσια των σχεδίων απαλωτρίωσης. Ήδη έχουν λάβει όμως σχετική δράση οι ελληνικές αρχές, έχει σημειωθεί ήδη πρόοδος και ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα οδηγηθούμε πλέον σε μία μόνιμα βελτιωμένη διαδικασία. Μια διαδικασία που δεν θα λύνει τα προβλήματα μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Σα ευχαριστώ πολύ για όλε αυτέ τι πληροφορίε και για την ανταλλαγή των απόψεών μα. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και πολύ χρήσιμη για μα για να αντιληφθούμε βέβαια τι κρύβεται πίσω από αυτά τα προβλήματα τα οποία και εμεί ε, εμπιστώσαμε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλου ε, καλή επιτυχία. Πραγματικά για το έργο σας από εδώ και πέρα και ε, ήταν πολύ σημαντικό το, το οποίο το γεγονό ότι ήρθατε σήμερα εδώ στι ε, Βρυξέλλε για να σα ακούσουμε. Ε, ολοκληρώσαμε λοιπόν με το πρώτο τμήμα του workshop και περνάμε στο δεύτερο τμήμα, δηλαδή την ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά τι εργασίε τη Task Force για την Ελλάδα. Ε, και ε, θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τον ε, κύριο Μουγκουρούτσα, ε, ο οποίο είναι το αρμάδιο μέλο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ο δικό μα εισηγητή είναι ο κύριο Στόιρα, ο οποίο εκπροσωπείται σήμερα από τον κύριο Άλλη. Και να δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Μουγκουρούτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλου. Αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Ε, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά ε, για την πρόσκλησή σας ε, προκειμένου να σας παρουσιάσω τα πορίσματα μιας ακόμα μελέτης την οποία διεξήγαμε από την πλευρά του Ελεκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έγγραφο το οποίο συνέταξε ο εισηγητής σας ο κύριος Τόιρο. Το εν λόγω έγγραφο συνοψίζει αντικειμενικά ε, την ε, έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου και θεωρώ πως ε, μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για την συζήτηση της έκθεσης. Έκθεση λοιπόν αυτή την οποία θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι η πρώτη του Ελεκτικού Συνεδρίου που ασχολείται με την ελληνική κρίση και καλύπτει την τεχνική βοήθεια που έλαβε η Ελλάδα υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα στο πλαίσιο της Task Force για την Ελλάδα ή με τα αρχικά γνωστό TFGR. Θα ήθελα επίσης να σας ανα πέρο ότι αυτή την περίοδο προετοιμάζουμε μία άλλη ε, έκθεση που επίσης αφορά την ε, κρίση στην Ελλάδα και ασχολείται ειδικότερα με την διαχείριση του προγράμματος χρηματοδοτικής ε, συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν λόγω έκθεση λοιπόν θα είναι έτοιμη ε, για δημοσίευση στις αρχές ε, του 2017. Ας εστιάσω όμως τώρα στην ε, έκθεση για την οποία μιλάμε σήμερα. Η εν λόγω λοιπόν έκθεση αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, δηλαδή την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο σύστημα, ε, πρόγραμμα ε, χρηματοδοτικής ε, συνδρομής για την Ελλάδα. Η εν λόγω λοιπόν υποστήριξη παρασχέθηκε από την Επιτροπή μετά από σχετικό αίτημα της Ελλάδας και προκειμένου να ανταποκριθεί και να δώσει αυτή την βοήθεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε αυτή την Task Force για την Ελλάδα η οποία ανέλαβε τις εργασίες της τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Ελλάδα και το Φεβρουάριο του 2015 είχε προσωπικό 65 άτομα. από αυτή την άποψη θεωρούμε πως ε, ε, η τεχνική αρρωγή ε, που δόθηκε στην Ελλάδα έτυχε μιας αποτελεσματικής διαχείρισης και συνέδραμε στις διαδικασίες της μεταρρυθμιστικές. Θα ήθελα να εστιάσω ειδικότερα σε τρία ζητήματα. Καταρχήν τη δημιουργία της Task Force σε ό,τι αφορά δηλαδή, την οργανωτική της φύση, τη χρηματοδότησή της, τον, το χρονοδιάγραμμα των δρασιών Δεύτερον μετά, ε, τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε στην εντολή της αυτή η Task Force, όπως αναφέρεται και στο, στον πίνακα 1 ε, της έκθεσης. Και ε, τρίτον, στο πώς συνέβαλε στην πρόοδο που επιτέθηκε σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Και για να το επιτύχουμε αναλύσαμε ένα δείγμα των αναθέσεων που είχε η, η Task Force αυτή για την τεχνική αναλογή σε πέντε τομείς πολιτικής και όπου εστιάσαμε ειδικότερα στην δημόσια διοίκηση, φορολογικέ μεταρρυθμίσει και το επιχειρησιακό περιβάλλον. Ποια είναι λοιπόν τα συμπεράσματά μα. Είναι μεικτού χαρακτήρα, ήταν μεικτά τα συμπεράσματα. Δηλαδή, από τη μία πλευρά δημιουργήθηκε πράγματι ένα ευέλικτο μηχανισμό για τον συντονισμό ενό ευρέω προγράμματο τεχνική βοήθεια. Ε, αυτή η βοήθεια ε, δόθηκε αποτελεσματικά, ε, αφορούσε τα λόγω προγράμματα και ευθυγραμμιζόταν με το πρόγραμμα αναπροσαρμογής. Ε, επίσης, ε, ανέπτυξε η Task Force διαφοροποιημένα συστήματα για την παροχή της τεχνικής ε, βοήθεια και για, την, για τον συντονισμό των project, η οποία βοήθεια ήταν και καινοτόμα Επίσης και η παρακολούθηση της προόδου της τεχνική βοήθειας ήταν αποτελεσματική. Από την άλλη πλευρά ωστόσο θεωρούμε πως η τεχνική ε, συνδρομή η οποία δόθηκε δεν επηρέασε πάντοτε την ε, πρόοδο που επιτέχθηκε σε ε, σχέση με τις μεταρρυθμίσεις και αυτό βέβαια αποτελεί ένα από τους βασικούς δείκτες τελικά για την επιτυχία των εργασιών της Task Βέβαια το πολύ μετάβλητο πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έπαιξε τον αποφασιστικό ρόλο. Επίσης η Task δημιουργήθηκε πάρα πολύ γλίγορα ακριβώς για να ανταποκριθεί στην κρίση στην Ελλάδα και έτσι η Επιτροπή δεν ανέλησε πλήρως τις άλλες εναλλακτικές που είχε στη διάθεσή της ούτε προέβλεψε ένα ξεχωριστό προπολογισμό για την Task Force. Επίση, δεν υπήρχε κάποιο στρατηγικό έγγραφο το οποίο θα ανέφερε και με βάση το οποίο θα μπορούσαν ε, να ε, ιεραρχηθούν ως προς την τους οι διάφορες δράσεις τεχνικής συνδρομής της Task Force. Ε, συγκεκριμένα δηλαδή στην πράξη η Task Force συχνά δεν, είχε, δεν αναλάμβανε την πρωτοβουλία για την ε, παροχή της βοήθειας και ενεργοποιούνταν μετά από αίτημα της της ελληνικής ε, πλευράς ε, και θεωρούμε ότι θα μπορούσε να έχει παρακολουθήσει καλύτερα η Task Force τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές της Ελλάδας ακολουθούσαν τις συστάσεις και τον αντίκτυπο της τεχνικής ε, βοήθειας. Τέλος, διαπιστώσαμε ότι σε ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα η δημόσια διοίκηση, ο φορολογικός τομέας, η πρόοδος σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις όπως αυτή επηρεάστηκε ακριβώς από τη τεχνική βοήθεια, δεν ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη. Οπότε τι ποιε είναι οι συστάσει από τη δική μα πλευρά. Έχουμε, ε, έχουμε κάνει μια ε, σειρά από συστάσει, ούτω ώστε να υπάρχει μια σαφή στρατηγική με καλώ ορισμένου στόχου και καλώ ορισμένε προτεραιότητε. Θεωρούμε πω ε, θα πρέπει να ενδυναμώνεται μέσω της τεχνικής βοήθειας η δυνατότητα που έχουν οι εθνικές ε, δημόσιες διοικήσεις, ώστε να υπάρχει και υπηρεσιακή συνέχεια και βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων. Επίσης, έχουμε κάποιες συστάσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την Επιτροπή να εκτελέσει και άλλα τέτοια ε, ε, προγράμματα τεχνικής βοήθειας, άλλα κράτη-μέλη. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, Παρότι λοιπόν η Task Force ε, απέδειξε την αξία της ως ένας μηχανισμός για την παροχή τεχνικής ε, βοήθειας και μάλιστα περίπλοκης τεχνικής βοήθειας, υπήρχαν κάποιες αδυναμίες σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό της όλης διαδικασίας και υπήρξαν και μεικτά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο τελικά που είχε αυτή η τεχνική βοήθεια στην πρόοδο των ε, μεταρρυθμίσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και βρίσκομαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήματα. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο κατευθείαν στον κύριο, κύριο Άλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητέ εκπρόσωπε του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, δυστυχώς ο κύριος Στόιερ δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας, γι' αυτό μου ζήτησε εξ ονόματός του να, να παρουσιάσω τη δήλωσή του αυτή για την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα αποτελέσματα στα πλαίσια της παροχής τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα. Έκθεση 19 του 2015 ολοκληρώθηκε το 2015 ο έλεγχος αυτός και παρόλα αυτά κρεμούν πάρα πολλά ακόμα ζητήματα όσον αφορά τα έργα εκείνα τα οποία έλεγξε το Ευρωπαϊκό Αλλακτικό Συνέδριο. Οι πιο βασικές δυσκολίες έγκυται στο ότι δεν υπήρχε καταρχάς ένας ειδικό προπολογισμό, αυτό οδήγησε σε μια κάποια σύγχυση όσον αφορά την πρόσληψη των εμπειρογνωμόνων. Παρόλα όλα αυτά υπήρχε μια συγκεκριμένη εντολή που πήρε τη μορφή Task Force, η οποία έπρεπε παράλληλα να ασχοληθεί με πολλά διαφορετικά έργα σε πολλού διαφορετικού τομεί. Η Task Force επίση δεν κατάφερε να υποβάλει τριμηνία έκθεση προόδου και μέχρι στιγμή δεν έχει υποβάλει τελική ακόμα έκθεση τον Νοέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία πρόταση για το πρόγραμμα το οποίο θα διαδεχθεί την Task Force. Πρόκειται για το πρόγραμμα υποστήριξης διαστροτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020. Και στο πρόγραμμα αυτό προβλέπονται πολλές από τις συστάσεις που έκανε το ελεκτικό συνέδριο το, τη διαδικασία απαλλαγή του 2015 θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της ε, Task Force, καθώς επίσης και η έκθεση αυτή του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντλήσουμε τα παρέτα διδάγματα από την έκθεση αυτή του λεκτικού συνεδρίου που θα πρέπει να αποτελέσουν βάση για οποιοδήποτε μελλοντικό πρόγραμμα τεχνική βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον να υπάρχει ειδικό προπολογισμό, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένοι στόχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιτηρεί εκ του σύνεγγυ την πρόοδο των διαφόρων έργων για τα οποία δίδεται τεχνική υποστήριξη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συμφωνεί μαζί με τα κράτη-μέλη για μια απλουστευμένη διαδικασία πρόσληψης εθνικών εμπειρογνωμόνων. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση από τα κράτη-μέλη που θα βασίζεται στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα και κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά όσο και το Κοινοβούλιο να συμβάλλει για την καλύτερη χρησιμοποίηση του ειδικού αυτού προπολογισμού. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και το σύνολο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για την επικοδομητική τους αυτή έκθεση και να ευχαριστήσουμε επίση την κυρία Σνάιντερ και του υπόλοιπου συναδέλφου για τη συμβολή του. Ο κύριο Στόιερ επίση μου ζητά να θέσω κάποια ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και πιο συγκεκριμένα αν έχουν ήδη κάποιες ενδείξεις για την υποβολή της τελικής έκθεσης αλλά και της τριμηνιαίας έκθεσης η οποία δεν είχε υποβληθεί και η οποία βέβαια προβλεπότανε. Εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού μπορούμε να επιτελέσουμε το έργο μας αν υποβάλλονται οι συγκεκριμένες εκθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση των προγραμμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην βρεθούμε στην να μην βρεθούμε στο μέλλον στην κατάσταση που βρεθήκαμε με αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνική υποστήριξη. Επομένω, ποια είναι τα διδάγματα τα οποία έχουμε αντλήσει μέχρι στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό επίση να μεταρρυθμιστεί το σύστημα τη διοργάνωση των προγραμμάτων αυτών, ιδίω όσον αφορά την πρόσληψη πυρογνωμόνων. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντική και ενδιαφέρουσα έκθεση. Και ε, με οδήγησε σε κάποιες σκέψεις, γιατί μέσω ακριβώς ε, ε, αυτής της έκθεσης προσπαθούσαμε να, προσπαθήσαμε να δούμε και τι ακριβώς έκανε η Task ποιες ήταν τα αρμοδιότητά της και τα αποτελέσματα της. Ε, η κυρία Γιαλά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους συναδέλφου που δεν ήταν δυνατό να βρεθεί σήμερα εδώ γιατί είχε κάποιο άλλη, κάποια άλλη εκδήλωση στο πρόγραμμά του. Μου ζήτησε να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Παρνιό τονίζει στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου πως η τεχνική βοήθεια δεν επέτρεψε να προοδεύσουν αρκετά οι μεταρρυθμίσεις, δεν προώθησε αρκετά τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, δεν είναι ικανοποιητικές οι μεταρρυθμίσεις ε, στο βαθμό που έγιναν. Η Task Force παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης χωρίς όμως να πρικοδοτηθεί με ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει εκ των προτέρων. Και επίσης αυτό που εντοπίζει στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι οι αδυναμίε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν ε, κάποια έργα ή τα κριτήρια επιλογής, ε, το γεγονός ότι αρκετές φορές δεν ενευνήθηκε σε βάθος αυτό που έπρεπε να γίνει και ο κύριος Παρνιό ε, συμμερίζεται τις συστάσεις του κύριου Τόιρερ και συμφωνεί πως είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης πριν προσφέρεται τεχνική βοήθεια. Επίσης, θεωρεί πως είναι θλιβερό το γεγονός πως η Task Force δεν ε, υπέβαλε τακτικές εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο θα προωθούσε με καλύτερο τρόπο τις μεταρρυθμίσεις που ήταν απαραίτητε και τα άλλα θέματα που είχε στην ατζέντα της η Task Force και κάτι που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ότι στήθηκε στα γρήγορα Πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις συστάσεις και στην μονάδα για τη στήριξη των, ε, των διαστατικών μεταρρυθμίσεων έχει κάνει πολλές βελτιώσεις που θα βοηθήσουν στο μέλλον. Ωραία. Έχω μία ερώτηση για το ελεγκτικό συνέδριο. Στην έκθεση δεν βρίσκω α, πόσο κόστισε το εργαλείο αυτό, η Task Force. 11 ή 14 εκατομμύρια. Δηλαδή, να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει με τα υπόλοιπα εκατομμύρια τα οποία έχουν χορηγηθεί και να δούμε σε ποσοστό η τεχνική βοήθεια τι κόστησε. Γιατί έχουμε τα όσα συνέβησαν με το 2011, έχουμε και την περίοδο 2011-2014. Ε, Δεύτερον, από τα έργα τα οποία εντοπίζονται ε, που, στον κατάλογο που μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να μου πείτε οι ομάδες για την τεχνική βοήθεια που φαίνονται στη σύσταση 4 και όπου μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως οι ομάδες αυτές αποτελούνται από εμπειρογνώμους διεθνείς της Κομισιόν, ε, εθνικούς, ε, αποσπασμένους κτλ και έκανα και κάποιες αποστολές μακράς διάρκειας και κάποιες βραχίας διάρκειας. Δηλαδή είχε μια μεγάλη, ε, μια πληθώρα ε, τύπων ε, εμπειρογνωμόνων. Θα θέλαμε να δούμε τι κόστησαν όλα αυτά, τι είδους ήταν αυτές οι ομάδες εμπειρογνωμόνων, ε, με πιο πολλές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ε, κάτι αντίστοιχο είδαμε και στην Ουκρανία. Δηλαδή το πώς επιτροπές ε, δημιουργούνται για την υποστήριξη της χώρας και ούτω ε, This is another example of where the European Ευχαριστώ. Νομίζω πως εδώ πρόκειται για ένα ε, τομέα όπως εκείνος για παράδειγμα κατά τη δημιουργία του ευρώ που δεν υπήρχε, υπήρχε πλήρης απουσία του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν υπήρχε σχεδιασμό και ούτω καθεξής ε, κάτι είχαμε εδώ αυτή τη στιγμή αλλά δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό οπότε εγώ θα ήθελα να θέσω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα ε, αναφέρεται ω ελεκτικό συνέδριο ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητε και του ε, στόχου και θα πρέπει να υιοθετείται και από το ε, δικαιούχο, δηλαδή το κράτο μέλο, το οποίο θα λάβει αυτή την αρρωγή. χαμογέλασα όταν το διάβασα αυτό, γιατί τι σημαίνει ότι δηλαδή το κράτο μέλο θα είναι υποχρεωμένο να αποδέχεται οτιδήποτε τελικά το επιβάλλεται από αυτήν την task force ω τεχνητή βοήθεια. Δηλαδή, εάν δεν συμμορφωθεί, τότε δεν θα λάβει την υποστήριξη. Από εκεί και μετά αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει feedback στοιχεία δηλαδή από τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν την ε, τεχνική βοήθεια. Αυτό τι σημαίνει ότι θα είναι δυνατόν και ε, ε, οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, για παράδειγμα, να κάνουν τα σχόλιά του σε ό,τι αφορά την ε, τεχνική βοήθεια και την αποτελεσματικότητά του. Σε ό,τι αφορά την έκθεση του εισηγητή, πραγματικά συμφωνώ ότι είναι ελπιδό το γεγονό ότι δημιουργήθηκε σε τέτοιο καθεστώ επανικού μια τέτοια task force και πράγματι θα πρέπει να υπάρξει καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό κατά την δημιουργία μια τέτοια ομάδα. Και από εκεί και μετά ελπίζω ότι θα έχουμε λάβει τα διδάγματά μα από, ε, όσα έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη λήψη υπόψη και των απόψεων των οργανώσεων τη κοινωνία ε, ε, των ε, πολιτών κατά τη δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων. Πάντω, πραγματικά έκανε καλή δουλειά ο συγκεκριτή. Ευχαριστώ. Ε, Κύριε κυρία Μακάρτη, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα εδώ. Έχετε το λόγο, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ε, θα ήθελα καταρχήν ε, να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα και μετά να δώσω στον συνάδελφο το λόγο σε σχέση με το ερώτημα που ε, τέθηκε. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σχολιάσουμε αυτή την έκθεση του Ελεκτρικού Συνεδρίου και ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη συστάση της έκθεσης του. Πραγματικά θεωρούμε πως έρχεται σε κατάλληλη χρονική στιγμή η εν λόγω έκθεση γιατί αυτή την, ε, σε αυτή τη χρονική συγκυρία ξεκινάει ακριβώς τη συζήτησή του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά ε, την πρόταση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά ένα ε, πρόγραμμα διαρθωτικής υποστήριξης το οποίο ε, θα αντικαταστήσει ακριβώ το μηχανισμό τη τεχνική βοήθεια προ όλα τα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο δημιουργείται αυτή την ε, περίοδο βασίζεται στα διδάγματα τα οποία αντλέσαμε από την ε, Task Force για την Ελλάδα και την Task Force για την Ελλάδα και τη σχετική τεχνική βοήθεια. Το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι η βοήθεια η οποία παρασχέθηκε αφορούσε τους σχετικούς στόχους και ευθυγραμμιζόταν με το γενικότερο πρόγραμμα της ε, χρηματοδοτικής ε, ε, συνδρομής και χαιρόμαστε το γεγονό ότι αναγνωρίζω ότι παρά τα πάρα πολύ στενά χρονικά περιθώρια που είχαν παρά το, το, την κρίση και παρά το δύσκολο πολιτικό κλίμα, η Task Force κατάφερε να δημιουργήσει ένα ευέλικτο σύστημα παροχή τεχνική βοήθεια προ τι αρχέ τη Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει που αντιμετώπισαν στο επίπεδο τη εθνική οικονομία και μάλιστα πάρα πολύ Ε, Θα ήθελα να να αναφέρω ότι η ε, επιτυχής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ε, ε, αποτελεί ευθύνη τελικά των εθνικών αρχών. Εμείς παρέχουμε δηλαδή τεχνική βοήθεια, αλλά από εκεί και μετά αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών να εφαρμόσουν τα όσα λαμβάνουν στο επίπεδο της τεχνικής βοήθειας. Κατά πώς θεωρούν πως είναι το καλύτερο. Επίσης θα θέλαμε να πούμε ότι η υπηρεσία διαρθρωτικής ε, υποστήριξης ε, δημιουργήθηκε τον Ιούλιο ε, του 2015 και βρίσκεται ακριβώς σε προπαρασκευαστική φάση προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί από το 2017. Εν λόγω λοιπόν η υπηρεσία που αναφέρθηκε στην έκθεση θα παρέχει στόχοθετημένα τεχνική βοήθεια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος τη ζητήσει. Επίσης, η πρόταση για το πρόγραμμα, για αυτό το νέο πρόγραμμα διορθωτικής υποστήριξης ε, υιοθετεί κάποιες από τις συστάσεις που έγιναν ε, με βάση ε, τα αποτελέσματα των εργασιών της Task Force για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προβλέπει μια πιο στρατηγική προσέγγιση σε ό,τι αφορά ακριβώ την παροχή της τεχνικής βοήθειας. θέτει συγκεκριμένους στόχους σε ό,τι αφορά και τον σχεδιασμό της παρεχόμενε βοήθειε και επίση ε, προβλέπει ένα μηχανισμό παρακολούθηση των δράσεων ε, που λαμβάνονται ε, και επίση τη βοήθεια η οποία παρέχεται. Οπότε βλέπετε ότι ήδη σε αυτό το πρόγραμμα που προετοιμάζουμε έχουμε λάβει υπόψη μα σχετικέ συστάσει. Άρα λοιπόν η Επιτροπή ελπίζει όπω και ο εισηγητή πω το εν λόγω αυτό πρόγραμμα θα αναδειχθεί σε ένα σημαντικό εργαλείο για την παροχή της θερμικής βοήθειας και ελπίζουμε πως επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου θα αποτελέσει το πρώτο σωστό βήμα προ αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, απαντώντα στα ερωτήματα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τι εκθέσει τη ε, Task Force για την Ελλάδα. Να πούμε ότι δεν είχε προβλεφτεί να συνταχθεί μια τελική έκθεση. Δηλαδή, είχαμε τίσσε εκθέσει που είχαν ε, προβλεφθεί από την Task Force, απλά για να το διευκρινίσω. Επίση, ε, η Task Force απορροφήθηκε τελικά από το Παγκόσμιο Σύστημα SRSS, οπότε ε, συνεχίζεται αυτή η παροχή της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του SRSS και SRSS και από εκεί και μετά. Ε, σε ό,τι αφορά τα 115 έργα τα οποία με τα οποία ασχολήθηκε η Task Force ε, και το πώς, δηλαδή πόσο χρόνο δαπάνησε στην εξέτασή του η Επιτροπή. Ε, αυτό δεν αποτελούσε έργα για τα οποία υπάρχει τεχνική βοήθεια η Task Force, απλά έργα τα οποία ελοποίησε με χρηματοδότηση των διαφορετικών ταμείων ε, η Ελλάδα. Είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε σχέση με αυτά τα project. Από εκεί και μετά. Ε, να πούμε ότι συμφωνούμε ε, με το συμπέρασμα της έκθεσης ότι δηλαδή δεν ήταν θετικό το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένα ξεχωριστό ταμείο, ένας ξεχωριστός προϋπολογισμός. Άρα λοιπόν ε, τα κονδύλια που χρησιμοποιήθηκαν εδώ ήταν κονδύλια τα οποία είχαν επιστραφεί από τι χρηματοδοτήσει των ιδιωτικών ταμείων από την Ελλάδα στην Επιτροπή. Και αυτό βέβαια αποτελεί ε, πάντοτε ένα μειονέκτημα τέτοιο μηχανισμό, όταν δηλαδή δεν έχουν το δικό του ταμείο, το δικό του προπολογισμό. Και προσπαθούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα μέσω ακριβώ του ε, προγράμματο τη ιδιωτική Υποστήριξη. Δηλαδή ζητάμε εκεί σε αυτό το πρόγραμμα να υπάρχει ένα ε, ταμείο, ένα ξεχωριστό προπολογισμό, ο οποίο θα μα επιτρέπει ακριβώ τον κατάλληλο σχεδιασμό παροχή τεχνική τις βοήθεια με βάση τα αιτήματα που θα λαμβάνουμε. Σα ευχαριστώ για τα ερωτήματα που μα θέσατε. Συνάδελφος Βόγκεν, ένα ερώτημα προς την Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο πράγματα θα ήθελα να θίξω και συγγνώμη που παίρνω μόλις τώρα το λόγο. Ερωτήματα και παρατηρήσεις προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ελληνικό Συνέδριο. Πρώτον, όσον αφορά την τεχνική βοήθεια η οποία δόθηκε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει, αλλά και για προγράμματα τη πολιτική συνοχή υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες προγραμμάτων. Από κοινού, από ό,τι κατάλαβα, γίνανε πολλά πράγματα και εφόσον παρέχει κανείς τέτοια τεχνική βοήθεια από πολλές διαφορετικές πλευρές, είναι σημαντικό να δούμε αν υπάρχουν συνέργειες. Πρώτον αυτών, δεύτερον. Γενική καταρχάς ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπήρχαν συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα από τις διαρθρωτικές αυτές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να είναι πολύ πρόημο για να μου δώσετε μία απάντηση, ενδεχομένως όμως να μπορούσε να ασχοληθεί περαιτέρω με αυτό ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ελεκτικό Συνέδριο, προκειμένου να αξιολογηθούν τελικά οι ήδη επιτευχθήσεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. κυρία Γιάλα ήθελε να θέσει επιτευχθησεις διαρθρωτικε μεταρρυθμισεις στην ελλαδα η κυρια να θεσει Ευχαριστώ καταρχήν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντηση που μας έδωσε, αλλά δεν ήταν πολύ στοχευμένη, ήταν λίγο γενικόλογη και λίγο για το μέλλον. Θα ήθελα να μου στείλετε τα στοιχεία, αν δεν μπορείτε να μου το δώσετε τώρα, αλλά θέλω και το κατάλογο αυτό για τα 218 έργα, με το ποιες ήταν οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων που ασχολήθηκαν και πόσο κόστησαν και ποιο οργάνωσε αυτέ τι ομάδε, γιατί είπαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πω η εφαρμογή ε, έγινε από το κράτος μέλος, αλλά το κράτο μέλος δεν οργάνωνε το ποιοι εμπειρογνώμονε θα πάνε. Αυτή η τεχνική βοήθεια από ποιους προσφέρθηκε. Πώς επιλέχθηκαν οι εμπειρογνώμονες αυτοί, με ποιο τρόπο και πόσο κόστησε. Γιατί αποφάσισε ποια θα είναι οι ομάδε αυτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φαντάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση μετά έπρεπε με του εμπειρογνώμονε αυτού να κάνει κάποια δουλειά. Είχαμε αυτόν τον κατάλογο με 118 έργα προτεραιότητες στα έγγραφά μας νομίζω. Δηλαδή είχαμε λάβει αυτό τον κατάλογο πριν από την επίσκεψή μας, ε, επιλέξαμε 7 αιματοληπτικά. 118 περιλαμβανόνταν ε, αρχικά σε αυτό το κατάλογο, εν πάση περιπτώσει θα μπορεί να σας αποστείλει αυτά τα, αυτό το κατάλογο. Θα την αποστείλουμε λοιπόν. Λες απλά να πούμε ότι υπάρχει, αυτή, ε, υπάρχει αυτός ο κατάλογος. Ε, και πάλι από την Επιτροπή. Uh, λοιπόν, καταρχάς να απαντήσω το ερώτημα αυτό που έχει να κάνει με τη διασύνδεση ανάμεσα την πολιτική συνοχής και την τεχνική βοήθεια. Να σε εξηγήσω λίγο το πλαίσιο παροχής της τεχνικής αυτής βοήθειας. Κάθε κράτος έχει τα επιχειρησιακά του προγράμματα καθώς επίσης και τι συμφωνίε εταιρική σχέσης, στα πλαίσια των οποίων χρησιμοποιούν τα διαρθρωτικά ταμεία για συγκεκριμένα προγράμματα. Η τεχνική βοήθεια είναι κάτι το ξεχωριστό και διαφορετικό. Πρόκειται για τεχνική υποστήριξη, τεχνική βοήθεια, που δίδεται σε ορισμένε περιπτώσει για την διαχείριση των προγραμμάτων αυτών στα κράτη-μέλη. Επομένω, η τεχνική βοήθεια έρχεται και συμπληρώνει αυτό το οποίο γίνεται στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων, ιδίω προγραμμάτων πολιτικής συνοχής. Με άλλα λόγια δηλαδή, παρασχέθηκε βοήθεια η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή, στην καλύτερη λειτουργία και απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Πρόκειται ουσιαστικά για μια επικουρική, αν θέλετε, βοήθεια που δόθηκε σε σχέση με την πολιτική συνοχής και τα προγράμματα που υπάγονται σε αυτή την πολιτική. Όσον αφορά τώρα το δεύτερο ερώτημά σας, Νομίζω ότι απαντήσατε εσείς το άλλο το ερώτημα, έτσι δεν είναι, για τα έργα. Χρειάζεστε όμως περαιτέρω λεπτομέρειες, εκτός μικροφώνου. Κοιτάξτε και πάλι εδώ έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, έχουμε τις ομάδες εκείνες που χρησιμοποίησαν οι ελληνικές αρχές και που προσέλαβαν οι ελληνικές αρχές τελικά, που βρίσκονταν υπό την άμεση ευθύνη και λογοδοτούσαν σε ελληνικές αρχές. Στα πλαίσια των διαφορετικών ταμείων προβλέπονται κονδύλια για την πρόσληψη εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία όμως και με διεθνείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα μπορούν λοιπόν οι ελληνικές αρχές να έχουν άμεση επαφή με εμπειρογνώμονες είτε σε τοπικό επίπεδο είτε με διεθνείς εμπειρογνώμονες. Τι κάνουμε εμεί για τα σχέδια στα οποία παρεμβαίνουμε ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν μεσολαβούμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν κράτο μέλο μα ζητά να διαχειριστούμε ένα έργο, εμεί κοιτάμε, αξιολογούμε το έργο αυτό, προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι οι διάφοροι πάροχοι οι οποίοι θα μπορούσαν να εμπλακούν στο έργο αυτό και στη συνέχεια σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές εν προκειμένου λέμε κοιτάξτε αυτοί είναι οι πάροχοι υπηρεσιών, αυτοί μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση του έργου και να πρόκειται όμως το κράτος μέλος να αποφασίσει τελικά ποιους θα προσλάβει και ποιους όχι. Εμείς παρέχουμε απλώς συμβουλές. Την τελική απόφαση τη σύσταση τη ομάδα των εμπειρογνωμόνων τη λαμβάνει το κράτο μέλο και προκειμένου οι ελληνικέ αρχέ. Εμεί δίνουμε απλώ συμβουλέ για τα κράτη-μέλη στα οποία δίνουμε και τεχνική βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την απάντηση που μας δώσατε για το ποιος παρέχει τις υπηρεσίες αυτές αλλά επειδή και τα δύο είδη βοήθειας και για τις διαφορετικές ε, μεταρρυθμίσεις και για την πολιτική συνοχής ε, έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τη δημόσια δίκη, ίσως υπάρχει κάποια επικάλυψη. Και επίσης αναρωτιέμαι αν χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Επικάλυψη. Όχι, δεν γνωρίζουμε να υπάρχει επικάλυψη, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι ο εξή. Όταν λαμβάνουμε μία, ένα αίτημα για τεχνική βοήθεια, και μιλάω για το πώς λειτουργούμε τώρα, που είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε και η ομάδα δράση για την Ελλάδα. Όταν λάβουμε αίτημα τεχνικής υποστήριξης από ένα κράτος μέλος, το πρώτο που κάνουμε είναι το αίτημα αυτό το μοιραζόμαστε με όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλες τις γενικές διευθύνσεις και τους ρωτάμε, έχετε κάτι εσείς που να τρέχει σε αυτό το θέμα και μας απαντούν ναι ή όχι. Αν πούν όχι, τότε προχωράμε. Αν πούν ναι, τότε βέβαια ψάχνουμε για άλλου είδους τεχνική βοήθεια και λέμε στο κρατός μέλος έχετε ήδη χρήματα που καλύπτουν αυτού του είδους την τεχνική βοήθεια. Υπάρχει κάτι επιπλέον που θα θέλατε να ετηθείτε σε αυτό το πλαίσιο. Και με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε τις επικαλύψεις. Επίσης τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη να μας αποκαλύψουν εάν έχουν. Γιατί αν ζητούν από τη μία αλλά ήδη λαμβάνουν, τότε θα πρέπει και τα ίδια να γνωρίζουν πως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Οπότε, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει καμία επικάλυψη ε, με, τις, ε, με την τεχνική βοήθεια. Τώρα για τη χρηματοδότηση, στα πλαίσια της χρηματοδότησης για την Task Force για την Ελλάδα, τα χρήματα τα οποία διατέθηκαν στην ε, Task Force προέρχονταν από δύο πηγές. Πρώτον, από, την, από τον προϋπολογισμό κεντρικής τεχνικής βοήθειας που διαχειρίζεται η Κομισιόν, δηλαδή τα κονδύλια που είχαν μείνει από τον προϋπολογισμό αυτό στα τέλη της χρονιάς και τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιήθηκαν για την Ελλάδα. Και το υπόλοιπο, η άλλη πηγή χρηματοδότησης ήταν το άρθρο 25 του CPR που προσφέρει ένα μηχανισμό στην Ελλάδα μέσω του οποίου επιστρέφει χρήματα στην, στην Κομισιόν για να ε, υπογράψει συμβάσεις με παρόχους τεχνικής βοήθειας ε, εκ μέρους της. 15 εκατομμύρια επέστρεψαν έτσι από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τα χρησιμοποιήσουμε εμείς για τους ίδιους και να υπογράψουμε συμβάσεις ε, και να αναθέσουμε έργα τεχνικής βοήθειας. Άρα λοιπόν τα έστειλαν οι Έλληνες πίσω από τα δικά τους διαστατικά ταμεία και χρησιμοποιήσαμε και ε, κοντήλια από τους προϋπολογισμούς ε, και, από τον προπολογισμό κεντρική τεχνική βοήθεια που έχουμε στη διάθεσή μα. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με τον εθνικό προπολογισμό τεχνική βοήθεια. Ναι, νομίζω πω δεν έχουμε άλλε απορίε. κύριε Μακάρτη, υπήρχαν και κάποια εκπρόσωποι ε, στο πλαίσιο τη αποστολή, από την πλευρά τη γενική Διεύθυνση Γενικής ε, Ρίτζιο και πραγματικά ε, είδαμε πω αυτοί οι εκπρόσωποι τη Επιτροπή ήταν συνάδελφοι οι οποίοι ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για αυτά τα ζητήματα και ήξεραν πολλά και πραγματικά είδαμε πόσο ενεργητικά εσείς πιέσατε για να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτά ακριβώς τα ζητήματα και του ownership μας ε, οδήγησαν και εμάς σε περαιτέρω σκέψεις. Ε, δηλαδή και η ύπαρξη μία σειρά από προβλήματα κάποια από τα οποία ακούσαμε στη σημερινή συζήτηση, μα οδήγησαν και εμά σε κάποιε περαιτέρω σκέψει ω προ το τι μπορεί να γίνει. Και γνωρίζουμε ότι πραγματικά είναι δύσκολη ε, η κατάσταση. κύριο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Θα ήθελα να δώσω μια γενική απάντηση, ε, δίνοντα έμφαση στις συστάσεις τις οποίες κάνουμε στην εκθεσή μα. όπως ε, μόλις τώρα είπε και Γενική Διευθύντρια από την πλευρά τη Επιτροπή. Οι εν λόγω συστάσει λοιπόν έχουν ληφθεί υπόψη από την πλευρά τη Επιτροπή και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσουν ε, τη βάση για τις ε, περαιτέρω εργασίες της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα. Ε, δεν γνωρίζουμε ακόμα κάτι περισσότερο σχέση με την υπηρεσία που δημιουργεί αυτή την περίοδο η Επιτροπή, το πρόγραμμα δηλαδή της διαστατικής υποστήριξης. Δεν αξιολογήσαμε λοιπόν αυτό το ε, πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του καθώς συζητείται αυτή την περίοδο και στο Κοινοβούλιο και βέβαια αν ε, η Επιτροπή εδώ ελέγχου του ζητήσει μια γνωμοδότηση από πλευρά του Λακτικού Συνεδρίου θα την συντάξουμε. Άρα λοιπόν η δική μας έκθεση αφορούσε τα όσα έκανε η Task Force ε, και δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα ακριβώ ε, που δημιουργήθηκε τώρα ή θέλει να δημιουργήσει τώρα η Επιτροπή σε συνέχεια τη Task Force και επιλύει κάποια από αυτά τα προβλήματα. Ε, τώρα, το ερώτημα που έθεσε καταρχήν ο κύριο ό,τι αφορά τι ε, τριμηνιαίε εκθέσει. Εμείς ε, τονίσαμε εμείς ε, τα ορίσματά μας, αναφέραμε το τι βρήκαμε η Επιτροπή μπορεί να δώσει από και μετά συνέχεια στα όσα διαπιστώσαμε, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ιδιότερα στη θέση υπαριθμών 6, όπου καλούμε την Επιτροπή να προβεί σε μια ε, πλήρη εξπόστα εκ των υστέρων, δηλαδή αξιολόγηση των εργασιών της Task Force. Κατά συνέπεια, υπήρξαν κάποια συμπεράσματα τα οποία βγάλαμε εμείς με τη δική μα έκθεση, αλλά υπάρχουν και άλλα συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσατε να αντιλέσετε ακριβώς μέσω μιας τέτοιας ε, εκ των υστέρων αξιολόγηση από την πλευρά της Επιτροπής. Επίσης, έγιναν κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ των δύο προγραμμάτων, δηλαδή το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και το ε, πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής. Ε, το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας, λοιπόν, είναι ένα εργαλείο το οποίο δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματο των ελληνικών αρχών προκειμένου αυτές να ανταποκριθούν καλύτερα στις ε, απαιτήσει ε, που έθετε ε, μέσω του Μνημονίου Κατανόηση στο πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής. Και αυτό ακριβώς επεξηγεί και τις δυσκολίε που αντιμετώπισε και τις οποίες αναφέρουμε και εμείς στην εκθεσή μας η Επιτροπή. Ότι δηλαδή δεν είχε προβλεφθεί αυτό το πρόγραμμα τεχνική βοήθεια όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα χρηματοδοτική συνδρομή. Και ήδη αναφέρθηκε και η διαδικασία εδώ σε ό,τι αφορά την ανάληψη ευθύνη του ownership, ε, δηλαδή και από την Επιτροπή. Επίση, εμεί ε, στην σύσταση υπαριθμών 6 τονίζουμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει feedback σχόλια δηλαδή από τα ε, κράτη-μέλη που λαμβάνουν την ελόγω τεχνική βοήθεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αναφέρεται δηλαδή ότι η τεχνική αυτή βοήθεια παρασχέθηκε μετά από τα αιτήματα των κρατών μελών, αλλά από την άλλη πλευρά εμεί λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράση, θα πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητε και στόχοι. Και έτσι θα πρέπει να υπάρχουν και ακριβώ τα σχόλια που θα κάνει το κράτο μέλο που οποίο θα λαμβάνει τεχνική βοήθεια για να γίνεται μια ενημέρωση και αναλλαγή των σχετικών ε, στόχων ε, και του προγράμματο. Οπότε ε, αυτή εδώ η σύσταση θεωρούμε πω είναι μία από τι πλέον σημαντικέ μα. Και λέμε ότι η τεχνική βοήθεια θα πρέπει να εστιάζει στη ενίσχυση της, των διοικητικών αν θέλετε, δυνατοτήτων που έχουν οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Αναφέρθηκα και Κάποια ακόμα ζητήματα. Ε, τα οποία νομίζω πως κάλυψε ειδικότερα δηλαδή την ανησυχία που εξέφρασε ο κύριος Ευπλάναγκαν δηλαδή ε, μας είπε ότι ενδεχομένως να υποχρεωνόταν το κράτος μέλος να συμμορφωθεί με τις ενλογές Όχι, είπαμε ότι απλά είναι σημαντική η τεχνική βοήθεια για το κράτος μέλος. Και σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ε, τίποτα δεν υπάρχει στη διαδικασία που να εμποδίζει τη συμμετοχή του ε, και εδώ ε, στο έγγραφο θα βρείτε και ένα κατάλογο των ενδιαφερομένων φορέων, οι οποίοι γνώμοδοτησαν στο πλαίσιο ακριβώ τη σύνταξη τη εν λόγω έκθεση και στο πλαίσιο ακριβώ τη έκθεση που προετοιμάζουμε για το πρόγραμμα χρηματοδοτική ε, συνδρομή, ε, έχουμε προβλέψει διαβούλευση με μία σειρά από ε, ενδιαφερόμενου φορεί, μεταξύ αυτών και μη κυβερνητικέ οργανώσει. Από εκεί και μετά εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες από την πλευρά τη κυρία. Η κυρία Γιάλα έκανε μια ερώτηση σχετικά με τα διάφορα σύστημα, συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή τεχνικής βοήθειας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τονίσαμε και εμείς ιδιαίτερα και θεωρούμε πως ήταν μεγάλη επιτυχία το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να βάλει, ε, να δρομολογήσει αυτές τις ομάδες τεχνικής βοήθειας είτε σε συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών, είτε με διεθνείς οργανισμούς όπως επίσης με αποστολές των ίδιων των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν η τεχνική βοήθεια η οποία συνεργαζόταν με τις ελληνικές αρχές σε μόνιμη βάση. Και αυτό, για να είναι αποτελεσματικό τελικά, θα πρέπει κάπως να συντονίζεται. Και εκεί εμείς υπογραμμίζουμε το γεγονός πως υπήρξαν τέτοιου είδους δυσκολίες. Αναφερόμαστε πιο συγκεκριμένα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εθνικές αρχές και οι εθνικές υπηρεσίες συνεργασίας για την ανάπτυξη πρόσφεραν τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα και έδρασαν ως υποεργολάβοι για κάτι που με έναν πιο καλό προγραμματισμό θα μπορούσε να έχει γίνει πιο απλά. Αυτή είναι μία από τις συστάσεις που έχουμε συμπεριλάβει και είναι στην σύσταση παρθμό 1 μία καλύτερη περιγραφή αρμοδιοτήτων κτλ. Αυτό το streamlining δηλαδή όλων των διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη πως θα πρέπει να καλύπτει όσους συμμετέχουν. Επίσης, τονίζουμε πως υπήρξαν δυσκολίες με, κάποιες, ε, ε, με κάποιους διεθνείς οργανισμούς, για παράδειγμα το Δουνουτού ή το ΝΟΣΑ... οι οποίοι σε κάποιο βαθμό πήραν και αυτοί μέρους. Για το κόστος, έχετε δίκιο, κυρία Γιάλα. Στην έκθεση τη δική μας, γράφουμε πως δεν μπορέσαμε ούτε καν κατά τη διάρκεια της δικής μας ε, αποστολής και του δικού μας ελέγχου να δούμε ακριβώς ποιο ήταν το κόστος της τεχνικής βοήθειας. Είχαμε χρηματοδότηση, έχουμε το σημείο 24 της δικής μας έκθεσης όπου το περιγράφει, χρηματοδότηση η οποία προέρχεται από κονδύλια που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποια κονδύλια προέρχονται από τα διαφορετικά ταμεία είναι πολύ σημαντικό και το τονίζουμε στη συστάση μας να υπάρχει ένα συγκεκριμένος προϋπολογισμός και ένα συντονισμός όλων των πηγών χρηματοδότησης. Σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία τώρα, ο κύριος Βόγκαν νομίζω ότι έθεσε ένα σχετικό ερώτημα. καταλήγουμε στο εξή συμπέρασμα. Τα διορθωτικά ταμεία είναι στο μέσο που τελικά λειτουργήσε η τεχνική βοήθεια. Βοηθήσαμε δηλαδή μέσω της τεχνικής βοήθειας την καλύτερη απορρόφηση των διαθροτικών αυτών ταμείων. Είχαμε πολύ θετικά παραδείγματα εκεί και είχαμε και μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της ομάδας δράσης για την Ελλάδα και των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των διατροτικών ταμείων. Εντοπίστηκαν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση, τη φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά στην ε, έκθεση αυτή δεν κάνουμε μια γενική αξιολόγηση των επιπτώσεων που είχε τεχνική βοήθεια στα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά λέμε ότι η τεχνική αυτή βοήθεια βοήθησε στον εξορθολογισμό των διαδικασιών και στην αύξηση του ποσοστού απορρόφησης των διαρθρωτικών κονδυλίων. Απαντά τώρα τα, στα ερωτήματα τα οποία θέσατε απευθεία στο ελεγκτικό συνέδριο. Εναπόκειται πάντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις, τις συστάσεις μας και να δημιουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο τη νέα αυτή υπηρεσία υποστήριξης διαφροντικών μεταρρυθμίσεων, καθώς επίσης και το σχετικό ταμείο. Εμείς στο μέλλον θα συνεχίζουμε να δίνουμε συνέχεια στην έκθεση αυτή και να παρακολουθούμε την εφαρμογή της και αν μας ζητηθεί θα υποβάλουμε γνωμοδότηση και για το νέο αυτό πρόγραμμα υποστήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εκπονεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ναι, κύριε Μογορούσα. Πραγματικά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να θα μπορούσατε να ετοιμάσετε κάτι. Κύριε Αγιάλα, Sí, Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι αυτό που έχετε στην γραφική παράσταση 4. Είπατε ότι δεν μπορέσατε να βρείτε 100% πόση ήταν η χρηματοδότηση. Εδώ όμω φαίνεται πω το μεγαλύτερο τμήμα και φαίνεται εδώ η διαφορά, η Δύο χώροι λοιπόν στην οποία ε, δόθηκε περισσότερη τεχνική βοήθεια είναι ο χώρος υγείας και ε, τα εργασιακά θέματα και η κοινωνική ασφάλιση. Είναι δύο πολύ βασικά θέματα για την ε, Πολύ, πολύ, σημαντικό λοιπόν για την Κομισιόν, όπως επίσης ήταν η συνεργασία με τις εφορίες για τα δημοσιονομικά θέματα, όπως επίσης και το κτηματολόγιο. Πείτε μου λοιπόν, γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια απέτηση για τη δημόσια υγεία σε τεχνική βοήθεια. Το επαληθεύσατε, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη διαφορά με τα κονδύλια εδώ και σε σχέση με τα όλα τα υπόλοιπα. Δημόσια υγεία, βλέπω το πρόγραμμα το οποίο έχει πιο πολλά σημεία, για παράδειγμα, σε άλλα έργα 218 έχει πάρα πολλά που είναι η δημόσια υγεία, αλλά έχουν και άλλα με πολύ περισσότερα υποέργα. Γιατί λοιπόν ήταν τόσο πολύ δαπανηρή η βοήθεια στην δημόσια υγεία. Ήταν τόσο χάλια τα νοσοκομεία. Τι συνέβη. Αυτό ρωτώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Αν κοιτάξετε τον πίνακα αυτό, 4 δηλαδή, θα δείτε πως ε, στον τρόπο που ε, παρακολουθήσαμε το πώς πήγε η χρηματοδότηση για τους διάφορους κλάδους τεχνικής βοήθειας βασιζόμενοι στα στοιχεία τα οποία καταφέραμε να ε, συγκρίνουμε με την Task Force και με την ίδια την Επιτροπή είδαμε πως από τα έργα τα οποία χρειάστηκαν περισσότερα χρήματα ήταν η υγεία. Η υγεία παρόλα αυτά δεν είναι ένας από τους χώρους ε, τους οποίους εμείς ελέγξαμε οικονομικά ε, για να καταλήξουμε στα δικά μας ε, συμπεράσματα. Σας είπα πως κάποιους κλάδους τους ελέγξαμε με προσοχή στις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τα όσα έχουν να κάνουν με τον κόσμο του επιχειρήν, την ανταγωνιστικότητα. Όμως είχαμε και άλλους χώρους όπως η ιδιωτικοποίηση, το κτηματολόγιο, η χρήση γης, που νομίζω ότι σήμερα ήταν και το αντικείμενο μιας πολύ ενδιαφέρουσας ε, συνάντησης. Είναι χώρες τους οποίους εμείς δεν ελέγξαμε ε, λογιστικά. Είχαμε κάποιες δυσκολίες με τους κλάδους αυτούς, το γνωρίζουμε. Και η μελέτη που κάναμε για την τεχνική βοήθεια σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Το έδειξε αυτό, αλλά δεν έχουμε κάποια τεκμήρια που να μας οδηγούν στο να κατανοήσουμε πώς η τεχνική βοήθεια χρησιμοποιήθηκε και στους υπόλοιπους κλάδους στους οποίους εσείς αναφερθήκατε. Επιμένω πως αυτό δεν έχει, ε, δεν μας δεσμεύει, γιατί στο ε, πλαίσιο της επόμενης μας έκθεσης όπου θα έχουμε ελέγξει όχι την τεχνική βοήθεια αλλά την οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα που να καλύπτουν και τους χώρους αυτούς ε, στους οποίους αναφερθήκατε. Εδώ μας καλέσατε γιατί έχουμε ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών οργάνωσαν την προσφορά τεχνικής βοήθειας και κατά πόσο ήταν αποτελεσματική. Σα ευχαριστώ θερμά. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιο άλλο συνάδελφο ε, το λόγο, οπότε έχουμε ολοκληρώσει αυτό το workshop. Ευχαριστώ όλου ε, του ομιλητέ, ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο του Συνεδρίου, ευχαριστώ την Επιτροπή, ευχαριστούμε και την Γραμματεία ε, και το Policy Department. Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η διοργάνωση τέτοιων workshops, αλλά πραγματικά νομίζω πω ήταν πολύ σημαντικό. Α, όχι. Ε, Σουλάνκα, να είχε ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Απλώς να πω πως ε, ε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε σήμερα. Εγώ είμαι βέβαια καινούργιο το νέο μέλος της ε, Επιτροπής και πολλά από όσα ακούνε πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά εκείνο που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε το ελεκτικό συνέδριο το οποίο βρίσκεται σήμερα εδώ και να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα παρότι δεν έχουμε σχεδόν κανέναν ευρωβουλευτή. Δηλαδή σε κάποια φάση εδώ στη συνεδρία έχουμε τρία μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παρευρίσκονται και 54 διερμηνείς. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Προφανώς είναι απαραίτητο να κάνουμε τέτοια workshops, αλλά γιατί να, πραγματικά να έχουμε τέτοιες συνεδριάσεις όπου έχουμε τόσους πολλούς εξαιρετικούς διερμηνείς ε, που κοστίζουν και τόσο ακριβά να εργάζονται εδώ. The members get paid quite a lot to be here. They should... Ε, και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν μια παχυλαία αποσμίωση για να βρίσκονται εδώ. Οπότε θα ήθελα απλά να γνωρίζω ε, πόσο κόστισε για παράδειγμα η σημερινή συνεδρίαση όλων, δηλαδή ε, και η μέρες αποσμίωση των βουλευτών, των διερμηνέων, των, του διοικητικού προσωπικού και ούτω καθεξής. Αλλά βλέπω ότι είστε όλοι πάρα πολύ σκεπτικοί. Ε, μισό λεπτό, λέει Πρόεδρος εγώ εδώ προγράμμα τη συνεδρίαση, οπότε επιτρέψτε μου λίγο να συνδυνώσω τα πράγματα. Μπορούμε να σας πούμε ακριβώς εμείς εδώ ποιο είναι το κόστος, ε, για παράδειγμα, του να έχουμε ε, διερμηνία όλο τον χρόνο σε συνεδρίαση μας. Τώρα, έχουμε αυτούς τους συναδέλφους που έχουμε στην αίθουσα ε, και εσείς είστε ένας από αυτούς. Ε, πραγματικά χαιρόμαστε για όσους βρίσκονται εδώ. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες αυτής της Επιτροπής εδώ και 12 χρόνια και πραγματικά λέω σε πολλούς συναδέλφους ότι είναι σημαντικό να συμμετέχουν σε αυτή την Επιτροπή και για την Ευρώπη αλλά και επειδή ε, θα πρέπει να μπορούμε να δείξουμε ότι μα ενδιαφέρουν τα όσα συμβαίνουν και πραγματικά ευχαριστώ όσους παρευρίσκονται σήμερα εδώ για να ακούσουν αυτή τη συζήτηση. Το πρόβλημά μα είναι ότι όταν ε, θα, μας, ε, όταν θα μπορούσαν να μας πούν οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν θα παρευρεθούν, ότι δεν θα παρευρεθούν και έτσι θα μπορούσαμε να μην ζητήσουμε τη διερμηνία στις σχετικές γλώσσες, αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Ε, πάντως, ε, ε, το κόστο το οποίο υπάρχει στα διερμηνέα και ούτω καθεξή, νομίζω πω αποζημιώνεται και με το παραπάνω με τι εργασίε τη Ενλόγω Επιτροπή και δεν μπορούν, να, δεν μπορούν να το πούν άλλες επιτροπές ε, κοινοβουλευτικέ. Ναι, υπάρχουν εδώ κάποιε αδυναμίε, αν θέλετε συστημικού χαρακτήρα. Εδώ και αν ε, τελικά μπορούσαμε να οργανώσουμε τα πράγματα με άλλο τρόπο θα, θα το κάναμε, αλλά είναι όπω είναι και πραγματικά χαίρομαι για κάθε ένα από του συναδέλφου οι οποίοι παρευρίσκονται σε τέτοιου είδου workshops. Ευχαριστώ λοιπόν ε, για μία ακόμα φορά και την Γραμματεία και το Policy Department. Νομίζω πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το εν λόγω ζήτημα και να το κάνουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης, δηλαδή το ε, σημείο υπαριθμών 13. Και θα δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφο Γιάννη Σκάι, ο οποίο είναι ο Γενικό Συγητή τη Επιτροπή Προπολογισμού για τον προπολογισμό του 2017. Γιάννη, χαιρόμαστε που είσαι και πάλι εδώ μαζί μα και στην πρωινή μα συνεδρίαση ζουν εδώ, ε, για να μας ενημερώσεις ε, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας ε, των δύο επιτροπών δηλαδή. Η, δική μας συγκίτρια για το ζήτημα είναι η Ματίνα Λαπαγιώβα. Οπότε ξεκίνα εσύ Γιάννης, πες μας ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι θέλεις, σε τι θέλεις να στεγάσουμε σε αυτόν τον προβλησμό και θα δώσουμε και στη Ματίνα στην συνέχεια το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Για να καθησυχάσω εδώ και το συνάδελφο Φλάνναγκαν, εγώ είμαι πρόεδρο τη Επιτροπή ε, Προπολογισμού και ε, είμαι και γενικό γενικός για τα ζητήματα προπολογισμού. και ε, μόλι τώρα έρχομαι από μια συνεδρίαση τη Επιτροπή Ήτρε όπου έκανα μια αντίστοιχη παρουσίαση και Βέβαια διατρέχω όλες τις κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, ακριβώ γιατί είμαι γενικός Ε, Αλλά νομίζω είχαμε και τη δυνατότητα κύριε Φλάνακα να συμμετέχουμε σε μια συνεδρία στην Επιτροπή Οπότε επειδή ακριβώς παρακολουθώ τα όσα σημαίνουν σε διάφορες ε, επιτροπές ε, και επειδή κάνω ένα, ε, ένα έντος hopping σε συνεδριάσεις σήμερα, διαπιστώνω ότι πράγματι υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα ερμηνεία, δεν αξιοποιούνται πάντοτε και ούτω καθεξής. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πολύγλωσσο κοινοβούλιο, δεν νομίζω ότι μπορούν να οργανωθούν καλύτερα τα πράγματα από ό,τι είναι τώρα. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημά μας εδώ και δύο-τρεις εβδομάδες θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει ε, αυτήν την ε, διαδικασία καθώς η αρχική προθεσμία ήταν 25η Μαΐου που είχε τεθεί από την Επιτροπή για την δημοσίευση του σχεδίου του προπολογισμού, αλλά ε, τελικά αναβλήθηκε αυτή η προθεσμία με τη δικαιολογία από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έπρεπε να λάβει υπόψη και τι πρόσθετε δαπάνε σε συνέχεια τη κρίση. Οπότε στα τέλη αυτού του μήνα θα υποβάλει αυτό το σχέδιο. Ε, και ε, είμαι σίγουρος, λέει ο μιλητής, ότι αποτελεί συγκυρία η σύμπτωση αυτός, αυτή η χρονική συγκυρία σε σχέση και με το δημοψήφισμα ε, στη Μεγάλη Βρετανία. Εν πάση περιπτώσει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία του προπολογισμού, έγκριση του προπολογισμού, ακολουθεί το να πάει πρώτα ε, το σχέδιο στο Συμβούλιο, να τροποποιείται από αυτό και από εκεί και μετά το Κοινοβούλιο να ε, ξεκινάει ε, τις εργασίες του με βάση το σχέδιο όπως έχει τροποποιηθεί από το Συμβούλιο. Είναι ε, δύσκολη βέβαια μια τέτοια διαδικασία, είναι στενά τα χρονικά ε, ε, περιθώρια, αλλά επειδή ακριβώς είχαμε και τις εκλογές μας το 2015, ακριβώς τότε ήταν δυνατόν να συντομέσουμε την όλη διαδικασία σε έξι εβδομάδες, οπότε είναι δυνατό. Οπότε, ε, καταφέραμε να έχουμε την οθέτηση στην Ολομέλεια των σχετικών κατευθυντήρων γραμμών σε ό,τι αφορά τον, τον από την πλευρά του Κοινοβουλίου και είναι σημαντικό ακριβώς να γνωρίζουμε ότι τελικά και είναι οι γενικές πολιτικές κατευθύνσεις ε, με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Με τον προπολογισμό που εκτελείται αυτή τη στιγμή, δηλαδή τον προπολογισμό για το έτος 2016 στις κατηγορίες 3 ζητήματα μεταξωτερική πολιτική και 4 ζητήματα μεταξωτερική πολιτική λόγω ακριβώ τη ε, προσφυγική κρίση, έχουμε βρεθεί στα ανώτατα όρια, τα έχουμε εξαντλήσει στα λογοθέματα του προπολογισμού. Όπως δηλαδή αυτά προβλέπονται από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλα περιθώρια. Από εκεί και μετά υπάρχουν και άλλες επιτυχίες στις οποίες θα αναφερθώ, αλλά πραγματικά δεν θεωρώ πως μέχρι τα τέλη τουλάχιστον το 2016 το σενάριό μας θα βελτιωθεί. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν μπορώ να, να φανταστώ ότι θα χρειαστούμε λιγότερα κονδύλια για το έτος 2017, το δημοσιονομικό έτος 2017, σε σύγκριση με το 2016. Και το λέω γιατί αυτό, γιατί το Συμβούλιο ε, πάντα ακολουθεί την τακτική του να διαγράφει στοιχεία, για παράδειγμα δαπάνες δηλαδή της Επιτροπής όπως ε, βλέπω, ώστε να εξασφαλίσει ακριβώς μια καλύτερη ε, προσέγγιση με βάση δηλαδή το, μεταξύ του σχεδίου του προπολογισμού και του εκτελούμενου προπολογισμού. Άρα λοιπόν η προσφυγική κρίση δεν βλέπουμε να αμπλύνεται. Η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλύτερη, δεν θα είναι καλύτερη δηλαδή το 2017, ούτε ε, το 2016 υπήρξε καλύτερη σε σύγκριση με το 2015. Και το πολιτικό κλίμα μας επιβάλλει ε, να ε, αποδεσμεύσουμε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ ως ε, χέρια για το ΕΣΥ. Οπότε, με βάση αυτό το υπόβαθρο, κατά τη δική μου τουλάχιστον άποψη, το σχέδιο προπολογισμού βασίζεται σε κάποιες προβλέψεις υπερβολικά ευνοϊκές. Δηλαδή βασίζεται σε ένα πλαίσιο ε, το οποίο ενδεχομένω θα ήταν έγκυρο κατά έτη 2012-2013. Ε, και τότε δηλαδή αποφασίστηκε ότι το βασικός μας και πρωταρχικός στόχος είναι να επιτύχουμε ε, μείωση των δαπανών. Ε, αλλά εδώ και ε, δύο χρόνια ουσιαστικά ε, αυτό που κάνουμε είναι ότι όταν υπάρχουν κάποιες έκτακτες ανάγκες λαμβάνουμε κάποια κονδύλια από ένα τμήμα του προπολογισμού, κάνουμε εκεί κάποιες περικοπές για να μπορέσουμε να καλύψουμε ακριβώς το κενό που προέκυψε. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί πρόθεσμα. Τώρα, ένα δεύτερο ζήτημα. Ένα στόχο στο οποίο θέλαμε να διεκδικήσουμε είναι να έχουμε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή, αν θέλετε, υπεραξία, προστιθέμενη αξία ε, ε, του προϋπολογισμού και χαίρομαι που η Ολομέλεια αποφάσισε ότι πράγματι κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποτελέσει η προτεραιότητά μας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να προσανατολίζεται περισσότερο στι ε, χρηματοοικονομικού χαρακτήρα συστάσει τη Επιτροπή. Δηλαδή, όπως το 2015 υπάρχει αυτή η πρόβλεψη των δημοσιονομικών τάσεων, υπάρχει και ε, η έκθεση σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού του προηγούμενου έτους και υπήρξε και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και εκεί λοιπόν στο πλαίσιο όλων αυτών των διαδικασιών είδαμε ότι ε, το βασικό στόχος πλέον για τον προπολογισμό είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια θα πρέπει να προσανατολιστούμε προς τα εκεί, δηλαδή στις συγκεκριμένες συστάσεις που κάνει η Επιτροπή σε σχέση με αυτούς, αυτές τις προκλήσεις. Θα ήθελα δηλαδή να γίνει μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις γιατί ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμενο ε, γίνονται μια σειρά από προτάσεις τις οποίες μπορούμε να διαφωνούμε και εγώ προσωπικά πολιτικά αλλά έχουν σημασία και θα πρέπει λοιπόν να συζητηθούν, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και μετά το Κοινοβούλιο να αποφασίσει ώστε να ε, ακριβώς αντληθεί περισσότερη άξια από την αξιοποίηση των κοντιλίων του προϋπολογισμού της Ένωσης. Και από εκεί και μετά ε, υπάρχουν κάποια λήματα τα οποία προέκυψαν ε, σε, συνέχεια της στρατηγικής 2020. Δηλαδή, ακριβώ η σημερινή οικονομική μα κατάσταση μα οδηγεί σε περισσότερη ανεργία. Αυτή η ανεργία οδήγησε στην ανάγκη για την θέσπιση του ε, προγράμματο για την καταπολέμηση ανεργία ε, των νέων. και ε, λίγο ε, τα, όσα βελτιώσαμε σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του προπολογισμού είναι οι πληρωμέ, ε, που εκεί βέβαια ήταν μάλλον τεχνικού χαρακτήρα οι βελτιώσει, cash flow και ούτω καθεξής. Και επειδή όσοι συμμετέχουν στι εργασίε τη Επιτροπή του Προπολογισμού, στο πλαίσιο της, του, του, δημοσιονομικού πλαισίου, έχουμε θέσει πιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων υψηλότερε κατά 50 ε, σε σύγκριση ε, με τις ε, πιστώσει πληρωμών, τι σημαίνει ουσιαστικά ότι κάποια στιγμή θα οδηγηθούμε σε, στο να μην μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τον προπολογισμό. Και κάτι τέτοιο δεν μπορεί βέβαια να ισχύσει ω χρηστή δημοσιονομική πρακτική. Αν δεν ισχύσουν δηλαδή αυτέ οι προβλέψει, τότε ουσιαστικά εκείνο που κάνουμε είναι να μεταθέτουμε αυτές τις ε, πληρωμές για το μέλλον, αυτές τις υποχρεώσεις. Ε, αυτή είναι λοιπόν η γενικότερη κατάσταση. Ε, ε, όπως είπαμε θα έπρεπε να είχε ήδη δοθεί η εντολή, να έχει δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσει ο τριμερής ε, διάλογος. Τελικά μάλλον η διαδικασία θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. Εγώ πάντως θα συντάξω μια επιστολή με τις συστάσεις μου, ώστε ακριβώς να ακολουθήσουμε τις συστάσεις της Επιτροπής όλα τα θεσμικά όργανα, ούτως ώστε να δούμε το φθινόπωρο τελικά στο πλαίσιο της συζήτησης θα ξεκινήσει με το Συμβούλιο πού ακριβώς βρίσκεται το Συμβούλιο, ποιες είναι οι θέσεις του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ματίνα, έχει λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την καλή πρακτική που όσοι είναι ε, υπεύθυνοι για θέματα προπολογισμού έρχονται εδώ για να συζητήσουν μαζί μας. Παραδοσιακά στην περίπτωση αυτή της συζήτησης εμείς θίγουμε τις βασικές ανησυχίες που έχουμε διαπιστώσει πως εκκρεμούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής. Και ξέρετε φέτος ποιες ήταν αυτές οι αναζητήσεις πολλές γραμμές προϋπολογισμού δεν μας αφορούν. Παρ' όλα αυτά θα επιμείνουμε ε, ότι δεν χρειάζονται περίπου προγράμματα όπως το Περικλής, το Ηρακλής ή επίσης στο σύστημα κατά στο, στο σύστημα πληροφοριών κατά της απάτης. Γιατί όλα αυτά θα βοηθήσουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα στηρίξουν τα κράτη-μέλη και τα ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης. Είναι ακόμα πιο περίεργη η κατάσταση φέτος γιατί δεν έχει εγκρίνει σχέδιο προϋπολογισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα λοιπόν, χωρίς σχέδιο κειμένου, τι να σχολιάσουμε. Υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία έδειξαν κατά την απαλλαγή οι συνάδελφοι, για παράδειγμα οι περικοπές στο Horizon 2020, το, η εγγύηση για τους νέους, θέματα μετανάστευσης στα ευρωπαϊκά σχολεία, η πολιτική για τους Ρωμά κτλ. Θα ήθελα να επανέλθω στην βασική, ε, στον πυρήνα της έκθεσης μου για την απαλλαγή που είναι η αποδοτικότητα. Και θα ήθελα στο συσχείο αυτό να κάνω δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Ίσως η πρώτη να είναι πιο πολύ προς τον εισηγητή και η δεύτερη παρατήρηση να απευθύνεται πιο πολύ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην έκθεση για τον ενσωματωμένο ολοκληρωμένο εσωτερικό έλεγχο της 13ης Ιουνίου το Κοινοβουλίο δέχτηκε την άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου πως δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε την απόδοση χωρίς να έχουμε ε, εγγράψει στον προϋπολογισμό κονδύλια βασιζόμενη σε δείκτες αποδοτικότητας. Είπαμε πως χρειάζεται ένα σύστημα ε, κατάρτισης προϋπολογισμού που να βασίζεται σε δείκτες και κάθε γραμμή να συνοδεύεται από ε, παραδοτέα και από δείκτες αποδοτικότητας. Αυτό το αίτημα το αντιμετώπισε θετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τις λειτουργικές ε, δαπάνες που από το 2015 έχουμε στο σχέδιο προϋπολογισμού νομίζω ότι εδώ σε κάποιο βαθμό καλύπτονται οι ανησυχίες μας για τους δείκτες, για τα αποτελέσματα και για τα παραδοτέα. Παρόλα αυτά αυτά πλησιώσουν τις βασικές ε, ε, προσπάθειες που γίνονται με κάποια στοιχεία αποδοτικότητας, αλλά δεν είναι ο προπολογισμό που θα βασίζεται σε στόχους που εμείς ζητάμε. Νομίζω ότι θα πρέπει σε επαφές που έχετε με τις, ειδικές, ε, με τις αρμόδιες επιτρεπές να εκφράσουν την άποψή τους για τους στόχευση αυτών των δικτών αποδοτικότητας, γιατί μιλάμε για πολιτικούς στόχους και θα έπρεπε να ορίζονται από τις πολιτικές αρχές και όχι μόνο από τις υπηρεσίες και μάλιστα πριν να εγκρίνουμε ε, την, ε, τις πολιτικές δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει η Επιτροπή Προϋπολογισμού να ελέγξει το κατά πόσο κάθε γραμμή προϋπολογισμού στα πλαίσια της δουλειά που έχει γίνει από τις προηγούμενες επιτροπές είναι σωστή. Και η δεύτερη παρατήρηση απευθύνεται περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο έλεγχος δημοσιονομικού ελέγχου, ε, ε, ελέγχου του προπολογισμού ζητά απλουστεύσεις. Στη διαδικασία απαλλαγής ζητήσαμε πάρα πολλές απλουστεύσεις. Δεν υπάρχει λόγος να εγκρίνουμε κι άλλον ένα και άλλη μια ομάδα ε, δικτών και για να διευκολύνουμε και να απλουστεύσουμε τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει η Γενική Διευθύνση Κομισιόν να παραμένουν στους πολιτικούς στόχους και στους δείκτες που έχουν ε, στα προγράμματα ε, για τις λειτουργικές δαπάνες όταν εγκρίνουν το ε, σχέδιο διαχείρισης και την έκθεση πεπραγμένων για τις δράσεις τους. Έχουμε την έκθεση αξιολόγησης που βρίσκεται ήδη στις συνθήκες, είναι το άρθρο 13 και πιστεύω πως ε, τα σημεία αυτά στα οποία στάθηκα θα πρέπει να ενταχθούν στο ψήφισμα που θα συνοδεύει τον προϋπολογισμό και ελπίζω πως θα, εφραθείτε, ε, θα σταθείτε θετικά ε, στην άποψή μου πως θα πρέπει και για τους πολιτικούς στόχους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτεί για κάθε γραμμή του προϋπολογισμού. Είμαι ανοιχτή και περιμένω με προσδοκία να ακούσω τις απόψεις όλων των συναδέλφων. Νομίζω πως δεν είναι η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Uh, Κύριε Βόγκαν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την Μαρτίνα για την παρουσίαση που έκανε, αλλά και το Γένς για τα όσα μας είπε και για το τι ήρθε σήμερα εδώ. όντω έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το σχέδιο προπολογισμού τέλη Ιουνίου του 2017. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο σύμπτωση το τι γίνεται μετά το δημοψήφισμα για το Brexit. Πάντως, στον Ηνωμένο Βασίλειο ενδιαφέρονται πλέον πάρα πολύ για τις προτάσεις προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν πολλοί που περιμένουν να δουν τελικά τι θα προβλέψετε, αν θα έχετε κάποιες αυξήσεις πληρωμές ή όχι. Όσον αφορά τον ρόλο που έχετε αναλάβει εσεί, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι πήγατε σε διάφορε επιτροπέ. Προφανώ οι επιτροπέ οι οποίε ασχολούνται με δαπάνε θα ασχοληθούν πάρα πολύ με τι προτάσει, αλλά και εμεί εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώ παρακολουθεί την εξέλιξη του προπολογισμού και πώ εκτελείται ο προπολογισμό αυτό και πώ δαπανούνται τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρώμαστε περισσότερο στα αποτελέσματα, Ένα προπολογισμό ο οποίο θα πρέπει να επικεντρώνεται στις επιδόσεις. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, το ανέφερε και η Μαρτίνα. Νομίζω πάντως ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιφέρουμε ανάλογε τροποποίησει στο μελλοντικό προπολογισμό σε σχέση με αυτέ που μπορούμε να κάνουμε μέχρι σήμερα ενδεχομένω να πρέπει να περιμένουμε και την ολοκλήρωση τη αναθεώρηση του πολυτελού δημοσιονομικού πλαισίου ή μέχρι την ολοκλήρωση του νέου πολυτελικού δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το 2020 δηλαδή, για να κάνουμε πλέον ουσιώδει τροποποιήσει στον προπολογισμό. Α επικεντρωθούμε και σε κάποιε αλλαγέ που ενδεχομένω να γίνουν στον προπολογισμό του 2017, ενδεχομένω να υπάρξει μια αύξηση των κονδυλίων όσον αφορά την αντιμετώπιση τη προσφυγική κρίση Πρέπει να δούμε από πού θα προέλθουν όμως τα χρήματα αυτά. Και επίση η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα θέλει να παρακολουθεί επίση τον τρόπο με τον οποίο θα δαπανώνται τα χρήματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μα απασχολήσει και αυτό περισσότερο στο μέλλον. Επίση γνωρίζουμε ότι πήραμε χρήματα από τον ορίζοντα του 2020 και από, την, από το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε τα χρήματα αυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια του ΕΦΣΥ, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπήρξε σημαντική μείωση χρηματοδότησης και των δύο αυτών προγραμμάτων. Επίσης, η Επιτροπή μας, όπως γνωρίζετε, επιθυμεί κάθε φορά να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των πόρων αυτών και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ποιες δεσμεύσεις είμαστε σε θέση τελικά να λάβουμε. Είναι ιδιαίτερα λανθασμένη πρακτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει υποχρεώσεις και έπειτα να μην μπορεί να πληρώνει. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι 2 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ μέχρι το τέλος του έτους θα είναι τα χρήματα εκείνα τα οποία δεν θα καταφέρει τελικά να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα και για τους μελλοντικού προπολογισμού πόσο μάλλον αν στου μελλοντικού προπολογισμού δεν καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε τα ποσά αυτά τα οποία πρέπει να πάνε συγκεκριμένου δικαιούχου. Η κυρία Γιάννα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο ο οποίος ήρθε να μας επισκεφθεί και να ευχαριστήσω και τη Μαρτίνα που είναι η συγγήτρια και για τα όσα είπε που είναι τόσο συνεκτικά και συμπίπτουν ε, τόσο πολύ με τα όσα είχα προετοιμάσει εγώ ως ε, νεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε. Θα ήθελα να σχολιάσω όπως έχει συμβεί το ελεγκτικό συνέδριο να δηλώσει πώς, γιατί το είπε όχι μόνο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά προς το Κοινοβούλιο, πώς ήταν λάθος τη στιγμή που όταν σχεδιάζουμε ένα έργο ήταν τότε το Μάρκο Πόλο στις μεταφορές, να έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο χωρίς ε, ε, έργο, χωρίς ε, επαρκή προπολογισμό. Αυτό το θεωρούν σφάλμα. Και το λέω αυτό γιατί ισχύει. Το να φανταστούμε λοιπόν εδώ ένα προπολογισμό ο οποίος ήδη έχει αυτό το μικρόβιο σφάλματος γιατί θα είναι ηλιματικό ο προπολογισμό μας είναι ήδη η λάθος βάση γιατί μετά το Συμβούλιο θα μας υποχρεώσει να έχουμε αυτό το ανώμαλο μόρφωμα. Και κάτι το οποίο λέμε συχνά είναι πως ε, χρειαζόμαστε ριζικά μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιες κυρώσεις για το Συμβούλιο που μας υποχρεώνουν να δράσουμε κατά τις συνθήκες. γιατί μας οδηγεί το Συμβούλιο σε μια κατάσταση όπου χρόνο σε χρόνο εμείς πέφτουμε κάθε φορά σε πιο μεγάλο ε, σφάλμα επειδή ακριβώ μα περικόπτουν τον προπολογισμό. Να μια ιδέα. Να δημιουργήσουμε έναν τρόπο να φτάνουμε σε μια πραγματική απειλή και να πούμε, εάν δεν μας επιτρέπουν να συμμορφωθούμε με τη συνθήκη και μας οδηγούν σε ένα προπολογισμό που ήδη ε, συμπεριλαμβάνει το σφάλμα τη στιγμή της έγκρισή του, τότε θα πρέπει να υπάρχει κάποια δυνατότητα και όχι απλώς να κάνουμε κάποιες πολιτικές δηλώσεις. Δεύτερον, ανησυχώ πολύ με απασχολεί πολύ ποιος είναι η ποια είναι η στόχευση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Ωραία. Ξέρω πως το Ελληνικό συνέδριο ετοιμάζει ε, μία έκθεση για πολύ ανησυχητικά στοιχεία που έρχονται με τα ε, χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία εμεί θεωρούμε φυγή προ τα εμπρό. Ωραία, δεν υπάρχει χρήμα, ας μοχλεύσουμε. Αυτό συμβαίνει, γιατί χρηματοδοτούμε και να χρηματοδοτούμε την ΕΤΕ χωρί να πετυχαίνουμε αποτελέσματα. Και έχουμε σημαντικέ ε, ευρωπαϊκές πολιτικές που οδηγούνται σε χώρους που δεν μπορούμε εμείς να ελέγξουμε, γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που το αναλαμβάνει. Και αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το δούμε, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Γι' αυτό το έθεσα. Γενικό Διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού, κ. Γκάφα, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, ε, κυρία Πρόεδρε, για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε να σχολιάσω εγώ τα πολύ ενδιαφέροντα που ανέφερε ο Γενικός Συγητής για τον προπολογισμό του 2017 αλλά και για την ολοκλήρωση του προπολογισμού του 2015 και όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε ότι ε, η Επιτροπή ακόμα δεν έχει υποβάλει το σχέδιο προπολογισμού και όχι αποτελεί σύμπτωση ε, το ότι λαμβάνει η χώρα και το, δημοψήφισμα της, το βρετανικό δημοψήφισμα, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη μας ε, και τα ζητήματα μεταναστευση και ασφάλειας. Αυτό το σχέδιο προπολογισμού. Και βέβαια, εμεί συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας βάση τη συνθήκη, ότι δηλαδή έως την 1η Ιουλίου θα πρέπει να έχουμε υποβάλει ακριβώς ε, τις αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τις ε, δαπάνε, τον προπολογισμό δηλαδή. Ε, σε αυτό το σχέδιο προπολογισμού θα σεβαστούμε τις ε, προτεραιότητε που συμφωνήθηκαν τον, στον Ερνό Διάλογο στι 26 Μαρτίου με το Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο και αναφέρθηκαν ήδη κάποια στοιχεία σημαντικά αυτή τη συμφωνία, για παράδειγμα υποστήριξη των ευρωπαϊκών οικονομιών σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασία και τι επενδύσει και επίση η διασφάλιση ε, μια αποτελεσματική ανταπόκριση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσφυγική κρίση και τα αισθήματα ασφαλεία. Επίση, ε, εμεί θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό μια πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των κονδυλίων του προπολογισμού, όπως αξιώθηκε από την κυρία Τροβαγιώβα, την συγγήτρια, και θα λάβουμε υπόψη μας ε, τα όσα μας ζήτησε και το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την ολοκλήρωση του ε, τελευταίου προπολογισμού. θα λάβουμε υπόψη μας και τις συστάσεις μας για τον προσανατολισμό του προπολογισμού σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και θα λάβουμε υπόψη μας τα όσα υπόθηκαν σε ό,τι αφορά ε, τα, τους ε, δείκτες επιτυχίας, τα ορόσημα, τα χρονοδιαγράμματα και ούτω καθεξής. Γιατί με αυτόν τον τρόπο οι δύο ε, ε, επιτροπές, επιτροπές, ειδικότερα οι προπολογισμού και ελέγχου του προπολογισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τον διάλογό τους ε, και να υιοθετήσουν ε, ε, αυτά τα στοιχεία τους ώστε εμείς να είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες ε, πληροφορίες ε, στην, ε, την, στις εκθέσεις εκτέλεσης του προπολογισμού εάν εφαρμόσαμε σωστά, ακολουθήσαμε σωστά τους στόχους του προπολογισμού ή όχι. Και όπως αναφέρθηκε από την κυρία Καλμένη, θα έχουμε Ε, θα έχουμε αυτήν την πάρα πολύ διεξοδική έκθεση όπου θα αναφέρεται ακριβώς το τι επιτύχαμε ως προς τους στόχους, τα ορόσημα και το καθεξής. Επίσης θα ήθελα να ε, σας τονίσω ότι η Επιτροπή θα ε, σας παρουσιάσει έναν αποτελεσματικό προπολογισμό που θα κάνει θα είναι αποδοτικό και θα λαμβάνει υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση από τα μέλη τη Επιτροπή σα. Ευχαριστώ, λέει ο Να δώσω και πάλι το λόγο στον Γιάννη ε, Σκάια και στη συνέχεια στην εισηγητριά μα. Νομίζω πως η πρόταση που έκανε Μαθήνα είναι πάρα πολύ σημαντική, δηλαδή ε, οι ίδιες οι επιτροπές να κάνουν προτάσεις και να ασχοληθούν με το ζήτημα της μέτρησης της, των επιδόσεων, αν δηλαδή της επίτευξης αποτελεσμάτων με βάση τον προπολογισμό. Ε, δεν ξέρω βέβαια ε, σε ποιο βαθμό η Επιτροπή έχει προχωρήσει σε ό,τι αφορά ακριβώς το, αυτό το performance based budgeting, δηλαδή το σχεδιασμό του προπολογισμού με βάση ακριβώς ε, την ε, τις επιδόσεις ε, και νομίζω πως ε, θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες παραμέτρους τις οποίες εμείς ε, θα προωθήσουμε ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο οι οποίες θα πρέπει να αποτελέσουν την, τα στοιχεία με βάση τα οποία θα κρίνεται αυτή η αποδοτικότητα του προπολογισμού. Ο συνάδελφος έφυγε ο συνάδελφος ότι δηλαδή και είχε αναφέρει ότι δεν ε, λάβαμε ακόμα κάποια απάντηση από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ε, προτινόμενη αύξηση των κονδυλίων του προπολογισμού από την πλευρά μας. Εντάξει, εκείνο που εμείς λέμε είναι ότι οποιασδήποτε εντολές δίνουμε αν θέλετε ως θεσμικά όργανα θα πρέπει να πρικοδοτούνται από τα κατάλληλα κονδύλια του προπολογισμού. Αλλιώς δεν έχει νόημα, δεν έχει συνέπεια αυτό που κάνουμε εδώ. Δηλαδή, εάν συγκεκριμένε προτεραιότητε, τι οποίε θεσπίζουμε εμεί οι ίδιοι, δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα κονδύλια, τότε ε, ουσιαστικά βρισκόμαστε ενώπιον ενό διλήμματο. Ή θα υπάρχουν λιγότερα κονδύλια, ε, και θα, υπάρχουν, ε, θα υπάρχει και λιγότερη πολιτική, αν θέλετε, σε όλου αυτού του τομεί, είτε ακριβώ θα υπάρχουν και τα απαραίτητα κονδύλια για να υπάρχει και πολιτική. Και αν δεν θέλουμε κονδύλια, τότε μπορούμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί και μετά. Αλλά όταν το Συμβούλιο ε, προτείνει τέτοιε περικοπέ, τότε τελικά θα πρέπει να συζητήσουμε μαζί του και να δούμε τι τελικά θέλει να χρηματοδοτήσει το Συμβουλίο. Δηλαδή, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ε, δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερη πολιτική, περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα κονδύλια. Για κάποια χρόνια ε, ήταν δυνατό να κάνουμε κάτι τέτοιο για να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα, αλλά νομίζω πω ήδη ξεπεράσαμε τα όρια του τι μπορεί να γίνει σε αυτό το επίπεδο. Εδώ και 1,5 χρόνο αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά να ανοίγουμε τρύπε στον προπολογισμό από τη μία πλευρά ε, και να τις ε, κλείνουμε ουσιαστικά παίρνοντα ε, χρήματα από τον ίδιο τον προπολογισμό από άλλου τομεί για να κλείσουμε αυτέ τι τρύπε. Τώρα, αυτό που αναφέρθηκε ότι δηλαδή δεν υπάρχουν τα ε, απαραίτητα κονδύλια και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση αν διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια, τότε νομίζω εκείνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι ότι εάν βλέπουμε ότι για συγκεκριμένε πολιτικέ προτεραιότητες δεν προβλέπει ο προπολογισμό στα κατάλληλα κονδύλια, δεν θα πρέπει να δώσουμε την έγκρισή μας. Δηλαδή, ε, ε, εγώ δεν θεωρώ γιατί θα πρέπει εγώ να δώσω την έγκρισή μου για ένα σχέδιο προπολογισμού, ένα προπολογισμό ο οποίο θεωρώ πω δεν είναι βιώσιμο, ο οποίο δεν θα αντέξει μέχρι τα τέλη εν λόγω έτους. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ξεκινήσει ένας επικοδομητικός διάλογος για να δούμε τελικά τι θέλει το Συμβούλιο, τι δεν θέλει το Συμβούλιο και να αρχίσει τελικά τις προτεραιότητες του το Συμβούλιο. Και όταν και στα σημεία που θεωρεί ότι δεν έχει προτεραιότητα να γίνουν και αντίστοιχε περικοπές. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω όλους για την πρώτη αυτή αλλαγή απόψεων. Ήταν λίγο περίεργη αυτή η ανταλλαγή απόψεων για ένα σχέδιο προπολογισμού το οποίο δεν το έχουμε ακόμα ενώπιόν μας. Πάντως εγώ προσβλέπω σε δύο πράγματα καταρχάς. Θα ήθελα πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά να αρχίζει να εφαρμόζει όλες τις συστάσεις από τις εκθέσεις απαλλαγής και θα ήθελα επιτέλους να δω και το προσχέδιο προπολογισμού για το έτος 2017. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ε, ήσασταν πολύ σύντομοι. ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο τη μέσα μεταξύ μα και συνέβη και τη συνεδρίασή μα. Ε, οπότε διάφορα δεν έχει ζητήσει κάποιο συνάδελφο να αναφέρει κάτι. Ε, να σα πω ποιε θα είναι οι επόμενε συνεδριάσει μα. 27 Ιουνίου ε, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση ό,τι αφορά και τον ψήφο από την ε, Μάλτα, Οπότε θα πρέπει να είμαστε όσο δυνατό περισσότερο, ώστε ο Υπουργό να μπορεί να ληφθεί μια απόφαση με βάση την πλειοψηφία των μελών τη Επιτροπή. Μετά, ε, σημειώστε 4 Ιουλίου στο Σασούργο ότι έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την ε, Επιτροπή Ήτρε και ε, ο Επιτρόπος δεν ε, θα παρευρεθεί δυστυχώ, αλλά ο Γενικό Διευθυντή από την πλευρά τη Επιτροπή ε, θα περαστεί και θα έχουμε κάποιε παρουσιάσει από την πλευρά τη Ήτρε και στι 14 Ιουλίου ο Επίτροπο μα είπε ότι θα μπορέσει να παραστεί στη δική μα συνεδρίαση, ούτω ώστε όταν εκεί θα συζητήσουμε την δεύτερη έκθεση του το τότε θα είναι και ο Επίτροπος ε, εκεί, ε, ανέτη, ναι, στις 14 Ιουλίου, στην συνεδρίασή μας, εγώ συμφωνείτε και εσεί. Σας τα αναφέρω όλα αυτά για να γνωρίζετε εκ των προτέρων. Ε, πραγματικά. Λεπάμε που είμαστε τόσο λίγοι και όταν θα έχουμε αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον αριθμό συνεδριάσεων, θα έχουμε και περισσότερα μέλη που θα παρευρίσκονται στι επιτροπέ μα. Σα εύχομαι όλου καλό απόγευμα και σα λέω από τώρα ότι μάλλον θα βρέξει. Porque antes de que se el, compañero Flanagan, es que me he quedado con, la, con la, la Αυτό που θα ήθελα να μου δώσετε είναι αυτό που θέλω είναι να πω ότι δεν περισσεύουν οι διερμηνείς. Είμαστε λίγοι αλλά δεν θα ήθελα να ξεχάσετε πως γίνεται και web streaming. Υπάρχουν άτομα εκτός της αίθουσας. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, που δεν μιλούν τόσο καλά τα αγγλικά όπως εσείς κύριε Φλάνακαν και μας ακούνε. Και με το θέμα του Κάστορ, για παράδειγμα, μου στείλανε και μια πλατφόρμα με ένα σχόλιο που έλεγε «Μπείτε και ακούστε». Δηλαδή, είναι περισσότεροι εκτός αυτοί που μα ακούνε και έχουν δικαίωμα στη διερμηνία. Σας παρακαλώ, μην το ξεχνάτε. Δεν λέω πως θα πρέπει να πετάμε τα λεφτά μας, αλλά νομίζω πως σε αυτό ε, θα πρέπει να το επιτρέψουμε στους ε, συμπολίτες μας. Νομίζω πως αυτοί που μας ακούνε μέσω web streaming έχουν το δικαίωμα να βλέπουν και τους βουλευτές τους οποίους ψήφισαν και οι οποίοι πληρώνται καλά για να έρχονται στις συνεδριάσεις. Ρωτήσατε, μια, ερω... ρωτήσατε κάτι όταν έκανα αυτό το σχόλιο. Ξέρετε πόσο κόστησε αυτή η Επιτροπή. Καλύπτεται το κόστος αυτό από αυτό το οποίο λαμβάνουμε. Δηλαδή τι λαμβάνουμε. Είναι σημαντική η Επιτροπή μας, είναι ουσιαστική. Ξέρω πω οι ευρωβουλευτέ πρέπει να πάνε και σε άλλε επιτροπέ. Ανακοιτάξατε κοιτάξατε εσεί τα μέλη αυτή τη επιτροπή σήμερα. Να δείτε, είναι σε άλλε επιτροπέ. Γιατί αν το κάνετε, νομίζω θα δείτε ότι πολλοί απλώ δεν ήρθαν. Και αν πρόκειται εμεί να ελέγχουμε, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε του εαυτού μα. Ναι η ελευθερία ε, των ε, Ευρωβουλευτών και γενικά των βουλευτών ε, είναι ο απόλυτος και η πρωταρχική προτεραιότητα και αν επιλέγουν να μην παρευρίσκονται είναι δικαίωμά τους. Αυτά και καλό απόγευμα σε όλους.